Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ανάπτυξης που σήμερα αφιερώνεται πλήρως στο θέμα της επισητιστικής ασφάλειας. Θα ξεκινήσουμε με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Μήπως υπάρχουν αντιρρήσεις ή σχόλια για το σχέδιο ημερήσιας διάταξης? Όχι. Οπότε εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξή μας. Με ιδιαίτερη χαρά εγγενιάζω τη δημόσια ακρόασή μας, στην οποία έχουμε προσκαλέσει κορυφαίους εμπειρογνώμονες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συμμετέχοντες και κυρίως αυτούς που πραγματοποίησαν πραγματικά ένα μεγάλο ταξίδι για να έρθουν εδώ σήμερα. Θα ήθελα να σας επισημάνω μια αλλαγή στο πρόγραμμα. Δυστυχώς ο κύριος Ρούντολφ Μπούντζελ, που είναι εμπειρογνώμονα από το δεύτερο πάνελ, κολλείεται και δεν θα λάβει μέρο στην δημόσια ακρόαση. Έχει στείλει όμω γραπτό την εισήγησή του και ένα σχόλιο από την κοινωνία των πολιτών. Το θέμα της επιστηστικής ασφάλειας ή μάλλον της επιστηστικής ανασφάλειας είναι τόσο κορυφαίο και δυστυχώς και τόσο επίκαιρο που αποφασίσαμε κατά εξαίρεση στην Επιτροπή μας να διοργανώσουμε ολοήμερη δημόσια κρόαση. Ελπίζουμε έτσι να συζητήσουμε εκτενώς και βρυθώς τόσο πολυσύθετα αλλά και επίμαχα θέματα. Η ισχύουσα ανθρωπιστική κρίση που έχει πλήξει το κέρας Αφρικής και απειλεί περίπου 13 εκατομμύρια ανθρώπους, ε, χρήζει άμεσης και έκτακτης ε, απάντησης, αλλά και κάποιες βιώσιμης απόκρισης, προκειμένου να διαραγεί ο κύκλος ε, της πείνας και της επιστημιστικής ανασφάλειας στην περιοχή αυτή του κόσμου. Δεδομένη της έκτασης της κρίσης, η Επιτροπή μας αποφάσισε να μεταβεί και επιτόπου στα τέλη Οκτωβρίου, προκειμένου να αναλύσει την κατάσταση και να αξιολογήσει τον αντίκτυπο της ευρωπαϊκής αρρωγής. Η σημερινή συζήτηση δεν αφορά την τωρινή κρίση, αλλά θα επικεντρωθεί στα διαφορετικά αίτια αυτής τη επισητιστικής ανασφάλεια και τις πιθανές πολιτικές λύσεις που μπορούμε να δώσουμε μέσο και μάκρο πρόθεσμα Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω ότι η δημόσια αυτή ακρόαση διοργανώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να ενθαρρύνει και την ανταλλαγή απόψεων στα όρια του χρόνου φυσικά που έχουμε. Οπότε θα δώσω το λόγο όχι μόνο στα μέλη της Επιτροπής αλλά και στους υπόλοιπους συμμετέχοντες για να θέσουν ε, ερωτήσεις ή να κάνουν σχόλια προς τους επιρρογνώμονες. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω θερμά να σεβαστείτε το χρόνο αγόρευση, γιατί όλοι έχουν τον πειρασμό ε, μπαίνουν στον πειρασμό να μακρηγορήσουν. Όλοι έχουμε πολλά να πούμε, αλλά θέλουμε να εξασφαλίσουμε σε όλους το δικαίωμα να μιλήσουν. Από σεβασμό, μη τι άλλο, προ του υπόλοιπου συμμετέχοντε. Παρακαλώ να σεβαστείτε ευλαβικά το χρόνο αγόρευση. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Νταβίτ Ναβάρο, που είναι ο ειδικό απεσταλμένο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την επιστημική ασφάλεια και την διατροφή και ταυτόχρονα είναι συντονιστή τη ειδική ομάδα υψηλού επίπεδου για την παγκόσμια κρίση επισητιστικής ασφάλειας. Στην παρουσίασή του, ο κύριος Ναμπάρο θα μας εξηγήσει την πρόοδο και τις προκλήσεις ό,τι αφορά την ε, γενική ε, αντιμετώπιση της ε, κρίσης. Έχουμε και τον κύριο Μαμαντού Σοκό, πρόεδρο του Δικτύου Γεωργικών Οργανώσεων και Παραγωγών της Δυτικής Αφρικής, ΡΟΠΑ, θα μας δώσει την προοπτική του Νότου σε ό,τι αφορά την ε, επιστημιστική ασφάλεια και τι απαραίτητε πολιτικέ. Πριν δώσω το λόγο στου δύο βασικού ομιλητέ όμω ε, του πρώτου πάνελ, η πρόεδρο τη επιτροπή μα, η κυρία Ζολή, θα μα κάνει ενημερωτικά κάποια εισαγωγικά σχόλια. Για πέντε λεπτά λοιπόν δίνω το λόγο στην κυρία Ζολή. Σα ευχαριστώ. Καλώ ήρθατε όλοι καταρχήν. Είναι μια πολύ σημαντική αυτή η μέρα και αυτή η δημόσια κρόση για την Επιτροπή Ανάπτυξης, γιατί θεωρούμε το θέμα της επιστημιστικής ασφάλειας είναι από τα πιο σημαντικά ζητήματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Όταν αποφασίσαμε να διοργανώσουμε αυτή την ολοήμερη δημόσια ακρόαση, αγνοούσαμε το τραγικό τέλος που θα είχε η κατάσταση στο κέρας της Αφρικής. Διαπιστώνουμε ότι οι διαστάσεις της ε, επιστημιστικής κρίσης αυτή τη στιγμή είναι τεράστιες. Ε, εκτινάχθηκαν στα ύψη οι τιμές των τροφίμων, το ίδιο και οι τιμές του πετρελαίου. Έχουμε ένα λυσαλαίο ανταγωνισμό για την πρόσβαση στα, στο έδαφος, στη γη και στο νερό και τεράστια δεινά για τις ε, χώρες και τους πληθυσμούς τους. Μια κατάσταση που δυστυχώς ε, παρατείνει αυτή την επιστηστική κρίση. Και μάλιστα 100 εκατομμύρια άνθρωποι εξωθήθηκαν στη φτώχεια από την κρίση του 2008 και η επιστηστική κρίση από τον Ιούνιο του 2010 οδήγησε ακόμη 44 εκατομμύρια ανθρώπους στη φτώχεια. Δηλαδή δύο φορές το γαλλικό πληθυσμό. Έχουμε ανθρώπους που εδώ και τρία χρόνια λιμοκτονούν. Το 2011 λοιπόν ένα στους επτά ανθρώπους υποσυτίζεται και οι προβλέψεις δυστυχώς μόνο αισιόδοξε δεν είναι. Όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Και η δική μας ευθύνη είναι βαριά. Δεν θα ήθελα να προεξοφλήσω τα συμπεράσματα της ε, δημόσιας αυτής ακρόασης, αλλά θα ήθελα να επισημάνω ορισμένα θέματα που ευελπιστώ ότι θα γίνουν αντικείμενο επικοδομητικής και καρποφόρας συζήτησης. Θα πρέπει να εξετάσουμε τη συνάφεια της, των ευρωπαϊκών πολιτικών με την αναπτυξιακή πολιτική. Γιατί προστεί η αύξηση των γεωργικών επιδοτήσεων και των, α, της αναπτυξιακής βοήθειας αν η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα υπόλοιπα μέλη της G20 εξακολουθούν να επιδοτούν τη γεωργία τους και τις α, γεωργικές τους εξαγωγές. Αν δεν επιτρέψουμε στις αναπτυσσόμενες χώρες να καθορίσουν τη δική τους επισητιστική στρατηγική, ε, και να παραγάγουν κυρίως για τον πληθυσμό τους, ε, δεν θα δώσουμε λύση. Γιατί λοιπόν ε, δημιουργούμε νέα, νέους μηχανισμούς καταπολέμησης της πείνας, ενώ οι αναπτυγμένες χώρες επενδύουν στα βιοκαύσιμα που περιορίζουν τις καλλιεργήσιμες γέες για τα τρόφιμα και επιτείνουν την επιστημιστική ανασφάλεια. Πώς θα ε, παράγουμε τα 70% επιπλέον ε, τροφίμων που θα χρειαστεί ε, ένας πληθυσμός που θα αυξηθεί στα 3, κατά 3 δις μέχρι το 2050 όταν το ισχύον επιστηστικό σύστημα έχει αποτύχει χωρίς να αμφισβητήσουμε τον, τον καταστροφικό τρόπο παραγωγής και τον σπάταλο τρόπο κατανάλωσης. Στην αναπτυξιακή πολιτική διαπιστώνουμε ότι μειώνεται η υποστήριξη στη Γεωργία, ενώ έχουμε μια ταυτόχρονα ε, πολύ αρπακτική εμπορική πολιτική που καταπνίγει την τόπια παραγωγή. Αυτό όμως που είναι απαράδεκτο είναι ότι δεν καταφέραμε να εξαλείψουμε την κερδοσκοπία σε ό,τι αφορά τις γεωργικές πρωτεσίλες. Οι κερδοσκόποι που ψάχνουν επενδύσεις ε, στράφηκαν προς την αγορά των ε, τροφίμων και δημιουργήσαν τέτοια ρευστότητα και μεταβλητότητα των τιμών που έπληξαν τις ανα, ε, αναδυόμενες οικονομίες και ε, σε συνδυασμό με τις κλιματικές αλλαγές και την αύξηση των ε, γεωργικών τιμών ε, για την παραγωγή βιοκαυσίμων επιδίνωσε την κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρόλα αυτά φαίνεται ότι προτιμά να ικανοποιήσει το χρηματοπιστωτικό λόμπι αντί να ρυθμίσει τις χρηματοπιστωτικές αγορές στην Ευρώπη όπως έκαναν οι ΗΠΑ και να πλήξει τις ανισορροπίες και τις διαρθρωτικές ανισότητες που πλήττουν το παγκόσμιο επιστημιστικό σύστημα. Και στην Ευρώπη, η Γεωργία και αλλού θα έπρεπε να μας επιτρέπει να θρέφουμε τον πληθυσμό μας. Παρ' όλα αυτά οδήγησε στον πλουτισμό των μεγαλοκαλλιεργητών εις βάρος των μικρών καλλιεργητών και στο βορρά και στο νότο, οδήγησε στη διάφρωση των ε, δαφών, στη σπάνη των πηγών, στην ε, μείωση της βιοπικιλότητας, στην αύξηση των καυσαερίων και των αερίων του θερμοκηπίου. Θα πρέπει ε, να χρησιμοποιήσουμε τη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής ως ευκαιρία για να την κάνουμε συνεπή με τους αναπτυξιακούς μας στόχους. Το γεωργικό μας μοντέλο είναι δυσβάσταχτο και υποκριτικό. Δεν μπορούμε να λέμε ότι θέλουμε ε, να καταπολεμήσουμε τις κλιματικές αλλαγές και να πατάξουμε την επιστηστική ανασφάλεια όταν εξαρτώμαστε από μαζικές εισαγωγές σόγιας που η παραγωγή της στηρίζεται στην απερίμωση των δασών θα πρέπει να τροποποιήσουμε τον τρόπο παραγωγής μας, να περάσουμε από την υποτιθέμενη πράσινη επανάσταση που δεν τήρησε τους υποσχέσει τη, στην αγροοικολογία που θα διασφαλίσει την παραγωγικότητα, προστατεύοντα όμως και το φυσικό πλούτο και τους φυσικούς πόρου, όπως πρόβλεπε η παγκόσμια πρόβλεψη ε, στο, για, τις, ε, για την κατάσταση αυτή στην ε, στην έκθεση του 2008. Η Αιθιοπία εγκαταλείπει τη γεωργία της ε, σε ανταλλαγή με παγκόσμιες επενδύσεις. Και μάλιστα περιοχές που βρίσκονται σε κατάσταση κρίσης ανθρωπιστικής ε, βοήθειας δίνουν τις πιο έφορες γεές τους ε, ενώ η παραγωγικότητα, η κατάσταση του πληθυσμού τους είναι τραγική. Και παρόλα αυτά εκχωρούν αυτές τις γέες. Στη Λιβύη είχαμε συμβάσεις μεταξύ Λιβύης και Μαλή και είδαμε ότι ο Καντάφη είχε αγοράσει εκατοντάδες χιλιάδες εκτάρια με μηδενικό τίμημα. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες λοιπόν φυτεύουν φοινικόδεντρα, κατασκευάζουν ε, φράγματα και μάλιστα ε, εμποδίζουν ε, τη χρήση της άρδευσης για τους τοπικούς πληθυσμούς. Δεν συμβάλλουμε έτσι στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Οι πληθυσμοί αυτοί που ζούσαν από τη γεωρική τους πολιτική εργάζονται τώρα για 70 λεπτά του ευρώ τη μέρα σε τέτοιου είδους καλλιέργειες που είναι φθηνότερες και από τα φυτοφάρμακα. Δεν μπορούμε λοιπόν ε, να συνεχίσουμε έτσι την αναπτυξιακή μα πολιτική. Οι στόχοι τη οδηγία για τι ανανεώσιμε ενέργειε θα πρέπει να αναθεωρηθούν. Ένα μορατόριο στην αγορά γεωργικών εδαφών θα πρέπει να ισχύσει αμέσω στι περιοχέ που λιμοκτονούν και να εξεταστεί και για άλλε περιοχέ. Έχουμε όλο και μεγαλύτερη σπάνη πόρων και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ε, εφαρμογή μιας πραγματικής ε, επισητιστικής δικαιοσύνης χάρη του κοινού μα μέλλοντος και του μέλλοντο του πλανήτη μα, Και αυτή η μέρα θα είναι το πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Ζολή. Και τώρα ο λόγο των κύριο Ναβαρό για 10 λεπτά. Καταρχάς σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πρόσκληση που μου απευθύνατε να εκπροσωπήσω θα εκπροσωπήσω τον μπάνκι μου Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ σε αυτή την πάρα πολύ σημαντική δημόσια κρόση ε, η οποία γίνεται μετά από το πολύ σημαντικό ψήφισμα που ε, επικυρώθηκε, που ψηφίστηκε. Από ό,τι είπε και η πρόεδρος μας μόλις τώρα, ε, κατανοεί βασίτατα τα προβλήματα, όπως και πολλοί συμμετέχονται σήμερα στο ακροατήριο και ιδιαίτερο συνάδελφός μου Μαντού Σισόκο, ο συνάδελφοι οι οποίοι έχουν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες και έχουν δώσει μάχες για αυτό το θέμα. Πράγματι έγιναν πάρα πολύ σημαντικά, ε, σημαντικές δηλώσεις ε, από την πρόεδρο του πάνελ σήμερα εδώ και είναι γεγονός ότι τα τεράστια αυτά προβλήματα πολλών χωρών οφείλονται σε πολιτικές αποφάσεις που προέρχονται, που πηγάζουν είτε από την Ευρώπη, είτε από τη Βόρεια Αμερική, είτε από άλλες χώρες του ΟΣΑ. Δεν μπορούμε να υποθέσουμε ότι η επισητιστική ασφάλεια και το πρόβλημα του επισητισμού ε, ε, είναι καθαρά ευθύνη μόνο των τοπικών, των εθνικών κυβερνήσεων. Πρέπει να αναλάβουμε το θέμα αυτό με μεγάλη σοβαρότητα και να το αντιμετωπίσουμε. Στα επόμενα 8 λεπτά θα ήθελα να σας δώσω μία εικόνα των προσπασιών, μα, των μου να να διευθετήσουμε αυτό το πρόβλημα, να το χαλιναγωγήσουμε και να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις. Δεν είναι εύκολα θέματα αυτά, λύσεις δεν είναι εύκολες και γι' αυτό το έργο μου είναι να σας παρουσιάσω ε, τον τρόπο, την ανάλυση του ΟΗΕ ε, και τον τρόπο με τον οποίο ε, σκεφτόμαστε να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό από το 2008 και εντεύθε. Καταρχάς λοιπόν κάναμε μία ενδελεχή ανάλυση της κατάστασης και δημοσίευσαμε αυτό το πρόγραμμα δράσης της ομάδας υψηλού επίπεδου που ασχολείται με αυτό το θέμα. Αντί να επικεντρωθούμε μόνο ε, στην ε, παραγωγή τροφίμων και στα τρόφιμα, ε, βασίσαμε τη μελέτη αυτή στις πηγές από τις οποίες μπορούν οι άνθρωποι να προμηθευτούν τα τρόφιμα που χρειάζονται και ιδίως την τα τρόφιμα τα οποία έχουν διατροφική αξία για την επιβίωσή τους. Επικεντρωθήκαμε λοιπόν ε, κυρίως στη μελέτη των μικροκαλλιεργητών, των αγροτών που παράγουν ε, τα πολύτιμα αυτά τρόφιμα και ε, το περιβάλλον της γεωργίας μέσα στο οποίο παράγουν για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε μια σταθερότητα παραγωγής και υπάρχει νερού ε, η επισητιστική ασφάλεια δεν αναφέρεται πλέον αποκλειστικά και μόνο στον όγκο, στην ποσότητα των παραγωμένων τροφίμων, αλλά καλύπτει και περιλαμβάνει τους παραγωγούς, τις πηγές ε, ε, διατροφικής ενέργειας, τις πηγές των τροφίμων, τις πρώτες ύλες, τους ανθρώπους που παράγουν και τους ανθρώπους που καταναλώνουν. Ένα ολόκληρο πλέγμα λοιπόν. <clears throat> Αυτή τη στιγμή δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή, πρέπει να δώσουμε περισσότερη προσοχή στα, φρούστα προϊόντα ε, και ε, όχι όσο δίνουμε ε, προσοχή στο σημερινό κόσμο στην κτηνοτροφία, στην, στην αλληλεία, σε όλα τα τρόφιμα τα οποία έχουν επισητιστική αξία. Ε, όλα αυτά πρέπει να το δούμε μέσα σε, ένα, ε, σε μια ολοκληρωμένη δέσμη και να βοηθήσουμε ιδιαίτερα τους μικροπαραγωγούς και τους μικροκαλλιεργητές να τους δώσουμε δυνατότητα επιλογών, να τους ε, παράσχουμε τα εργαλεία και τις διαδικασίες μικρής κλίμακας που τους δίνουν τη δυνατότητα να παράγουν σωστά, να, να ε, αναπτύξουν τις ε, μικρές τους εκτάσεις, την μικροπαραγωγή τους και να δράσουν επιτυχώς σε μία μικροκλίμακα. Τώρα ποιος μπορεί να τα παράσει όλα αυτά, ποιος μπορεί να βοηθήσει. Ασφαλώς από τη μία πλευρά οι εθνικές κυβερνήσεις, αλλά δεν είναι μόνο οι εθνικές κυβερνήσεις. Ε, υπάρχουν βεβαίως και τα λόμπι τα οποία είναι πάρα πολύ χειρά και πιέζουν αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν και άλλοι φορείς οι οποίοι μπορούν εξίσου να συμβάλλουν. Ε, συνεταιριστικοί οργανισμοί, ενώσεις αγροτών παραγωγών, ε, περιφερειακές πρωτοβουλίες όπως ε, περιφερειακή πρωτοβουλία της, της Βόρειας Αφρικής για την αγροτική παραγωγή, τοπικές δηλαδή αγροτικές πρωτοβουλίες. Ε, η δημιουργία εταιρικών σχέσεων, συνεργασίας, ε, μεταξύ ε, παραγωγών και ομάδων ε, καταναλωτών παραγωγοί μπορούν να συνεργαστούν, να συνεταιριστούν, να οργανωθούν μαζί για να βελτιώσουν την, ε, την, παραγωγή τους και την, το, το, την μέθοδο εργασίας. Όλα αυτά πρέπει όμως να γίνουν χωρίς την αύξηση της γραφειοκρατίας, χωρίς ε, επαχθείς ε, διαδικασίες και ε, τίτλους, ηχηρούς τίτλους του ΟΗΕ ή άλλων μεγάλων οργανισμών, αλλά επαναλαμβάνω όλα αυτά μπορούν να γίνουν με μια συνεργασία σε μικρή τοπική ή περιφερειακή κλίμακα μεταξύ των ενδιαφερομένων μελών. Σας φαίνεται αυτό παράλογο, σας φαίνεται ουτοπικό, ιδεαλιστικό, ίσως. Όμως η πραγματικότητα μιας υπόλογης ε, δημοκρατικής κυβέρνησης δείχνει ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος να προχωρήσουμε και να βρούμε κάποιες λύσεις στην Αφρική και στην ε, Λατινική Αμερική. Βλέπουμε νέες προσεγγίσεις όσον αφορούν τα τρόφιμα, την παραγωγή, την κατανάλωση και την επισητιστική ασφάλεια και επάρκεια πολύ διαφορετικά από, ότι, από την προσέγγιση που είχαμε στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική τα τελευταία 40 χρόνια. Υπάρχει τώρα μια ε, κατεύθυνση η οποία προσπαθεί να παρακάμψει την επαχθή και βαριά γραφειοκρατία των, μεγάλων οργανισμών και να επικεντρωθεί στη μικρή κλίμακα. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό για μας ε, τους δημόσιους ε, ε, τους διεθνείς φορείς αλλά και τους πολιτικούς να αναλάβουμε τη συλλογική ευθύνη που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε με τα σωστά πολιτικά μέσα τα τεράστια προβλήματα τα οποία παραμένουν. Και είναι τα εξής. Πρώτον, το εμπόριο, οι διεθνείς εμπορικές συναλλαγές. Πολλά πράγματα ακόμα είναι, δεν είναι σωστά, είναι στραβά στο διεθνές εμπόριο, δεν λειτουργούν σωστά. Πρέπει να δώσουμε περισσότερη προσοχή στο τοπικό εμπόριο, στις τοπικές και περιφερειακές εμπορικές συναλλαγές μεταξύ διαφόρων μερών του κόσμου χωρίς να... Αυτός πρέπει να είναι και ο ρόλος δηλαδή και να ενισχύει αυτό το εμπόριο ο Παγκόσμιο Οργανισμός Εμπορίου. Μπορεί η επιστημιστική κατάσταση του κόσμου να βελτιωθεί όταν υπάρχει επάρκεια τροφίμων στις τοπικές αγορές. Παντού. Όμως αυτό το θέμα δεν μελετάται ε, σωστά ε, στις, ε, στους φορεί. φορείς. Η, πρόσβαση, η, η σωστή και εύκολη πρόσβαση στις αγορές τροφίμων πρέπει να ε, ε, επενδύσουμε προσεκτικά και επιλεκτικά ιδιαίτερα σε συνεταιρισμούς οι οποίοι είναι πολύ σημαντικοί ε, για, το τοπικό, για την τοπική γεωργία. Τι γίνεται τώρα με το ρόλο των γυναικών στη γεωργία. Ένα μεγάλο ποσοστό της γεωργικής παραγωγής γίνεται από γυναίκες οι οποίες ασχολούνται με την παραγωγή και θα πρέπει να βοηθήσουμε με, μία, ώστε να είναι η συμμετοχή των γυναικών πιο επικοδομητική και αηφόρο στην ανάπτυξη της γεωργίας. Πρέπει να επενδύσουμε στη γη, στις καλλιεργούμενες εκτάσεις και είδαμε σε πολλά μέρη της Αφρικής ότι οι τοπική παράγοντες, οι τοπικοί φορείς ε, θέλουν ήδη να κατευθύνουν τις επενδύσεις, θέλουν ήδη να ελέγχουν τις επενδύσεις και να αποφασίζουν εκείνοι ποια προγράμματα είναι καλύτερα να εφαρμοστούν. Τώρα, για τα βιοκαύσιμα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κανένας λόγος να έχουμε υποχρεωτικές ποσοστώσεις ή υποχρεωτικούς κανόνες παραγωγής ενός συγκεκριμένου όγκου βιοκαυσίμων έτσι ώστε γη που μπορεί να προσφερθεί για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων και τροφίμων να χρησιμοποιείται για βιοκαύσιμα και να χάνονται έτσι πολύτιμες καλλιεργούμενες εκτάσεις. Πρέπει να ε, βεβαίως να υπάρχει παραγωγή και να είναι ορθολογική η χρήση των βιοκαυσίμων αλλά πάντοτε να προσέχουμε ε, με ποιο τρόπο θα γίνει αυτή η της πολιτικής βιοκαυσίμων. Πρέπει να αποφύγουμε ε, κινδύνους και ρίσκα τα οποία είναι, δεν, είναι, δεν χρειάζονται ε, και πρέπει να δημιουργήσουμε ένα παγκόσμιο δίκτυο επιστημιστικής ασφάλειας. Τέλος, όταν λαμβάνονται πολιτικές αποφάσεις σε σώματα όπως αυτό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να κατανοούμε όλοι ότι υπάρχουν επιπτώσεις σε όλα τα μέρη του κόσμου. Έχετε ένα πάρα πολύ δυνατό ψήφισμα πλέον στα χέρια σας. Τώρα πρέπει να ανασκουμποθούμε και να δουλέψουμε σκληρά. Πρέπει να μετρατρέψουμε τα λόγια σε έργα και πρέπει να ε, ε, δημιουργήσουμε, να εξασφαλίσουμε μια επιστημιστική ασφάλεια και ένα ε, εισόδημα στους τοπικούς παραγωγούς και στους καλλιεργητές ώστε να μπορέσουν να αποφύγουν τις σοβαρότερες επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος και της έλλειψης τροφίμων. Αυτό το μεγάλο έργο μπορούμε να επιτύχουμε με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να διορθώσουμε ορισμένα από τα πολιτικά, από τα ασφάλματα της πολιτικής που, που έγιναν τις τελευταίες δεκαετίες και στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική. Και τώρα ο λόγος στον κύριο Σισόκο για δέκα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ευχαριστώ το Ευρωκοινοβούλιο και ιδίω την Επιτροπή σας που με προσκαλέσατε να συμμετάσχω σε αυτή την ακρόαση. Εκτίμησα ιδιαίτερα την παρουσίαση του κυρίου Ναβάρο. Είναι ένας πραγματικός σύμμαχός μας. Ένα σύστημα που θα προσπαθήσω και εγώ να το παρουσιάσω. Ίσως πρέπει να ξεκινήσω λέγοντας ότι η Αφρική νοτίως της Σαχάρας καθώς και ο νότος της Ινδίας εκπροσωπούν το 30% του παγκόσμιου πληθυσμού που βρίσκεται σε συνθήκες οικονομικής επισφάλειας. Η κατάσταση αυτή δεν είναι ούτε φυσική ούτε ανεπίλητη. Χρειάζονται Χρειάστηκαν μάλλον συγκεκριμένε στρατηγικέ ώστε να γίνουν διορθωτικά μόνιμα προβλήματα των περιοχών αυτών, οι καταστάσει αυτέ. Η Αφρική ξοδεύει 25 δισεκατομμύρια δολάρια για να εισάγει τρόφιμα και η Αφρικανή γεωργία είναι η μόνη ομάδα του ανθρώπινου πληθυσμού που όταν εργάζεται καλά χάνει χρήματα. Και χάνει χρήματα ιδίω όταν υπάρχει καλή σοδιά. Θα μου πείτε δεν είναι δυνατό αυτό. Φυσικά και είναι. Το ποσοστό των αγροτικών πιστώσεων είναι 15-30%. Ακόμη και όταν υπάρχει κινητοποίηση των εσωτερικών πόρων ε, στο όνομα της ασφάλειας οι εισρωές χρήματος ή άλλων ουσιών όπως τα φυτοφάρμακα, τα ζυζανιοκτώνα είναι ανεξέλεγκτες. Οι πολιτικοί βασίζονται σε γνωματεύσεις εμπειρογνωμόνων και σε συγκεκριμένα επιστημονικά μοντέλα αγνώντας πλήρως τα, τους πολίτες, τα άτομα, γυναίκες και άντρες που εργάζονται για να δημιουργηθούν αυτές τις πολιτικές και να υπάρχουν αυτοί οι πολιτικοί. Και όπως μόλις είπε ο κύριος Ναβάρο, συχνά λέγεται ότι πρέπει να αυξηθεί η παραγωγή για ένα 70 ή 40% για το μέλλον. Χάνουμε όμως 30% της παγκόσμιας παραγωγής. Για υπολογίστε, 30% της παγκόσμιας παραγωγής στη Δύση, τις απώλειες, τις έχουμε τη στιγμή της βαθμονόμησης. Θα ξέρετε όλοι ότι για να παραχθεί πατάτα υπάρχουν ας πούμε οι μεσές, οι μεγάλες και οι μικρές. Αλλά για να φτάσουν στο σούπερ μάρκετ πρέπει να έχουν τις σωστές διαστάσεις. Δεν πάει στο ράφι του σούπερ μάρκετ ό,τι παράγεται. Ενώ στην Αφρική έχουμε τα χωράφια και τα ποτάμια μεταξύ των σπιτιών και των χωριών. Η κατάσταση είναι πολύ καλά γνωστή. Και για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή θα πρέπει να είμαστε διορατικοί. Θα πρέπει η Αφρική να χρησιμοποιεί πλέον λοιπάσματα και να ανοιχτεί και στην αγορά. Αλλά σε ποια αγορά. Υπάρχουν δύο βασικά προϊόντα στην Αφρική. Τα προϊόντα προς τις εξαγωγές που δεν μας ανήκουν, οπότε πλήττεται η αγορά μας. Σκεφτείτε για παράδειγμα τον ανανά και προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται για τη διατροφή και τα οποία βρίσκονται στην αγορά μας. Δεν ανησυχούμε όμως για το πώς θα θεσπιστούν υποδομές, πώ θα ιδρυθούν υποδομές για την εσωτερική αγορά, αλλά διαρκώς πιεζόμαστε για να βρισκόμαστε σε συγχρονισμό με τις διεθνείς αγορές, ενώ δεν είμαστε καταναλωτές των ίδιων προϊόντων και δεν είμαστε και αγοραστές τους. Όταν λοιπόν κανείς θέλει να χτίσει τον πλούτο του σε προϊόντα που άλλοι τους δίνουν την αξία τους, ε, δεν είναι αυτή η σωστή κατεύθυνση για να είναι κανείς ανεξάρτητος. Επίσης πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι στην Αφρική περισσότερο από πουδήποτε και ιδίως από την Ευρώπη το 40% της παραγωγής χρησιμοποιείται για την διατροφή κατοίκων. Είτε μιλάμε για τα δημητριακά, είτε για τα λαχανικά, για τα προεκπαιχτικά. Αυτό είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Αφρικής. 40%, το 40% αυτό είναι εκτός τοπικής αγοράς. Και με τις διευθυντικές μεταρρυθμίσεις που εμποδίζουν τις κυβερνήσεις να χρηματοδοτήσουν τη γεωργία, ακόμη και όταν τα πλεονάσματα της παραγωγής έφτασαν στα ωριά τους στην Ευρώπη, δεν θα υπάρξουν συνθήκες να αλλάξουν τα πράγματα. Τα αποθηκευμένα τρόφιμα της Ευρώπης δεν μπορούν τουλάχιστον να φτάσουν ως εμάς. Έτσι, μέσα σε μια 25 ετία άλλαξαν τη τροφική συνήθεια των Αφρικανών. Και αυτό λειτουργήσε ως τροχοπέδι. για τη χρήση του κεχριού, για την παραγωγή του σόργου και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν έχει αλλάξει τελείως η εικόνα της αγοράς της, ε, των τροφίμων. Φανταστείτε τώρα, στα σχολεία, από το δημοτικό ως το πανεπιστήμιο, να μην γίνεται λόγος για τις διατροφικές αξίες των ε, πολιτισμών μας. Και πολλοί συχνά στις καντίνες των σχολείων τα προϊόντα που δίδονται και πολλούνται είναι εισαγόμενα για να φάνε τα παιδιά. Έχουμε αναθρέψει λοιπόν γενιές ολόκληρες ε, ώστε να γυρνάνε την πλάτη στις πραγματικές παραδοσιακές αξίες της τροφής. Κι όμως υπάρχει ένας καθοριστικός σύνδεσμος εδώ μεταξύ της βιοπικιλότητας που ουσιαστικά επιτρέπει την σπορά και την διασπορά της γεωργίας, κάτι που μόνο με το γεωργικό σύστημα μπορεί να αναπτυχθεί. Και με το γεωργικό σύστημα ε, καθορίζονται οι διατροφικές συνήθειες που είναι ε, βαθιά ριζωμένες στην οτροπία μας. Έτσι λοιπόν η καταστροφή αυτής της φυσικής διαδικασίας είναι καθοριστική όταν μιλάμε για τα τρόφιμα και τι διατροφικέ μα συνήθειε, όταν έχουμε να κάνουμε με τρόφιμα που εισάγονται από αλλού. Σε αυτή την κατάσταση, λοιπόν, όπω το είπατε, κύριε Ναβάρο, χώρες που πλήττονται στο κέρας της Αφρικής είναι χώρες όπου τα κτίρια χτίζονται σαν μανιτάρια και εμφανίζονται σαν μανιτάρια όπου ο δυτικός κόσμος εδώ και 25 χρόνια αντλεί τρόφιμα αλλά οι μικροί γεωργοί δεν έχουν κανένα δικαίωμα ούτε ως προς τις αρχές της χώρας τους ούτε καμία στήριξη από τον προπολογισμό της χώρας πολύ περισσότερο ασχολείται κανείς με τους πολιτικούς παρά με την πλειοψηφία του πληθυσμού. Έτσι λοιπόν με μια τέτοια κατάσταση νομίζω ότι την πρώτη στη ευθύνη την, ε, πρέπει να την αναλάβει η ίδια η Αφρική. Δεν είναι λογικό, δεν έχει νόημα η βοήθεια για τη διατροφή της Αφρικής να προέρχεται από το Ευρωκοινοβούλιο ή την ε, Ηνωμένε ή την διεθνή ανάπτυξη, αναπτυξική βοήθεια. Διότι στους ίδιους τους πολιτισμούς μας στα ήθη και στα έθιμά μας, σε όλη την Αφρική Νοτίου της Σαχάρας, όταν ο πατέρας μιας οικογένειας φτάνει στο συμπεράσμα ότι δεν έχει τα χρήματα για να ε, θρέψει την οικογένειά του, τότε πρέπει να εξαφανιστεί το πρόσωπο της γης. Είναι όνειδος αυτό, να μην μπορεί να καλύψει τις διτροφικές ανάγκες της οικογένειάς του. Και ας σκεφτούμε αυτό στο επίπεδο κυβέρνηση τι σημαίνει. Εμείς θα έπρεπε να είμαστε στο, στην πρώτη γραμμή. Να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, γιατί ε, και τους πόρους έχουμε και τις δυνατότητες. Έχουμε χωρικούς και γεωργούς που μπορούν να θρέψουν την Αφρική. Ο αδερφός μου, ο Μισεσάλ από την Δυτική Αφρική, θα σας παρουσιάσει το έργο του, την δουλειά γυναικών γεωργών από την Σομαλία, για να σας δείξει ότι Υπάρχουν γεωργοί στην Αφρική που μπορούν να θρέψουν την Ήπειρο. Όμω η γεωργία δεν σημαίνει μόνο παραγωγή και κατανάλωση. Θα πρέπει να τοποθετείται στα πλαίσια μια ευρύτερη πολιτική. Και εμεί μιλήσαμε για το ΚΑΝΤΕΠ στη χώρα μα. Ε, ένα πλαίσιο, αλλά βασίστηκε στο μοντέλο τη συγκέντρωση των εδαφών και των επενδύσεων. Με το σύστημα αυτό οι μικρότεροι γεωργοί βρίσκονται εκτό συστήματο ενώ το ΚΑΝΤΕΠ θα έπρεπε να ευνοεί την οικογενειακή γεωργία και ούτω καθεξής. Υπάρχουν λοιπόν πολιτικές δηλώσεις και υπάρχουν και δράσεις. Όμως γιατί, γιατί υπάρχει αυτή η αντίφαση. Διότι απλούστατα η Αφρική ακόμη δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει την απεικιοκρατία. Οι αναφορές μας είναι πάντοτε οι άλλοι εκτός Αφρικής. Ενώ θα έπρεπε να χτίσουμε το μέλλον μας στις δικές μας τις δυνατότητες μια εξέλιξη που να μας επιτρέπει να έχουμε πρόσβαση. Δεν είμαστε Ευρωπαίοι, δεν είμαστε Αμερικάνοι, δεν είμαστε Κινέζοι. Έχουμε τη δική μας ιστορία, το δικό μας πολιτισμό. Αυτό θα έπρεπε να καλλιεργήσουμε για να βγούμε από την ε, σημερινή κατάσταση. Και αυτό είναι η βασική αρχή που θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Όπως ξέρετε, η Αφρική είναι αόρατη και που θα έπρεπε να είναι εμφανέστατη. Μας αναφέρουν στις συζητήσεις του ΠΟΕ. Τι λένε όμως. Όλοι γνωρίζουν τι συμβαίνει στον ΠΟΕ. Μόνο η Αφρική δεν θα κερδίσει τίποτα από αυτές τις διαπραγματεύσεις για τη διεθνή αγορά. Διότι δεν διαθέτουμε τα εργαλεία, ούτε τα μέσα. Και να φτάσω τώρα στα συμπεράσματά μου. Εγώ θεωρώ ότι οι Αφρικανοί χωρικοί και γεωργοί έχουν την υποχρέωση να διοργανωθούν καλύτερα. Εμείς είμαστε πλειοψηφία και εμείς πρέπει να πούμε όχι σε αυτήν την ασυδοσία, την ανευθυνότητα των κυβερνήσεών μα που δεν δυσκολεύονται να ζητήσουν επισητιστική ασφάλεια, στήριξη και το κάνουν αυτό εδώ και 40 χρόνια. Δεύτερη πρόταση. Οι αφρικανικές κυβερνήσεις να υπολογίσουν πόσο επίγον είναι να βασιστούν σε αυτές τις αρχές. Η Αφρική και ο δυτικό κόσμο πολύ σύντομα θα βρεθούν εκείνοι σε κατάσταση επισητιστική ανασφάλεια. Βρίσκονται στα όρια τη παραγωγή του, τη διαδικασία που τι έκαναν μεγάλου παραγωγού δημητριακών. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Δεν είναι λοιπόν καθόλου ασφαλή η διεθνή αγορά. Ούτε πρέπει να υπολογίζει σε αυτή η Αφρική. Πρέπει στη δική τη γεωργία να υπολογίζει για να καλύψει τι ανάγκε του πληθυσμού τη. Η Αφρική νοτίω τη Σαχάρα. Θα είμαστε 780 εκατομμύρια σε 25 χρόνια. Και Τώρα, ενώ έχουμε το μισό πληθυσμό, πάλι δεν καλύπτουμε τι επιστημιστικέ μα ανάγκε. Θα πρέπει λοιπόν να χτίσουμε την επιστημιστική μα ασφάλεια όχι στη διεθνή αγορά, αλλά στι δικέ μα δυνατότητε. Γι' αυτό μιλάμε με την Ευρώπη, το λέμε αυτό στο δυτικό κόσμο, όπω πρέπει να το πούμε και στην ε, Αφρική, θα πρέπει την καλλιέργεια να την αναλάβουν οι ίδιοι οικογενειάρχε. Αυτό που δημιούργησε πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Γεωργία είναι αυτό που έπληξε τελικά και την Αφρικανική. Αμελήσαμε, υποτιμήσαμε τη σημασία της παραγωγή τροφίμων για την ίδια την εγχώρια κατανάλωση. Αυτό είναι το πρώτο καθήκον των γεωργών. Δεν είναι να βρίσκονται παντού στον κόσμο. Όχι. Στη δική του τη χώρα πρέπει να βρίσκονται. Εκεί που αποφάσισαν να ζήσουν ελεύθερα και να παράγουν τρόφιμα για αυτή την περιοχή του κόσμου όπου ζουν. Για τον ίδιο λόγο κανένα δίκαιο, κανένα νόμο στον κόσμο δεν μπορεί να εμποδίζει του ανθρώπου να επιλέγουν το επαγγελμά του, να το εξασκούν και να ζουν από αυτό. Κανεί γεωργό τον κόσμο δεν ζητά επιδότηση μόνο του. Όλοι θέλουν να εργαστούν απλώ και να ζουν από τη δουλειά του. Οι πολιτικοί του επιχρεώνουν για να υπερασπιστούν τα δικά του τα συμφέροντα. Εκείνοι θεσπίζουν συστήματα για να πούν ότι όχι, δεν μπορεί να έχει το τρόφιμο την τάδε τιμή. Ποιο όμω μπορεί να το δεχτεί αυτό, ποιο είναι εκείνο που αποφασίζει ότι πρέπει κανεί να ζήσει σε συνθήκε φτώχεια και να μην μπορεί να αγοράσουμε τα τρόφιμα σε κανονικέ τιμέ. Ποιο θα μα λέει ότι όχι πρέπει να πάτε στη διεθνή ας πούμε αγορά. Το θεωρώ σημαντικό λοιπόν αυτό. Το τρίτο στοιχείο <clears throat> είναι ότι η Ευρώπη και ο δυτικό κόσμο πρέπει να κατανοήσουν το εξή. Οι πολιτικέ γεωργίας, είτε σε νέα πλαίσια είτε όχι, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και τα όρια. Τα όρια των οικονομικών σα συστημάτων και ε, δυνατοτήτων. Το καταναλωτικό σύστημα είναι περιορισμένο. Δεν μπορεί να βασιστεί σε αυτό το μέλλον τη Ευρώπη και του κόσμου το καταναλώνουν χωρίς κανένα όριο και το παράγει χωρίς κανένα όριο δεν σημαίνει τίποτα. Θα εξαντλήσουμε όλοι μαζί τους φυσικούς πόρους του κόσμου. Δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό. Πρέπει λοιπόν να σας πω ότι τι οφορώ τιμή στην Ευρώπη. Ναι, είναι πιο προηγμένη από τις αφρικανικές κυβερνήσεις για τις συζητήσεις τουλάχιστον και τις διαπραγματεύσεις όπως φαίνεται από τη σημερινή μας συνεδρίαση. Ναι, από τι αφορούνται εμεί τους Ευρωπαίους γεωργούς που διαρκώς προσκαλούν Αφρικανούς γεωργούς για να τους λένε και να τους επαναλαμβάνουν ότι ναι, ανήκουμε στο ίδιο σύστημα και πρέπει να συνεργαστούμε, να εργαστούμε όλοι μαζί. Όμως πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει μέλλον. Δεν υπάρχει μέλλον για την Ευρώπη χωρίς την Αφρική και αντιστρόφως. Βρισκόμαστε λοιπόν στην ίδια βάρκα και πρέπει μαζί να κοπηλατήσουμε για να βγούμε στην ακτή. Για την ευημερία και στην Αφρική και στην Ευρώπη. Για να συνεχίσουμε μαζί να ζούμε σε συνθήκες παγκόσμιας ευημερίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Αρχίζουμε τη συζήτηση. Για ερωτήσεις, παρατηρήσεις, ο κύριος Μπέργκμαν ζήτησε πρώτα το λόγο. Έχετε το λόγο κύριε Μπέργκμαν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ γρήγοροι ήσασταν. Απλώ σήκωσα το χέρι. Ε, κύριε Σισόκο, έχω μία ερώτηση προς εσάς. Γνωρίζετε τη μοίρα των ιερέων, ε, των ε, βοσκών μάλλον στην Δυτική Αφρική, που είναι νομάδες και φυσικά δεν ε, κρατούν ε, τα κοπάδια τους ε, αρκετό καιρό στον ίδιο, στην ίδια περιοχή και είναι μόνοι τους, οι μόνοι ικανοί σε, αυτή, σε αυτές τις άγονες ή, ή μη άγονες περιοχές να καλλιεργήσουν. Οι μόνοι ικανοί και μάλιστα η συμμετοχή τους είναι πολύ σημαντική γιατί παράγουν, παράγουν και πολύ σημαντικό ποσοστό των πρωτεϊνών και πολυ σημαντικο ποσοστο των πρωτεινων έχουν δυνατότητες όχι μόνο επιβίωσης, αλλά και πραγματικής διαβίωσης ε, με τον τρόπο που επιλέγουν. Αλλά η Αιθιοπική κυβέρνηση, κυρίως η Αιθιοπική κυβέρνηση, αλλά και άλλες κυβερνήσεις, ε, περιφρονούν αυτό τον ομαδικό τρόπο ζωής, γιατί θεωρούν ότι η καθιστική ζωή, η ζωή στις πόλεις είναι ο πιο αξιοπρεπής τρόπος ζωής, είναι ο πιο ε, σύγχρονος τρόπος ζωής και περιφρονούν αυτή την ομαδική περιπλανόμενη ζωή των βοσκών αυτών. Ο κύριος Σεναρή πολύ πρόσφατα, ο Πρωθυπουργό, το εξήγησε σαφέστατα. Είπε ότι αυτός ο τρόπος ζωής, ο περιπλανόμενος, ο νομαδικός, είναι παλιαμοδίτικος και θα πρέπει να σταματήσει. Είναι αναχρονιστικός. Πώς πιστεύετε ότι οι κυβερνήσεις της Δυτικής Αφρικής ε, θα ενεργήσουν, θα δράσουν απέναντι σε αυτούς τους βοσκούς, αυτούς τους χωρικούς που θέλουν να επιβιώσουν, πώς μπορούν να αλλάξουν την νοοτροπία τους απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους ε, και να σεβαστούν τον τρόπο ζωής τους. Δεν θα πρέπει να γίνουν αυτοί οι άνθρωποι ένα αντικείμενο του ευρωπαϊκού συναισθηματισμού, γιατί πραγματικά αξίζουν κάτι καλύτερο, αξίζουν μια καλύτερη μοίρα. Γιατί αυτό είναι ο μόνος τρόπος παραγωγής εκεί και μάλιστα με βιώσιμο από οικονομική άποψη τρόπο σε αυτές τις ε, ε, άνυδρες περιοχές. Πώς πιστεύετε ότι μπορούμε να πείσουμε την αιθιοπική κυβέρνηση προκειμένου να σεβαστεί αυτόν τον τρόπο ζωής. Ευχαριστώ. Θα ήθελε κανείς άλλο το λόγο. Η κυρία Κρέτσου. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και έχω μία σύντομη πρακτική ερώτηση, πρακτικής φύσεως ερώτηση στον κύριο Ναβάρο. Για αυτή την ε, ομάδα ταχείας απέμβασης. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι τα προγράμματα αυτά και οι παροχές ε, ε, δίνονται στους σωστούς δικαιούχους. Έχουμε έναν μηχανισμό σωστό που μπορεί να παρακολουθήσει αυτήν την ροή της βοήθειας προς τους ε, δικαιούχους. Ξέρουμε ακριβώς ότι πηγαίνει εκεί που πρέπει. Θα ήθελα να μας εξηγήσει λίγο περισσότερο το μηχανισμό δράσης αυτής της ομάδας ταχείας ενέργειας, ταχείας παρέμβασης. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Ποιος άλλος θέλει το λόγο? Η κυρία Θεοχάρους. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Τρία ζητήματα έχω να θίξω. Το πρώτο είναι ότι συμφωνώ απόλυτα πως <clears throat> χωρίς να στηρίξουμε την πρωτογενή παραγωγή των μικρών καλλιεργητών δεν μπορούμε να βγούμε από αυτό το πρόβλημα. Το δεύτερο είναι ότι για να γίνει αυτό χρειάζεται η μεταφορά γνώσης, τεχνογνωσίας, ικανοτήτων και η παρακολούθηση και αυτά σας τα λέω από προσωπική εμπειρία και το τρίτο είναι ότι η ανθρωπιστική βοήθεια όταν φτάνει είναι πια σε πάρα πολύ κακή κατάσταση και αυτό το έχουμε βιώσει. Δηλαδή να ανοίγουμε τα κοντέινερς και να πετάγονται τεράστιοι αρουραίοι από μέσα. Ευχαριστώ. Merci Σας ευχαριστώ. Ποιος άλλος θέλει το λόγο παρακαλώ. Όποιος λαμβάνει το λόγο να είναι λακωνικός, να μας πει ποιος είναι καταρχήν και δύο λεπτά για τρία για τρει ομιλητέ. Ε, βέβαια το πρωί είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, το ξέρω. Ο κύριος Μποβέ. Ζωζέ Μποβέ, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξη Πέθρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχω μία ερώτηση προς τον ειδικό αποσταλμένο του Γενικού γραμματέα του ΟΗΕ. Άκουσα την ομιλία του, που φυσικά ήταν σωστή, με βρίσκει σύμφωνο, ήταν ενδιαφέρουσα. Πώς είναι δυνατόν όμως ο ΙΕ να έχει τόσο ωραίε ομιλίες και η κατάσταση να είναι τέτοια τραγική. Κάπου υπάρχει μία απόκληση, μία χασμοδία. Γιατί έχουμε καταπληκτικές ε, δηλώσει για τα δικαιώματα των μικροκαλλιεργητών, αλλά η κατάσταση δεν αλλάζει. Τι γίνεται, δύο άλλα λέμε και άλλα κάνουμε ή υπάρχει επικάλυψη ή αποκλίνουσες δραστηριότητε. Ο κύριος Σισόκο μίλησε για τον ΠΟΕ και τη θέση του απέναντι στην Αφρική. Σίγουρα και εκεί υπάρχει μια αντίφαση. Και η γεωργία στον ΠΟΕ ε, ε, οδήγησε σε όλεθρο τους μικροκαλλιεργητές σε πολλές περιοχές του κόσμου. Ο ΙΕ μπορεί να αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες και είναι και ένα θέμα διεθνούς δικαίου. Το δικαίωμα στη διατροφή είναι αναγνωρισμένο στα ε, δικαιώματα του πολίτη, στα πολιτιστικά και κοινωνικά δικαιώματα και κατοχυρώνεται. Αλλά δεν αρκούν αυτές οι διακήρυξεις. Θα πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι και πιο απαιτητικοί. Μήπως λοιπόν ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ θα μπορούσε να συμπεριλάβει και το δικαίωμα στην επιστηστική κυριαρχία, στα θεμελιώδη δικαιώματα, ώστε να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τους πληθυσμούς και τις χώρες απέναντι στον ντάμπινγκ, γιατί πολύ λόγος γίνεται γι' αυτό, αλλά πράξη μία και αλλαγή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπέργμαν. Αν μου επιτρέπετε μία ακόμα ερώτηση προς τον κύριο Ναβάρο. Θα μπορούσε κανείς να πει, αλλά παρακαλώ να μου το επιβεβαιώσετε, ότι αυτή τη στιγμή αλλάζουν τα πράγματα στη γεωργία στις αναπτυσσόμενες χώρες, δεδομένου ότι ο μισός πληθυσμός του κόσμου ζει σε αστικές περιοχές. Και αυτές οι αστικές ε, περιοχές κατοικούνται συνήθως από πρώην παραγωγούς, γεωργούς που άφησαν την Ήπεθρο και πήγαν στα, στα μεγάλα αστικά κέντρα. Όμως, Αυτές οι αστικές περιοχές ε, αυτή τη στιγμή έχουν κατοίκους ε, πληθυσμούς που δεν μπορούν να διατραφούν, δεν έχουν επάρκεια τροφίμων πολλές φορές. Υπάρχει λοιπόν μια νέα κατάσταση, μια νέα πρόκληση. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε με αυτή τη ε, νέα πραγματικότητα εάν έχει γίνει εκμετάλλευση αυτού του γεγονότους η, Γαλλική Υπηρεσία Ανάπτυξης έχει εκδώσει ένα θαυμάσιο εγχειρίδιο για το μέλλον των, της Αφρικανικής Υπήρου. Το μέλλον της Αφρικανικής Υπήρου. Ταυτόχρονα η επιστημιστική κρίση του 2008 δεν έχει περάσει ακόμα. Οπότε μας παρουσιάζεται μια δεύτερη ευκαιρία προς τους γεωργούς των αναπτυσσομένων χωρών. Διότι ξαφνικά οι κυβερνήσεις έχουν καταλάβει ότι το μέλλον τους δεν ε, ε, δεν θα είναι λαμπρό λόγω των κοινωνικών ε, αναταραχών και εντάσεων που παρουσιάζονται σε πολλές χώρες αλλά το μέλλον τους μπορεί να εξασφαλιστεί επιβίωση δηλαδή εάν έχουν ε, φροντίσει να εξασφαλίσουν τρόφιμα και τη διατροφική επάρκεια του πληθυσμού και έτσι να υπάρχει μια ηρεμία και μια σταθερή κατάσταση. Η επισητιστική κρίση λοιπόν μέσα στα πλαίσια μιας αυξανόμενης της αστικοποίησης των πληθυσμών δείχνει ότι υπάρχει μια διαφορετική ροή ε, στην γεωργική ανάπτυξη. Θα ήθελα να μας εξηγήσετε εάν αυτή η συζήτηση έχει, γίνεται, εάν αυτή η ανάλυση έχει εντοπίσει αυτές τις ενδεχόμενες λαμπρές ευκαιρίες, ενδεχομένως λαμπρές ευκαιρίες παρουσιάζονται τώρα στην Ήπεθρο. Και μία τελευταία ερώτηση από μια κυρία που δεν την γνωρίζω. Κάρενα Νιούς. Έχω μια ερώτηση προς τον κύριο Σισόκο. Μας μίλησε για τις αγωγές και τις δυσκολίες που έχουν οι γεωργοί στην Δυτική Αφρική στην προσπάθεια να ανταγωνιστούν τους γεωργούς των άλλων περιοχών του κόσμου. Είναι ενδιαφέρον το παράδειγμα που μας ανέφερε και θα ήθελα τη γνώση του κύριου Σισόκο ότι αφορά τα μέτρα που έλαβαν οι κυβερνήσεις της Δυτικής Αφρικής μετά την επισητιστική κρίση του 2008. Πώς προσπάθησαν οι κυβερνήσεις αυτές ε, να δώσουν ενάυσματα για την αύξηση της παραγωγής ρυζιού. Πώς αναλύει την κατάσταση. Θεωρεί ότι έχει λάβει χώρα κάποια βελτίωση. Ήταν επιτυχής η κυβερνήση στην προσπάθεια τόνωσης της ντόπια παραγωγής ή θεωρεί ότι απέτυχαν σε αυτό το έργο. Σας ευχαριστώ. Πρέπει να πω ότι είμαι πραγματικά λίαν εντυπωσιασμένος όταν ακούω ξανά και ξανά ότι οι Ευρωπαίοι δεν καταλαβαίνουν την Αφρική. Με εντυπωσιάζει αυτή η δήλωση. Ενώ εμείς κάνουμε κάθε προσπάθεια να καταλάβουμε την Αφρική από απόψεως παραδοσιακών ε, δομών οικογενειακής ζωής ε, και άλλων στοιχείων. Κύριε Ναβάρο, είπατε ότι υπάρχει ανάγκη ε, να βοηθήσουμε τους παραγωγούς να οργανωθούν, τους γεωργούς δηλαδή, να οργανώσουν καλύτερα τη δουλειά τους, την παραγωγή τους κλπ. Αυτό με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, διότι και εμείς αναγνωρίσαμε ότι οι συνεταιρισμοί στην ε, γεωργική παραγωγή έχουν μέλλον και φαίνεται ότι υπάρχουν διάφορα αίτια κυρίως από τις ε, παλαιότερες κομμουνιστικές, ε, κομμουνιστικά μοντέλα παραγωγής που, που, δεν έχουν προσφέρει τις κατάλληλες ευκαιρίες. Κύριε Ναβάρο, πιστεύετε ότι επενδύουμε αρκετά να βοηθήσουμε την Αφρική να, βρει το, το, να, να ξαναβρει τις παραδοσιακές της ρίζες. Σας ευχαριστώ. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στους προσκεκλημένους μας, στους εμπειρογνώμονές μας για να απαντήσουν, ξεκινώντας από τον κύριο Ναβάρο. Ευχαριστώ. Καλό θα ήταν να είχαμε μισή ώρα τουλάχιστον να συζητήσουμε όλα τα θέματα που προέκυψαν. Επειδή όμως αυτό δεν είναι δυνατόν, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, τηλεγραφικός. Και ζητώ και προτέρων συγγνώμη αν δεν μπορέσω να απαντήσω πλήρως. Καταρχάς απαντώ στον κύριο Μπέρμαν στην πρώτη του παρέμβαση. Τα τελευταία τρία χρόνια κατανοήσαμε ότι η αναπτυξιακή βοήθεια ήταν τυφλή όσον αφορά τις ανάγκες ε, των ε, αγροτοβοσκών και της αγροτικής βοσκής. Ε, αυτό φαίνεται καθαρά από την τεράστια κρίση που υπάρχει στο κέρας της Αφρικής. Τώρα κατανοούμε ότι το να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να επιβιώσουν μαζί με ε, τα κοπάδια τους ε, και να μπορέσουν να τα βοσκήσουν έτσι όπως πρέπει και εκεί όπου πρέπει είναι ένας πολύ καλύτερος τρόπος επιβίωσης η κτηνιατρική φροντίδα έχει τελείως παραμεληθεί ως στοιχείο της ε, αγροτικής, ε, του αγροτικού πλαισίου και της, αγροτικής, ε, της συζήτησης των αγροτικών θεμάτων. Κτηνιατρική βοήθεια, ένα πλαίσιο κτηνιατρικής παροχής υπηρεσιών, η ενίσχυση της βοσκής των βοσκοτόπων και των βοσκών, των είναι ε, αναγκαία. Δεν επαρκεί να, να ε, λένε κυβερνήσεις ότι η, ο παραδοσιακός τρόπος ε, βοσκής των κοπαδιών και επιβίωσης των κοπαδιών είναι τεράστιο πρόβλημα. Πρέπει να τους βοηθήσουμε να μπορούν να διατηρηθεί αυτή η παραδοσιακή βοσκή και αυτός ο παραδοσιακός τρόπος επιβίωσης των γεωργών και των κοινοτήτων, των κυρίως νομαδικών. Όσον αφορά τώρα για την δύναμη ε, κρούσης, αυτή η ομάδα υψηλών στελεχών, υψηλή ομάδα κρούσης, επικεντρώνεται ε, στην παροχή της επισητιστικής βοήθειας. Ο ρόλος της είναι να εξασφαλίσει όχι μόνο ότι η παροχή αυτή βοήθειας πηγαίνει στους κατάλληλους δικαιούχους, αλλά είναι η σημεοφόρος αν θέλετε οργάνωση για την παροχή της επιστημιστικής βοήθειας και γι' αυτό προσέχει ιδιαίτερα τα προγράμματά της που, και πώς διοχετεύονται. Ε, διαπιστώσαμε στη Σομαλία ότι η επιστημιστική βοήθεια δεν μπορούσε να πάει στους δικαιούχους, αυτούς τους ανθρώπους που έπρεπε, διότι υπήρχαν διάφορα παρακλάδια και διάφορες παράπλευρες αρτηρίες όπου χανόταν η βοήθεια και γι' αυτό ε, είπαμε ότι δεν θα ζητήσουμε πλέον χρήματα από τους φορολογούμενους και πολλοί από τους φορολογούμενους είναι ε, Ευρωπαίοι, ε, δικοί σας ε, ψηφοφόροι και πολίτες. Δεν θα ζητάμε λοιπόν χρήματα από τους φορολογούμενους για προγράμματα τα οποία είναι χαμένα εκ των προτέρων. Δηλαδή για μια ψητιστική βοήθεια που δεν πάει στους δικαιούχους, από την οποία δεν υποφελούνται οι πληθυσμοί που πρέπει. Σας διαβεβαιώ λοιπόν ότι προσέχουμε ιδιαίτερα αυτό το πρόβλημα. Αυτό το, το ζήτημα άπτεται και της επόμενης ερώτησης για την ποιότητα της επιστικής βοήθειας. Δεν είναι μόνο λοιπόν η παροχή στους δικαιούχους, αλλά είναι και η υψηλή ποιότητα της ψηφιστικής ε, βοήθειας για την οποία φροντίζουμε. Ε, κύριε Μποβέ, σα ευχαριστώ για την ερώτησή σας ε, και για τις παρατηρήσεις ε, σε αυτά που είπα εγώ. Θα ήθελα... Α, υποθέτω ότι ξέρετε την απάντηση στο ερώτημά σας, αλλά θέλατε να επεκταθώ λίγο. Για να απαντήσω λοιπόν πρέπει να επαναλάβω ζητήματα τα οποία ξέρω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά είναι μια γραφειοκρατία. Όμως διοικείται από κυβερνήσεις, 190 συν κυβερνήσεις, και πολλές φορές τα, οι φορείς μας, οι, οργανισμοί μας διοικούνται από διαφορετικούς ε, από διαφορετικούς διαφορετικά, από διαφορετικούς πολιτικούς φορείς και πολλές φορές υπάρχουν ασυνέπειες μεταξύ των διαφόρων οργανισμών του ΟΗΕ. Είτε είναι, ε, από τη μία πλευρά έχουμε ας πούμε την ε, Διεθνή Οργανισμό Τροφίμων, από την άλλη πλευρά έχουμε ε, οργανισμούς ανθρωπινών δικαιωμάτων και πολλές φορές δημιουργούνται πράγματι ασυνέπειες. Και δεν υπάρχει συντονισμός μεταξύ των διαφόρων οργανισμών και διευθύνσεων και υποδιευθύνσεων. Αυτό συμβαίνει και σε μια κυβέρνηση που πολλές φορές υπουργεία δεν... Η δουλειά μου είναι να αποφύγω αυτήν την ε, ασυνέπεια και αυτή την έλλειψη συντονισμού. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή τα πράγματα αλλάζουν. Προ το καλύτερο. Και επίση θέλω να τονίσω, εάν ο Πασκάλα Μη, ο γενικό Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, καθόταν στη θέση μου, θα ήταν ο πρώτο που θα έλεγε ότι ο ΠΟΕ πρέπει να κάνει περισσότερα για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, Ιδίω όσον αφορά τι ποσοστώσει και του δασμού. Ο Πασκάλα Μη έχει προσπαθήσει να πείσει τα μέλη του ΠΟΕ να αναλάβουν τις δικές τους ευθύνες πιο σοβαρά. Όμως, όπως πάντοτε, εμείς ως γραφειοκράτες λειτουργούμε μέσα σε ένα πολιτικό περιβάλλον. Τώρα, αλλάζει αυτό. Καταρχάς, το γεγονός ότι είπε τους αρμοστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ότι ο ειδικό εισηγητής ε, έχουν τέτοια μεγάλη επιρροή στην συζήτηση για την επιστική βοήθεια και ασφάλεια δείχνει ότι κάτι αλλάζει και ότι το θέμα των τροφίμων και του επιστητισμού έχει γίνει κυρίαρχο θέμα συζητήσεων και προσπαθειών και ότι συζητείται στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δείχνει ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει προς το καλύτερο γιατί υπάρχει μεγαλύτερη επιρροή. Όσον αφορά τώρα, αν υπάρχει μια γενική μετατόπιση προσεγγίσεων, θα ήθελα να σας ζητήσω τον Οκτώβριο να συμμετάσχετε στην Επιτροπή Επισητιστικής Ασφάλειας για στη δεύτερη ετήσια συνεδρίασή της με τη νέα σύνθεση για να ε, διαπιστώσετε ότι θα συζητήσουμε την ατζέντα μας η οποία περιλαμβάνει όλα αυτά τα θέματα που σας αφορούν την, την ασάφεια και την αβεβαιότητα τροφίμων την επάρκεια ύδατος την μικροκαλλι... μικρού μικρά... κλίμακας είναι λοιπόν μια νέα μορφή διακυβέρνησης αυτό το φόρουμ που πιστεύω ακράδαντα ότι θα βοηθήσει τα συμφέροντα των παραγωγών. Στον κύριο Μπέρμαν πάλι απαντώ. Εάν αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια νέα καμπή της γεωργίας, είπα στην ενακτήρια ομιλία μου ότι έγιναν πάρα πολύ μεγάλα σφάλματα τα τελευταία 50 χρόνια στην ευρωπαϊκή και βορειοαμερικανική αγροτική πολιτική. Και αυτό οδήγησε σε μια έξοδο τεράστια από την Ήπεθρο προσταστικά κέντρα. Όπως είπατε, η γεωργία, η αγροτική ανάπτυξη είναι προ, προ, θέμα προτεραιότητα στην ημερήσια διάταξη όλων των κυβερνήσεων. Βλέπουμε τεράστιες αλλαγές προσεγγίσεων όσον αφορά τη σημασία της αγροτικής ανάπτυξης ε, για τη βοήθεια των αστικών ε, περιοχών, για την ενίσχυση της εκτινοτροφίας και διατήρηση ε, των των κοπαδιών κλπ. Μέσα στο πλαίσιο βεβαίως των καιρικών αλλαγών, της αλλαγής του κλίματος, της ευαβαιότητας του καιρού και τα προβλήματα του περιβάλλοντος αυτό που βλέπουμε συνεχώς και είναι πολύ αισιόδοξο είναι νέοι άνθρωποι, νέοι σε ηλικία να ασχολούνται με τη γεωργία παρά να είναι όλη η παραγωγή μιας μεγαλύτερης ηλικίας αν θέλετε, ένας γερασμένος πληθυσμός. Αυτό μας δίνει ελπίδες. Νομίζω ότι πρέπει να ολοκληρώσω και καταλήγω λέγοντας ότι η επικεντρωμένη πολιτική στους ανθρώπους, η πολιτική που επικεντρώνεται στους ανθρώπους και στην επιστημιστική ασφάλεια είναι το, το έργο το οποίο πρέπει να εκτελέσουμε. Πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στους παραγωγούς και σε όλους τους ενδιαφερόμενους να οργανωθούν έτσι όπως θέλουν, έτσι όπως πιστεύουν ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για αυτούς. Και σας παρακαλώ να μας υποστηρίξετε στις προσπάθειές μας. Ωραία. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Σισόκο, αλλά παρακαλώ α στηρίσουμε το χρόνο αγόρευση. Παρόλο που είναι συναρπαστικό το θέμα, δεν πρόκειται να ολοκληρώσουμε ποτέ αν όλοι υπερβαίνουν συστηματικά το χρόνο αγόρευση. Το θέμα των ομάδων βοσκών το έθιξα και εγώ. Σας είπα ότι η Αφρική βιώνει μια κρίση ταυτότητας ε, σε ό,τι αφορά τα, τις αναφορές της αλλά και τη στρατηγική της το αφρικανικό πλαίσιο και οι εμπειρογνώμονες που είναι κυρίως παιδιά χωρικών είναι πεπισμένοι ότι είναι επιρχαιωμένε οι καλλιέργειές μας και ότι θα πρέπει να μοιάσουμε όλο και περισσότερο στην Ευρώπη. Αυτή η νοοτροπία είναι βαθιά ριζωμένη. Δεν μπορούμε να τους ε, φέρουμε εδώ στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων γιατί δεν έχουν σχέση πια με αυτούς που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα στην πράξη. Το πρόβλημα πραγματικά είναι σημαντικό άλλοι αυτοί που ετοιμάζουν τις πολιτικές και τα χαρτιά, η πολιτική και άλλη πραγματικότητα των χωρικών. Το θέμα είναι ποιος θα χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη της υπαίθρου. Η ανθρώπινη πόροι και η φυσική και η χρηματοπιστωτική είναι επαρκής για να καλύψουν τα θεμελιώδη προβλήματα. Και η συνεργασία δεν μπορεί παρά να διαδραματίσει ελάχιστο ρόλο, γιατί πώς είναι δυνατόν να πιστούμε ότι οι άλλοι θα πρέπει να έρθουν ε, και να μας βοηθήσουν να τους ανταγωνιστούμε, ακόμη και να τους ξεπεράσουμε. Δεν έχει νόημα κάτι τέτοιο, γιατί οι διεθνεί διαπραγματεύσει είναι ένα συσχετισμό δυνάμεων. Δεν μπορούμε να ζητούμε από του Ευρωπαίους να είναι τόσο ευγενικοί και γενναιόδοροι και να αγαπούν τόσο την Αφρική ώστε να εθετήσουν ε, πολιτικέ υπέρ τη Αφρική. Δεν έχει νόημα κάτι τέτοιο. Είναι ευθύνη τη Αφρική να βρεθεί σε ισχυρή διαπραγματευτική θέση απέναντι στην Ευρώπη. Και είμαστε πεπισμένοι ότι είμαστε συμπληρωματικοί ως προς την Ευρώπη. Κύριε Μποβέ, όταν ιδρύθηκε ο ΠΟΕ, αμέσως η Κνουσέντ έμεινε ε, κατά μέρο γιατί ήταν ένα όργανο των Ηνωμένων Εθνών όπου οι χώρες έχουν περίπου τις ίδιες ε, ευθύνες και δυνατότητες ε, και ισχύ. Αν η Αφρική δεν κινητοποιηθεί και δεν γίνει πιο ορατή, στις ε, διεθνείς διαπραγματεύσεις, όλα θα γίνουν εις βάρος μας. Δεν μπορούμε να κατηγορούμε τους άλλους, ενώ εμείς οι ίδιοι δεν ε, ασχολούμαστε με τα προβλήματά μας. Και αφήνουμε τα προβλήματά μας ε, στα χέρια των άλλων, θεωρώντας ότι θα μας τα επιλύσουν. Θα σας δώσω και ένα άλλο παράδειγμα. Στις διαπραγματεύσεις για την διαμόρφωση της γεωρικής πολιτικής της Δυτικής Αφρικής, κινητοποιήθηκαν οι χωρικοί και μάλιστα στην γεωργική πολιτική που υπέγραψαν οι αρχικοί κρατών συμπεριλάβαμε την εξασφάλιση της γεωργικής κυριαρχίας και ότι η, γεωργική, η οικογενειακή καλλιέργεια είναι ως λίθος της γεωργικής πολιτικής. Όταν όμως ολοκληρώσαμε αυτή την προσπάθεια, η Παγκόσμια Τράπεζα και όσα θεωρήθηκαν ως ηγέτες ε, της ε, ε, σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση αυτού του, αυτού του πλαισίου γεωργίας. Και αυτοί οι δύο θεσμοί ε, γονάτισαν την, την γεωργία στην Αφρική. Γιατί αυτοί οι δύο διεθνείς οργανισμοί μας έφεραν σε κατάσταση που τελικά δεν μπορέσαμε να χρηματοδοτήσουμε την ΚΑΤΕΚ. Πώς θέλετε λοιπόν να προχωρήσουμε αν έχουμε αυτές τις ωραίες ιδέες αλλά δεν μπορούμε να εκταμιεύσουμε τους πόρους ώστε να τις υλοποιήσουμε. Γιατί πάντα ζητούμε από την Ευρώπη, από τι Ηνωμένε Πολιτείε, από του άλλου, ακόμη και για την εκπόνηση των πολιτικών μα, χρειαζόμαστε πάντα να έρθει κάποιο από έξω και να μα τι χρηματοδοτήσει. Αυτό είναι. Αυτό είναι ο πρώτο περιορισμό. Πώ είναι δυνατόν να περιμένουμε από άλλου να έρχονται με κονδύλια και με εμπειρογνώμονε για να μα βοηθήσουν, ότι ενώ οι δικοί μας εμπειρογνώμονες βρίσκονται σε όλους τους οργανώσεις. Εκεί είναι που χωλαίνει η Αφρική. Εκεί είναι που δεν καταλαβαίνει ότι εμείς δίνουμε λαβή στους άλλους για να κάνουν ό,τι θέλουν μαζί μας. Η πρώτη κυριαρχία είναι η επισητιστική, αλλά και η δυνατότητα να εκπονεί κανείς μόνος του την πολιτική του, τη στρατηγική του, τα οράματά του. Όταν είμαστε ανίκανοι ακόμη και αυτό να κάνουμε, να εκπονούμε τις πολιτικές μας, πώς είναι δυνατόν να διεκδικούμε δικαίωμα ύπαρξης. Και στον ΩΣΑ η, δική μας οργάνωση είναι ανίκανη να απορροφήσει και τον προπολογισμό που έχουμε στη διάθεσή μα. Οπότε προ τι να τρέχουμε και να ζητούμε αναπτυξιακά κονδύλια, αν εμεί οι ίδιοι τα χρήματά μα δεν μπορούμε καν να τα απορροφήσουμε και να τα καταναλώσουμε. Αυτό είναι το θεμελιώδη ζήτημα. Αυτό που περιμένουμε εμεί είναι να λάβουμε το πεπρωμένο στα χέρια μας, να λάβουμε τη μοίρα μας στα χέρια μας και να εξασφαλίσουμε τους πόρους για να καθίσουμε στην Τράπεζα να διαπραγματεύσουμε, να σκεφτούμε, να συνεννοηθούμε, να συμφωνήσουμε και να δράσουμε. Και να έχουμε και μια συνένεση για τους ρόλους και τις ευθύνες. Να τα βρούμε πρώτα μεταξύ μας και μετά να συναντήσουμε τους άλλους. Γιατί αυτό έκαναν και άλλοι για να αναπτυχθούν. Και αυτό συνεχίζουν να κάνουν. Θα πρέπει να τους μιμηθούμε. Η Ντόχα έχει ε, διαφορές Ευρώπης Ηνωμένων Πολιτειών ε, και αντιδικίες για τη Γεωργία. Γιατί, ε, φυσιολογικό είναι, γιατί κάθε περιοχή προσπίζει τα ζωτικά της συμφέροντα. Εμείς δεν έχουμε αντιδικία με κανέναν. Συμφωνούμε για τα πάντα, αλλά δεν συμφωνούμε για τίποτα. Θέλουμε κάτι που να μας ανήκει και να το προσπίσουμε. Αυτό είναι το σημαντικό. Και θα ήθελα να πω στους ευρωβουλευτές το εξής. Έχουμε τις ισομερείς ε, διασκέψεις και συνελεύσεις. Στις συνελεύσεις αυτές ε, που γίνονται στις χώρες ακές, ελάτε, πάτε στους χωρικούς, δείτε την καθημερινότητά της, την καθημερινότητά τους ε, και μην αρκείστε σε μελέτες και αξιολογήσεις. Ελάτε επί τόπου, ώστε να δούμε πόσο εμπλέκονται στην κατάσταση οι βασικοί πρωταγωνιστές. Αυτό είναι σημαντικό αν θέλουμε να βοηθήσουμε κάποιους. Το πρώτο στοιχείο της βοήθειας είναι η αναγνώριση και ο σεβασμός αυτών που θέλουμε να βοηθήσουμε. Δεν μπορεί κανείς να με θεωρεί ως αντικείμενο και να με βοηθάει ε, να αναπτυχθώ. Θα πρέπει να με αναγνωρίσει και να με θέσει στο επίκεντρο της συζήτησης. Αυτό, αυτή είναι η έκκλησή μας προς όλες τις ομερείς ε, διασκέψεις και τη συνέλευση ΑΚΕ. Να αρθούν οι ευρωβουλευτές τόπου να συνομιλήσουν με τους χωρικούς, για να δουν ποια είναι η πραγματικότητά τους για να, και να δείτε πραγματικά αν η βοήθεια που στείλατε αξιοποιήθηκε, πώς χρησιμοποιήθηκε. Θα έχουμε τους τοπικούς ε, ερετούς, τους εκπροσώπους της κυβέρνησης, αλλά και τους χωρικούς. Οπότε θα είναι σαφής η συζήτηση και ξεκάθαρη. Γιατί έτσι πραγματικά θα αξιοποιηθούν τα εκατομμύρια που θέλετε να διαθέσετε για την Αφρική. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό ακόμη. Ε, με ρωτήσατε τι συνέβη ακριβώς. Όταν ε, οι αστεί θέλησαν να ανατρέψουν την κυβέρνηση. Φυσικά επικράτησε πανικός. Άνοιξαν τα σύνορα για να εισέλθουν εισαγωγέ μαζικά και δόθηκαν και επιδοτήσεις. Και σε πολλές χώρες δεν είχαμε επιδοτήσεις, ε, θεσμοθετήθηκαν επιδοτήσεις. Αλλά τη στιγμή της εκπόνησης της γεωρικής πολιτικής, της χάραξης της γεωρικής πολιτικής, είχαμε κοινό εξωτερικό δοσμολόγιο με την Ένωση και την Οικονομική και Νομισματική Ένωση της Αφρικής με χαμηλούς δεσμούς, γιατί το επίπεδο προστασίας των χωρικών μας ήταν το ασθενέστερο. Και με τις διαπραγματεύσεις ζητήσαμε με τη βοήθεια της Νιγηρίας να αυξηθεί αυτή η προστασία στα σύνορα. Αυτό που έκαναν όλε οι μεγάλε δυνάμει άλλωστε για να προστατεύσουν τη γεωργία του. Προστασία στα σύνορα. Αυτό επιδιώξαμε και εμεί. Από 20% να ανέλθουμε στο 50%. Και οι χώρε ε, που καλουπώνονται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα, οι κυβερνήσεις ε, των μπλόκαρων και τελικά πέσαμε στο 30% από το 50% που ζητήσαμε. Και μέχρι στιγμής δεν καταφέραμε ούτε καν αυτό το 30% να εφαρμόσουμε. Γι' αυτό δεν είχαμε επιτυχία. Γιατί δεν θέλουμε μόνο να υπεδοτούμε τις ε, εισόδου. αλλά θα πρέπει στη γεωργική πολιτική που χαράζουμε να εξασφαλίσουμε την προστασία και της περιφερειακής αγοράς. Ευχαριστώ και θα ήθελα να δώσω το λόγο στην πρόεδρό μας, την κυρία Εύα Νομίζω ότι τέθηκαν πια οι βασικοί όροι των προβλημάτων. Διαπιστώσαμε ότι δεν καταφέραμε να επιλύσουμε το πρόβλημα της πείνας στον κόσμο που έχει επιδεινωθεί από το 2008 παρά την ε, συνειδητοποίηση των διαστάσεων του προβλήματος από τον ΟΗΕ και νομίζω ότι είναι και η ώρα να δώσουμε και πάλι τη δύναμη στους ε, πολιτικούς. Δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε, δεν μπορούμε να αγνοούμε το ρόλο της κερδοσκοπίας και το παιχνίδι που γίνεται. Και μάλιστα ένα παράδειγμα είναι οι μεγάλες ξηρασίες που είχαμε το 2010 στην Ρωσία. Οι κερδοσκόποι και μάλιστα η Μπιανκόρ κυρίως είχαν ε, προεξοφλήσει μια μεγάλη αύξηση των τιμών. Δεν είχαμε σπάνι τελικά, δεν είχαμε έλλειμμα και ε, η Υπουργή Γεωργίας Ανήγγελο δεν θα υπήρχε σπάνι. Μετά από την αναγγελία αυτή ο Πούτιν απαγόρευσε τις εξαγωγές λέγοντας ότι υπάρχει έλλειψη σύτου. Οπότε η Γενκόρ επικαλέστηκε ανωτέρα βία και κατήγγειλε συμβάσει που θα ήταν επιβλαβής ε, για αυτήν αν είχαν εξελιχθεί κανονικά οι τιμές. Και αυτή η τεχνητή απόφαση μη εξαγωγή ρωσικού ΣΥΤΟΥ οδήγησε σε εκτείναξη των τιμών του σίτου. Και μάλιστα είχαμε θανάτου στην Αφρική, αλλά η Γκενκόρ ε, κερδοσκόπηση, κέρδισε πολλά χρήματα και μάλιστα δεν πλήρωσε καν φόρου για αυτά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και η κατάσταση για τα αποθέματα σιτηρών το 2010 είχε ω εξή. Τα αποθέματα των σιτηρών αυξήθηκαν το 2010. Δεν υπήρχε κανένα έλλειψη. Κάτι που δείχνει σαφέστατα ότι δεν υπάρχει καμία βούληση ελέγχου της κερδοσκοπίας. Και αυτό διαπιστώσαμε και στην κερδοσκοπία με το δημόσιο χρέος έχουμε κάποιες χώρες που είναι θύματα της κερδοσκοπίας του δημοσίου χρέους τους. Και, και παρόλα αυτά υπάρχει, ε, είναι κατά την εξάλληψη των CDS. Οπότε, τι γίνεται, Ποιος είναι, ποιος είναι ο σχετισμός δυνάμεων μεταξύ του χρηματοπιστωτικού κόσμου, των κανόνων και των πολιτικών που εφαρμόζουμε. Είναι πολύ σαθρή αυτή η κατάσταση και νομίζω ότι εμεί ω πολιτικοί έχουμε ευθύνη να θέσουμε επιτάπητο σε όλα αυτά τα προβλήματα από κοινού μαζί σα που είστε οι πρωταγωνιστέ. Γιατί μόνο εμεί θα μπορέσουμε να διορθώσουμε αυτή την κατάσταση. Δεν θα πρέπει λοιπόν να εθελοτυφλούμε, ούτε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μα. Δεν θα τα καταφέρουμε αν δεν ε, ε, ξανασκεφτούμε το θέμα της αναπτυξιακής βοήθειας και του ρόλου της Αφρικής. Και αναφέρθηκε μια μεγάλη αλήθεια, ότι το ίδιο το μέλλον μας θα εξαρτηθεί από το μέλλον της Αφρικής και από την εξασφάλιση του μέλλοντος της Αφρικής, γιατί το τα πεπρωμένα μας, οι μοίρες μας είναι αλληλένδετες. Θα περάσουμε τώρα στο δεύτερο πάνελ, στο οποίο θα εμβαθύνουμε σε όλα αυτά τα θέματα. θα ήθελα να παρακαλέσω τους πέντε προσκεκλημένους του δεύτερου πάνελ να ανέβουν στο Προεδρείο, παρακαλώ. για Και τώρα θα συζητήσουμε για δύο ζητήματα που έχουν εξέχουσα θέση και στο ψήφισμα που υιοθέτησε το Ευρωκοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα. Κερδοσκοπία για τα βασικά αγαθά και η αρπαγή των γεών. Τα δύο αυτά ζητήματα, προϊόντα της παγκόσμιας τη παγκοσμιοποίηση τη δημοσιονομική και τη οικονομική είναι αφιλεγόμενα ζητήματα μεταξύ των οπαδών τη απελευθέρωση των οικονομικών συναλλαγών από τη μια και τη καλύτερη διευθέτηση των αγορών από την άλλη. Σε ό,τι αφορά την κερδοσκοπία, το Ευρωκοινοβούλιο στο ψήφισμά του ζήτησε κυρίω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-μέλη και τον G20 να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για να αναχαιτήσουν την κερδοσκοπία σε σχέση με τα δημητριακά και τα τρόφιμα. Το ζήτημα του διακανονισμού είναι πολύπλοκο από πολιτική άποψη, διότι υπάρχουν ισχυρέ ομάδε πίεση και συμφερόντων εδώ. Και από τεχνική άποψη, διότι θέλουν να διευθετηθούν οικονομικέ συναλλαγέ, οι οποίε αρχικώ επιτρέπουν στι επιχειρήσει τη πραγματική οικονομία να αποφύγουν κινδύνου και να κερδοσκοπούν. Αλλά στο μέλλον αυτό δεν θα είναι δυνατό. Οι, οι επενδυτέ δεν θα μπορούν πλέον να στραφούν στι κερδοφόρε αγορέ. Στη συζήτησή μα εδώ έχουμε δύο εμπειρογνώμονε, τον κύριο Πιέρ Ζακέ, ο οποίο είναι επικεφαλή οικονομολόγο στον στον Γαλλικό Οργανισμό Ανάπτυξης και ο οποίος ανέλαβε ε, από την Γαλλική Δημοκρατία τον ε, Ιανουάριο 2011 ε, να εξηγήσει στο G20 τι μπορεί να γίνει με τη δικήμανση των γεωργικών τροφίμων προϊόντων στην αγορά τη γεωργική. Θα θέλαμε λοιπόν να λάβουμε τα συμπεράσματα τη μελέτη του. Ο δεύτερο εμπειρογνώμονά μα είναι ο Μάρκο Λίβιε Έρμαν, ο οποίο είναι υπεύθυνο για την πολιτική οικονομική δικαιοσύνη ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση και εργάζεται για την Oxfam International, η οποία ξεκίνησε πρόσφατα μια μεγάλη εκστρατεία για την επισητιστική ασφάλεια και για την κερδοσκοπία. Τι μπορεί να κάνει επίση η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν αναχαιτήσει. Αυτό είναι από τα ζητήματα που και εμά μα απασχολούν κατά προτεραιότητα. Κύριε Ζακέ, σα δίνω το λόγο για 10 λεπτά. Euh, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ για αυτή την πρόσκληση ώστε να σας παρουσιάσω κάποιες παρατηρήσεις μου σε αυτήν την ημερίδα και να συμμετάσχω στην άλλη σας συζήτηση. Σε σχέση με τα εισαγωγικά σας σχόλια θα πρέπει να διαχωρίσω κάπως τη θέση μου, διότι η αποστολή που μου ανέθεσε ο πρόεδρος της, Δημοκρατίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας ήταν να δω τι μέσα διαθέτουν οι αναπτυσσόμενες χώρες ώστε να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους που προκαλούν η διακύμανση των τιμών των γεωργικών τροφίμων. Οπότε δεν ασχολούμαι τόσο με την κερδοσκοπία αυτή καθεαυτή όσο του κινδύνου, οι οποίοι είναι πολλαπλοί και δεν έχουν να κάνουν μόνο με την μεταβλητότητα των τιμών. Ε, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σα τρία βασικά μηνύματα. Πρώτον, επίγει από τον κόσμο που αντιμετωπίζουμε τις κρίσεις να περάσουμε σε έναν κόσμο όπου μαθαίνουμε να διαχειριζόμαστε τους κινδύνους. Είναι πολύ διαφορετικά τα δύο αυτά πράγματα, διότι το να διαχειρίζεται κανείς τον κίνδυνο σημαίνει ότι βρίσκεται εκτός κινδύνου, πρωτού προκύψει μια κρίση. Ενώ όταν διαχειρίζεται μια κρίση σημαίνει ότι αντιδρά σε πράγματα τα οποία είναι απρόβλεπτα. Δεν... Και αυτό είναι πολύ δαπανηρό συνήθω. Δεν μπορεί επίση να αντιδράσει άμεσα και αυτό προκαλεί ακόμα υψηλότερο κόστος. Αυτό είναι που, που βλέπουμε να συμβαίνει σήμερα. Σε ό,τι αφορά τη γεωργία και την επιστημιστική ασφάλεια, περνούμε το χρόνο μας να τρέχουμε πίσω από τα, συνέπειε τη πιο πρόσφατης κρίση. ενώ θα έπρεπε να μπορούμε να προλαμβάνουμε. Το δεύτερο μήνυμα είναι ότι χρειάζεται διάρκεια και να έχουμε υπόψη ότι οι κίνδυνοι είναι πανταχού παρόντε. Κίνδυνοι υπάρχουν σε όλα τα σημεία του πλανήτη. Στην οικονομία επίση. Δεν μπορεί κανεί να επενδύει στην ε, ανάπτυξη εάν υπάρχει και κίνδυνο ε, πλήρου απώλεια των ενεργητικών. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε υπόψη ότι οι γεωργοί στι αναπτυσσόμενε χώρε, εάν δεν μπορέσουν να αντιμετωπίσουν του κινδύνου, ουσιαστικά γίνονται θύματα. Δεν μπορούν να επενδύσουν, δεν μπορούν να αναπτύξουν τι δυνατότητέ του. Υπάρχει λοιπόν και εδώ ένα θέμα πλούσιο που μπορούμε να εξερευνήσουμε. Και ένα τρίτο μήνυμα είναι ότι δεν υπάρχει καμία θαυματουργή λύση. Δεν υπάρχει ένα εργαλείο το οποίο να είναι κατασκευασμένο ως διαμαγείας, το μπορεί, μπορεί κανείς να επικαλεστεί και να μπορεί να αναχαιτήσει όλους τους κινδύνους. Όχι, χρειάζονται ολοκληρωμένες προσεγγίσεις, ώστε να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένους κινδύνους ε, με τοπική εμβέλεια που δεν είναι ίδιοι σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται πολλή δουλειά και μεγάλη ε, πολυμορφία στην προσέγγιση μα. Θα σταθώ στο καθένα από τα μηνύματα αυτά και θα ξεκινήσω με το πρώτο. Θα μιλήσω λίγο για το τι γίνεται ε, στο πλαίσιο το σημερινό. Γιατί τρέχουμε πίσω από τι κρίσει στην πραγματικότητα και είναι πρόβλημα αυτό σε σχέση με την επιστημιστική ασφάλεια. Κάτι που και προηγουμένω αναφέρθηκε για του αριθμού, τον έκταση του υποσυτισμού. Γνωρίζαμε την, κρίση, την κατάσταση αυτή και πριν τη σημερινή κρίση. Πρόβλημα αποσυτισμού και επιστημιστική ασφάλεια υπήρχε και πριν την κρίση. Η κρίση σημαίνει ότι ξυπνήσαμε βέβαια όλοι, αλλά είναι κάπως κρίμα που δεν μπορέσαμε πριν την κρίση να προβλέψουμε επαρκή μέτρα, ώστε να βεβαιωθούμε ότι θα σχηματιστούν απαραίτητες, απαραίτητα αποθεματικά. Να προσδώσουμε στη γεωργία και όλο τον γεωργικό κόσμο τα μέσα που χρειαζόταν για να αντιμετωπίσει τα θέματα αυτά. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη καθυστέρηση και οι προκλήσει τη σημερινή κρίση τι μα μαθαίνουν, τι μα διδάσκουν συλλογικά. Ότι θα πρέπει τώρα άμεσα να σηκωθούμε στα πόδια μα και να επενδύσουμε στο μέλλον. Αλλά το πρόβλημα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε για αυτέ τι μελλοντικέ επενδύσει είναι ότι θα πρέπει να αυξήσουμε παρκώ την γεωργική παραγωγή και να βελτιώσουμε και την ε, διοργάνωσή μα. Κατά τρόπο, ώστε τα τρόφιμα να διανέμονται εγκαίρως στους πληθυσμούς που τα χρειάζονται πρωτίστως. Η δημογραφική εξέλιξη και οι οικονομικές εξελίξεις και οι επισητιστικές καθώς και οι επιπτώσεις από τις κλιματικές αλλαγές και τις φυσικές καταστροφές σημαίνουν ότι υπάρχει πραγματικό πρόβλημα προσφοράς το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη στην κατάρτιση των γεωργικών μας πολιτικών. Άρα χρειάζεται επένδυση στη γεωργική πολιτική, βιώσιμη γεωργική πολιτική, ώστε να ληφθούν υπόψη σοβαρέ προκλήσει που προσωπούν το περιβάλλον και οι κλιματικέ αλλαγέ και η διοικητική μα διοργάνωση. Να μην υπάρχει διασπάθηση μόνο πόρων όπω γίνεται παντού στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Είναι θέμα διοργάνωση όλο αυτό. Εδώ μπορούμε να συμβάλλουμε τα μάλλα στην ανάπτυξη τη προσφορά. Το θέμα αυτό του περάσματο από τη διαχείριση κρίσεων στη διαχείριση κινδύνων είναι εξαιρετικά σημαντικό. Νομίζω ότι έχει υποτιμηθεί στις προσεγγίσεις μας ως σήμερα. Ακόμη και στην αναπτυξιακή μας προσέγγιση. Τον να επενδύουμε αναλαμβάνοντας κινδύνους είναι κάτι που το κάνουμε. Αλλά όσο καλύτερα καταλαβαίνουμε τους κινδύνους και τους αναλύουμε, τόσο ασφαλέστερα σχέδια μπορούμε να καταρτήσουμε. Κατά δεύτερον, οι κίνδυνοι αυτοί, όπως είπα, είναι πανταχού παρόντες και διαρκείς, μόνιμοι. Αυτό τι σημαίνει θα έπρεπε να δούμε και τον, την κερδοσκοπία καθώς και την ε, το πιστοτική διάσταση τη γεωργική αγορά. Θα πρέπει εδώ να το σκεφτούμε αυτό. Η διευθέντηση των αγορών είναι απαραίτητη. Σα καλώ να δούμε την διάκριση μεταξύ τη κερδοσκοπία από τη μια και έπειτα τη συμπεριφορά των κερδοσκόπων από την άλλη. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Διότι η κερδοσκοπία είναι χαρακτηριστικό του ανθρώπου από τότε που άρχισε να σκέφτεται το μέλλον του. Το να κερδοσκοπεί κανεί, να προσπαθεί να προεξοφλήσει, να ε, κάνει προβλέψει είναι κάτι που όλοι το έχουμε στο αίμα μα. Αυτό δεν είναι κάτι το αρνητικό. Είναι ένα χαρακτηριστικό ανθρώπινο τη ανθρώπινη φύση σε σχέση με τα ζώα λόγου χάρη στα κείμενα που υπάρχουν στα χέρια μας σε σχέση με την ιστορία των κινδύνων βλέπουμε τον ε, πρώτη στο ρόλο που έχει ε, διδραματίσει η δυνατότητα να σκεφτεί κανεί το μέλλον στην όλη οικονομική ανάπτυξη του κόσμου και τη ανθρώπινη κοινωνία. Αυτό μου φαίνεται λοιπόν ε, απαραίτητο από την άλλη. Η συμπεριφορά των κερδοσκόπων, ωστόσο, είναι κάτι το οποίο πρέπει να διευθετηθεί. Το πρόβλημα λοιπόν που έχουμε σήμερα δεν είναι η κερδοσκοπία αυτή καθεαυτή ω χαρακτηριστικό. Είναι ότι η κερδοσκοπία ε, εξασκείται σε ένα πλαίσιο συμπεριφορά που δεν είναι το κατάλληλο. Θα πρέπει λοιπόν να βεβαιωθούμε ότι η συμπεριφορά των κερδοσκόπων μπορεί να εξυπηρετεί την κοινωνία. Και υπάρχουν τέτοιοι τομεί εκεί όπου μπορούν να αναλάβουν κινδύνους που οι άλλοι θέλουν να αποφύγουν. Αυτό είναι κάτι που θα βοηθήσει τους χωρικούς ε, να ε, αποφύγουν συγκεκριμένους κινδύνους. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς λειτουργούν οι αγορές και τη συμπεριφορά της κερδοσκοπίας που είναι μια από τις βασικές συμπεριφορές του ανθρώπου να τις θέσουμε στην υπηρεσία των κοινωνικών μας αναγκών όπως της επιστημιστικής ασφάλειας. Το, το οποίο λοιπόν θα θέλαμε να είναι μαύρο ή άσπρο, να είναι νύχτα ή μέρα ε, για να ξεχωρίζουμε εύκολα τα πράγματα. Όμως ε, οι κρατικές πολιτικές και οι δημόσιες πολιτικές θα πρέπει να δουν τα πράγματα αγκρί και να αναλάβουν τη διαθέτηση των αγορών. Εδώ δεν μιλάμε για κάτι που συμβαίνει άπαξ και σε πλαίσια τα οποία είναι ήδη προκαθορισμένα. Όχι, όλα αυτά εξελίσσονται διαρκώ. Είναι μεταβαλλόμενο το τοπίο. Οι φορεί τη αγορά βρίσκουν τον τρόπο να δράσουν σε ένα δεδομένο νομοθετικό πλαίσιο και προλαβαίνουν τις ε, νομικές ε, αλλαγές. Οι νομοθέτες συνεχώς καθυστερούν. Άρα θα πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη δουλειά και σε σχέση με το ε, ίδιο το έργο των ε, ηθινόντων και το ρόλο τους. Τώρα, για τους κερδοσκόπους. όποια και είναι τα αποτελέσματα της συμπεριφορά τους και πάλι θα υπάρχει το θέμα της διαχείριση των κινδύνων. Οι κίνδυνοι στην παγκόσμια ιστορία είναι διαρκή και μόνιμοι. Όποια τα προβλήματα, η διακύμανση των ε, γεωργικών προϊόντων λόγου χάρη τη τιμή των γεωργικών προϊόντων ήταν ένα παγκόσμιο φαινόμενο ακόμη και όταν δεν υπήρχαν τοπικέ αγορέ. Άρα θα πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε κινδύνου κινδύνου που δεν αφορούν μόνο συγκεκριμένε χώρε, αν και οι χωρικοί των απτυσσόμενων χωρών αντιμετωπίζουν μέγιστο κινδύνου που έχουν να κάνουν με τι λειτουργίε των υποδομών, με την ανεπάρκεια τη δυνατότητα δημιουργία αποθεμάτων, με τι ασθένειε, με το κλίμα, με τι τιμέ τι ίδιε Χρειάζεται λοιπόν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για να τους βοηθήσουμε να τα αντιμετωπίσουν όλα αυτά. Τρίτο μήνυμα, δεν υπάρχει μαγική λύση, δεν υπάρχει ένα θαυματουργό εργαλείο για να προστατευτούμε. Υπάρχει, όπως ξέρετε, στις χρηματοπιστωτικές αγορές, υπάρχουν μάλλον προηγμένα εργαλεία, όπως οι μετοχές, τα ομόλογα πράγματα που μπορούν να επιτρέψουν μάλλον δεν επιτρέπουν στους ε, γεωργούς να προστατευτούν από τους κινδύνους. Κάποια συγκεκριμένα προϊόντα μπορούν να τα καλύψουν για ένα διάστημα στις αγορές. Όμως ε, στις αναπτυσσόμενες χώρες αυτό που χρειάζεται είναι η ίδια η εγχώρια παραγωγή. Για το ρύζι λόγου χάρη δεν υπάρχει θέμα αγοραπολισία στι χρηματοπιστωτικέ αγορέ. Όμω για το ρύζι θα πρέπει κάτι να γίνει που δεν, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σε επίπεδο οικουμενικής λύσης, λύσης για όλους. Η αγορά των γεωργικών προϊόντων λοιπόν δεν είναι ακόμη ανεπτυγμένη, υπάρχουν θεσμικές αδυναμίες και η κίνδυνη είναι εντοπισμένη κυρίως στο τοπικό επίπεδο. Αυτό λοιπόν που είναι σημαντικό είναι να υπάρχει ένα σύστημα πολύ συλλογικό με δυνατότητα τοπικής εξέτασης των προβλημάτων να δούμε τους χωρικούς, να, τους συζητήσουμε, να συζητήσουμε με τους ίδιους τους γεωργούς και μαζί να εξεύρουμε εργαλεία για να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους. Θα κλείσω λέγοντας ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση κάπως μοναδική σήμερα, διότι ίσως τρόπον την λόγω της κρίσης το G20 ασχολείται με το θέμα της επιστητικής ασφάλειας ακριβώς τώρα. Είναι σημαντικό, το ακούσαμε, το είπε προηγουμένως ο κύριος Μποβέ. Ακόμα βρισκόμαστε στο στάδιο των λόγων. Όμω, χωρί λόγου που θα μα κινητοποιήσουν, δεν μπορεί να υπάρξει και δράση. Αυτό που έκανα λοιπόν το Τζίκο σήμερα, νομίζω, και για την επιστημιστική ασφάλεια, είναι πολύ ενδιαφέρον. Ουσιαστικά προ... εξερεύνησε πολλέ ιδέε, όπω ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στην παραγωγή, την παραγωγικότητα και τι επενδύσει. Η δεύτερη ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στη συλλογική διαχείριση κινδύνων, ιδίω για να αποφύγουμε προβλήματα όπω αυτά που ανέφερε προηγουμένω ε, ο προλαλή με, ε, με του περιορισμού τη εξαγωγή. Και έπειτα είναι απαραίτητε οι εταιρικέ σχέσει. Υπάρχουν πολλοί φορεί που εμπλέκονται στην παραγωγή τροφίμων που θα μπορούσαν να, να έχουν αποθήκευση τροφίμων και δημητριακών. Εκεί λοιπόν οι σχέσει συνεργασία, ιδίω ιδιωτικού δημόσιου τομέα, θα μπορούσαν να είναι πολύ ενδιαφέρουσε. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα που δείχνουν ότι αυτό θα έπαιζε καθοριστικό ρόλο για την επιστημιστική ασφάλεια. Αυτά ήθελα να πω για να ανοίξει η συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ. Να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Χέρμαν για 10 λεπτά. Merci, <coughs> euh, merci, madame. Euh. Ευχαριστώ κυρία Ζολή. Θα ήθελα να αρχίσω λέγοντας ότι οι εργασίες της Επιτροπής σας είναι εξαιρετική και ιδίως η έκθεση της κυρίας Τσίμερ και η έκθεσή της που ήταν υψηλής ποιότητος και η οποία υιοθετήθηκε την περασμένη εβδομάδα. Θέλω σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα να σας εξέσω τις βασικές μου ιδέες και σκέψεις και έχετε και τα περισσότερες λεπτομέρειες ε, τυπωμένες στο φυλάδιο που υπάρχει στο φάκελό σας. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε μία πολύ ευάλωτη και ευαίσθητη χρηματοοικονομική διάσταση της αγοράς τροφίμων βλέπουμε μία αύξηση και μία έκρηξη των ε, παραγόγων, των ε, χρηματοοικονομικών παραγόγων στις διεθνείς αγορές ε, μετά το 2005. Μια έκρηξη λοιπόν των προϊόντων αυτών στις χρηματοοικονομικές αγορές, των παραγόγων που καλύπτουν πάρα πολλά βασικά αγαθά. Η άλλη πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε είναι μία εμπορία αγαθών που γίνεται OTC, over the counter, δηλαδή όχι μέσω των χρηματαγορών αλλά μέσω ιδιωτικών συμβάσεων και συμβολέων και αυτή η αγορά επηρεάζει τα βασικά διατροφικά αγαθά. Αν κοιτάξετε τον πίνακα, ε, το γράφημα στα δεξιά είναι του, του, του ΦΑΟ, του ε, ε, Διεθνούς Οργανισμού Τροφίμων και βλέπετε τον, τη διακύμαση των τιμών τροφίμων από το 2002 και πέρα. Βεβαίως η κερδοσκοπία και η επιζήτηση ε, του κέρδους ήταν πάντοτε μία ανθρώπινη ε, μία ανθρώπινη πράξη, ένα ανθρώπινο ενδιαφέρον ή συμφέρον. Και εμείς πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το γεγονός. Όμως η κερδοσκοπία έχει ξεπεράσει κάθε ώρα και πρέπει να αντιμετωπίσουμε μια νέα πραγματικότητα. Λόγω αυτού αυτών λοιπόν των εκτοξεύσεων των τιμών των τροφίμων οι φτωχοί σίγονται πολύ περισσότερο. Ε, ε, εάν αμείβεσαι πολύ χαμηλά, αισθάνεσαι έντονα τις διακυμάνσεις αυτές των τιμών και την αύξηση, την ραγδαία αύξηση των τιμών. Εάν τις φτωχότερες χώρες, κερδίζει στις φτωχές αστικές περιοχές που κερδίζει 20 ευρώ το μήνα, ε, μία αύξηση της τιμής ενός βασικού αγαθού μπορεί να, σημα... να σημάνει τη διαφορά μεταξύ επιβίωσης και θανάτου. Ε, δεδομένου ότι οι επιπτώσεις αυτής της ε, κερδοσκοπίας είναι λίγα πόδινες, η Oxfam πιστεύει ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια προληπτική προσέγγιση. Η Oxfam δεν παίρνει θέση στη συζήτηση που γίνεται για την, ε, για το, την κερδοσκοπία, την άκρατη κερδοσκοπία των, μεταξύ τραπεζών και ε, κερδοσκοπικών ε, χρηματοοικονομικών οργανισμών. Ε, από τη μία πλευρά λοιπόν έχουμε τους ε, φορείς που κερδοσκοπούν και από την άλλη πλευρά έχουμε την ακαδημαϊκή κοινότητα η οποία λέει ότι η επιθετιστική δεινή κατάσταση σήμερα στον κόσμο έχει σχέση με την κερδοσκοπία στις ε, χρηματαγορές. Ότι όποια και να είναι η αιτία πρέπει να ληφθούν μέτρα διορθώσεως των αγορών. Λοιπόν, δύο λόγια για το τι πραγματικά έχει στραβώσει ε, στις αγορές βασικών αγαθών τροφίμων. Καταρχάς, η απορρίσμηση των χρηματοοικονομικών αγορών. Ε, στην προηγούμενη δεκαετία, γύρω στο 2000, το καλύτερο παράδειγμα είναι οι Ηνωμένε Πολιτείες, όπου ε, καταργήθηκαν όλες ε, οι βασικές ρήτρε ασφάλειας στις χρηματαγορές οι οποίες εμπόδιζαν την κερδοσκοπία στα αγροτικά παράγωγα. Ε, έτσι λοιπόν κερδοσκοπική, παρουσιάστηκε μια τεράστια κερδοσκοπική ροή χρημάτων στις αγορές αυτές το δεύτερο γεγονός ήταν αυτό που οδήγησε στη στρέβλωση των αγρών και το τρίτο ήταν η, ε, το ότι επετράπη η εισαγωγή πολλών παραγόγων προϊόντων στα χρηματιστήρια για την κερδοσκοπία επί ε, βασικών αγαθών, διατροφικών ε, η κατάρρευση πολλών επενδυτικών αγορών όθησε πολλούς επενδυτές στα ε, διατροφικά, ε, στις βασικές ε, αγορές και στην κερδοσκοπία βασικών αγαθών τροφίμων. Όλη αυτή λοιπόν η απορρίθμιση, η αποελευθέρωση, η κατάργηση ρητρών ασφαλείας οδήγησε στην στρεβλωμένη αγορά παραγόγων στα χρηματιστήρια. Δεν θέλω να επισέλθω σε με πολλές τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά θα σας παρουσιάσω τη νέα πραγματικότητα. Έχουμε δύο καινούριους παίκτες. Απ' τη μία ε, μαζικούς επενδυτές, θεσμικούς επενδυτές που μπήκαν στις χρηματαγορές τροφίμων Ε, και όπως λέμε στις αμερικανικές χρηματαγορές έχουμε δημιουργήσει τα ε, ορισμένα funds, ορισμένες επενδυτικούς οργανισμούς που, που ονομάζονται Massive Passives. Δηλαδή έχουν επενδύσει 250 δισεκατομμύρια δολάρια σε παράγωγα τροφίμων. Η δεύτερη πραγματικότητα είναι αυτό η κερδοσκοπική επενδυτική ροή προς τις χρηματαγορές τροφίμων. Είναι μια νέα ε, κλάση, μια νέα τάξη ε, επενδυτικών προϊόντων. Ε, όταν είχαμε μια ξαφνική κρίση, μια ξαφνική πλημμυρίδα αυτών των επενδυτικών κεφαλαίων το 1996, είδαμε μία αύξηση της τιμής των σιτηρών από 12-65% σε ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα. Ποιοι είναι τώρα λοιπόν, ποιες είναι οι επιπτώσεις για τους επενδυτές, τους ε, χρηματιστές, ε, τους ε, παραγωγούς και τους πολίτες. Ε, όλη αυτή η κερδοσκοπική δραστηριότητα βλάπτει σημαντικότητα τους καταναλωτές και τους πολίτες. Θα σας δώσω ορισμένα παραδείγματα. Μία αρνητική επίπτωση είναι ότι αυτή η μαζική συμπεριφορά, κερδοσκοπική συμπεριφορά δημιουργεί ε, τι, τιμολογικές ε, φούσκες. Δηλαδή αυξάνεται οι τιμές χωρίς λόγο και έτσι δημιουργείται μία κερδοσκοπική φούσκα η οποία μοιραία να σκάσει. Η το δεύτερο γεγονός ε, είναι ότι οι τιμές ε, των τροφίμων συνδέονται πολύ περισσότερο από στο παρελθόν με την τιμή του πετρελαίου. Δεδομένου ότι το πετρελαίο, το πετρέλαιο ανέκαθεν ήταν κερδοσκοπικό προϊόν, καταλαβαίνετε ότι το στοιχείο της κερδοσκοπίας αυξάνεται λοιπόν με αυτή τη διασύνδεση και στα τρόφιμα. Τρίτον, <clears throat> δημιουργείται μια μεγάλη βραχυπρόθεσμη στρέβλωση στις τιμές των τροφίμων και το τέταρτο είναι το hedging, δηλαδή προληπτική κάλυψη ρίσκου από τους ε, παραγωγούς γίνεται όλο και πιο ακριβή. Γίνεται όλο και πιο ε, δαπανηρή η προληπτική κάλυψη ρίσκου. Και αυτό πραγματικά είναι μια τεράστια ευθύνη, διότι αν θέλουμε να βοηθήσουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες να διαχειριστούν το ρίσκο τους, πρέπει να μπορέσουμε να αμβλύνουμε την, τις τεράστιες επιπτώσεις της κερδοσκοπίας ε, του, του, των κινδύνων που γίνεται επί του ρίσκου, επί των κινδύνων, ενδεχομένων κινδύνων. Τι ζητάει λοιπόν η Όξα. Αυτό που θέλουμε είναι βεβαίως να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους έτσι ώστε όλοι στον πλανήτη μας να μπορούν να διατραφούν, να έχουν ε, τα τρόφιμα που χρειάζονται, Θέλουμε να ενισχύσουμε τους μικροπαραγωγούς στις αναπτυσσόμενες χώρες να βοηθήσουν και να βοηθηθούν τοπικά. Για να γίνει όμως αυτό πρέπει να ενισχύσουμε τις τοπικές, ε, πρέπει να ρυθμίσουμε τις χρηματοοικονομικές αγορές, να υπάρχει μια ορθολογική ρύθμιση και αυτό μπορεί να το επιτύχουμε ως εξή. Πρώτα να αυξήσουμε τη διαφάνεια έτσι ώστε να μπορούμε να παρακολουθούμε σε πραγματικό χρόνο τις συναλλαγές που γίνονται. Ε, δεύτερον, να αντιμετωπίσουμε την πάρα πολύ συγκεχημένη και αδιαφανή αγορά των ιδιωτικών συμβάσεων και συμβολέων που δεν γίνονται μέσω χρηματοοικονομικών αγορών, τα OTC δηλαδή, over the counter, και τρίτον να ε, μπορέσουμε να ελέγξουμε τις κερδοσκοπικές ε, συναλλαγές που γίνονται. Να τις ελέγξουμε και να τις περιορίσουμε. Ε, ιδίως τις ε, κερδοσκοπικές συναλλαγές που γίνονται με βραχυπρόθεσμο όφελος που έχουν πολύ σοβαρές επιπτώσεις. Και τέλος, το ερώτημα που μας απασχολεί όλους είναι θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει η αναθεώρηση που έγινε στο, στην Wall Street στις Ηνωμένε Πολιτείες το 2010 συνάδει με, την, ε, με, την, με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο των χρηματοοικονομικών αγορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2011 ε, και ένα από τα σημαντικά ε, θέματα που θα συζητηθούν στην ατζέντα των G20 ε, στις Κάνες το 2011 πιστεύω ότι θα είναι αυτή η, η αθέμητη και αλόγιστη κερδοσκοπία που γίνεται Αυτά λοιπόν τα χρηματοοικονομικά παράγωγα προϊόντα τα οποία διαπραγματεύονται εκτός χρηματοοικονομικών αγορών και χρηματιστηρίων πρέπει να περιοριστούν, πρέπει να ελεγχθούν και πρέπει να εφαρμοστεί αυστηρά η οδηγία χρηματοοικονομική κον μέσων για να μπορέσουμε να ελέγξουμε τις ξαφνικές εκτοξεύσεις τιμών και την, ε, τις ε, ε, αρνητικές, την αρνητική κατάσταση της αγοράς, της αγοράς τροφίμων. Συζήτηση τώρα, κύριε Κέλλερ. Σας ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και τους δύο εμπειρογνώμονες για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις. Δυστυχώς θα πρέπει να μιλήσω και να φύγω γιατί Έχω και άλλες συνεδριάσεις άλλες επιτροπές. Έχω κάποιες παρατηρήσεις. Ε, κύριε Ζακέ, αν σας ε, κατάλαβα καλά, είπατε ότι έχουμε κρίση παραγωγής και θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε αυξάνοντας την παραγωγή. Διαφωνώ. Δεν έχουμε τόσο κρίση παραγωγής, αλλά περισσότερο κρίση διανομής. Και υπάρχει και θέμα υποδομών, πρόβλημα υποδομών που συμβάλλει σε αυτή την κρίση διανομής. Γιατί βέβαια η διανομή είναι και θέμα εισοδήματο. Γιατί αν αυξάνονται τιμέ τροφίμων, κάποιο δεν μπορεί να αγοράσει τρόφιμα. Παρόλο που διατίθεται τρόφιμα, αδυνατεί ο καταναλωτή να τα αγοράσει. Και το θέμα τη ε, φτώχεια ε, ε, οφείλεται όχι στο ότι δεν υπάρχουν τρόφιμα, αλλά ότι ο κόσμος δεν δίνεται να τα αγοράσει. Κερδοσκοπία ήταν ανέκαθεν πρόβλημα, όπως είπατε, αλλά ιδιαίτερα στη γεωργική αγορά η κατάσταση ήταν πολύ διαφορετική στο παρελθόν. Παλιά είχαμε τους παραγωγούς που κερδοσκοπούσαν κατά κάποιο τρόπο προκειμένου να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο. Τώρα η κερδοσκοπία δεν έχει καμία σχέση με τους γεωργούς. Γίνεται από ανθρώπους που μπορεί να μην έχουν ε, δει ένα χωράφι στη ζωή τους. Οπότε συμφωνώ με τη θέση της Oxfam για το τι δημιουργεί το πρόβλημα και μας ενδιαφέρει και η δική σας ε, άποψη γιατί είπα ότι θα πρέπει να θέσουμε την κερδοσκοπία ε, στην υπηρεσία των παραγωγών και των καταναλωτών. Συμφωνείτε με την πρόταση της ε, Oxfam. Ναι, βλέπω, νεύεται, πολύ ωραία. Και η κερδοσκοπία μπορεί να αποτελεί ένα μικρό του προβλήματος, γιατί υπάρχουν και άλλοι συντελεστές στο πρόβλημα, αλλά μπορούμε την κερδοσκοπία να αντιμετωπίσουμε σχετικά τάχιστα. Γιατί είναι ένα τεχνικό πρόβλημα με την διανομή και με τις ε, αγορές θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και άλλα στοιχεία, πολύ πιο πολύ σύνθετα. Ενώ η κερδοσκοπία είναι κάτι τεχνητό. Δεν έχει σχέση ούτε με την ανοβρία, την ξηρασία, ούτε με διάβρωση του εδάφου ούτε με κλιματικέ αλλαγέ. Είναι ένα τεχνητό πρόβλημα η κερδοσκοπία. Μπορούμε πιο εύκολα να το αντιμετωπίσουμε. Εγώ θα έλεγα ότι το πρόβλημα υπάρχει περισσότερο στη διανομή, στι υποδομέ, αλλά, όχι αλλά περισσότερο στο εισόδημα και όχι στην παραγωγή. Σας ευχαριστούμε, κυρία Κέλλερ. Ο κύριος Γκερέρο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονές μας, τον κύριο Ζακέ και τον κύριο Χέρμαν. Αναφερθήκατε και οι δύο στις παρεμβάσεις σας στο G20. Όντως, ε, έχουμε την ευκαιρία να ζητήσουμε περισσότερες πιο αναλυτικές πληροφορίες από τον κύριο Ζακέ, γιατί συμμετέχει στο γαλλικό κλιμάκιο που θα οργανώσει το φθινόπωρο, το τη διάσκεψη του G20 στις Κάνες. Είπατε ότι είναι σημαντικές και οι διακηρύξεις ε, και οι ομιλίες στον πολιτικό βίο, γιατί οι διακηρύξεις δίνουν κίνητρα, παροτρύνουν και μπορεί να απευθύνουν έκκληση και να οδηγήσουν σε πολιτική δράση. Πάντως, από την πρώτη συνεδρίαση του G20, μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσης, ακούσαμε πολλές διακήρυξεις, πολλά επίβολα λόγια, αλλά είχαμε ελάχιστα έργα σε πολλούς και διάφορους τομείς. Και δεν μιλάω μόνο για τα επισητιστικά προβλήματα. Θα μπορούσα να αναφερθώ στη φοροδιαφυγή, στους φορολογικούς παραδείσους, στις ευθύνες του χρηματοπιστωτικού κλάδου για τη τεράστια ζημία που επέφεραν στην παραγωγική οικονομία και ούτω καθεξής. Έχω την αίσθηση ότι υπήρχε μεγαλύτερη πολιτική όθηση στις πρώτες, ε, στις πρωταρχικές ε, συνεδριάσεις του G20, αλλά στο μεταξύ εξασθένησε αυτή η πολιτική όθηση. Θα ήθελα να σας επισημάνω ότι υπάρχει μια εύλογη προσδοκία από την Γαλλική Προεδρία στην επόμενη διάσκεψη του G20 να δώσει νέα όθηση συνεχίζοντας ε, την καλή αρχή που έγινε το 2008 και 2009. Δεν χρειάζεται να μας αποκαλύψετε τη στρατηγική ή τα συγκεκριμένα στοιχεία και μυστικά της επόμενης συνεδρίας του G20, αλλά μπορείτε να μας δώσετε κάποια στοιχεία σε ό,τι αφορά ε, το πρόγραμμά σας για τα αναπτυξιακά ζητήματα στην επόμενη συνεδρία του G20. Και τέλος να πω ότι είναι ίσως μια χαρμόσυνη είδηση ότι ε, περιλαμβάνεται και ο εκπρόσωπος ε, της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Συνεργασίας σε αυτό το επιτελείο της διοργάνωσης της διάσκεψης του G20. Αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο. Σας ευχαριστώ κυρία Τσίμαρ. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ τους ε, δύο μιλητές που μας ε, εξέθεσαν τα θέματα σε κατανοητή γλώσσα έτσι ώστε να μπορέσουμε και εμείς να καταλάβουμε τις ε, πτυχές της οικονομικής κερδοσκοπίας εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί η Κομισιόν επέμενε συνέχεια ότι δεν υπάρχει διασύνδεση, δεν υπάρχει σχέση μεταξύ της ε, κερδοσκοπίας της αγορές πρώτων υλών και της ε, αστάσιας της τιμές των τροφίμων. Ε, εγώ άκουσα μια διαφορετική άποψη σήμερα, ότι αυτή η διασύνδεση υπάρχει σαφώς. Τα δύο πράγματα αυτά συνδέονται και δεν υπάρχει λόγος να το αρνηθούμε. Εάν αρνηθούμε την πραγματικότητα, αυτό σημαίνει ότι δεν θέλουμε να σκεφτούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, δεν θέλουμε νέα μέτρα και δεν θέλουμε την εφαρμογή πολιτικών μέσων. Μετά λοιπόν από όλες αυτές τις πληροφορίες που λάβαμε, με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων. Είπατε ότι βραχυπρόθεσμα ή μέσοπρόθεσμα μπορούμε ενδεχομένως να ελέγξουμε τις ε, αγορές ε, παραγόγων, τις ε, αγορές βάσει ιδιωτικών συμβάσεων, τις, βραχυπρόθετα, τις βραχυπρόθεσμες συμβάσεις, τα συμβόλαια, για να μπορέσουμε προσωρινά τουλάχιστον να μειώσουμε τη ζημιά. Υπάρχει μία προθυμία, υπάρχει μία βούληση να ενεργήσουμε πολιτικά για να αλλάξουμε, όχι μόνο να ελέγξουμε προσωρινά, αλλά και να αλλάξουμε την ε, κατάσταση αυτή στις αγορές. Ξέρουμε ότι μετά το 2008 εφαρμόζονται οι ίδιες διαδικασίες ε, οι ίδιες μέθοδοι, έγινε μια μεγάλη φασαρία, μια βαβούρα, αλλά πάλι τα ίδια πράγματα ισχύουν, τα ίδια γίνονται, οι ίδιες ε, ε πράξεις παρατηρούνται, ένα εκατομμύρια άνθρωποι λιμοκτονούν ε, και όλα πάλι επανήλθαν στην προηγούμενη κατάσταση. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω ποια συγκεκριμένα μέτρα που νομίζετε ότι μπορούν να εφαρμοστούν και ποια νέα ποιες νέες δομές μπορούν να, να υιοθετηθούν, πώς μπορούμε ε, δημόσια να ακουστεί η φωνή μας ε, έντονα ότι αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει. Σας ευχαριστούμε. Κυρία Τόγια. Χωρίς μικρόφωνο, κυρία Τόγια. Ευχαριστώ τους ε, προσκεκλημένους, τους κυρίους Ζακέ και Χέρμαν, οι οποίοι έκαναν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ανάλυση. Απλώς να σταθώ σε κάτι που και η κυρία Τσίμερ σχολίασε. Εδώ φαίνεται να υπάρχει ανάγκη θεσμική και η νομοθετική για το Κοινοβούλιο να ορίσουμε εργαλεία και μπορούμε να το κάνουμε αυτό για να λάβουμε τις ευθύνες μας. Οπότε χρειάζεται προσεκτική εξετασία όλων των θεμάτων. Ας κάνουμε όμως και ένα βήμα παραπάνω, μιλώντας για τα κανονιστικά πλαίσια που να δημιουργήσουμε. Τα αναφέρατε αυτά και οι δύο. Η πρόσφατη εκθεσή μας έδειξε ότι χρειάζονται τέτοια κανονιστικά εργαλεία για να μπορέσουμε να αναχαιτήσουμε τις κερδοσκοπικές ε, συμπεριφορές. Μας είπατε ότι αυτές, τις, αυτές οι συμπεριφορές καταφέρνουν να ξεπερνούν τους κανόνες που κάθε φορά ανανεώνονται. Τι κανόνες λοιπόν να προβλέψουμε, τι είδους, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει κάτι παραπάνω. Ακριβώς γιατί εργαλεία που έχουν δημιουργηθεί για να προλάβουν κινδύνους, να τους διαχειριστούν, να αποφύγουν την εμφάνισή τους, ε, εργαλεία που διασφαλίζουν που καλύπτουν τους πρωταγωνιστές της πραγματικής ε, οικονομίας τελικά γίνονται χρήσιμα για τρίτους, όχι για τους ίδιους τους γεωργούς, όχι τους ίδιους τις φορείς της οικονομίας, αλλά και κερδοσκοπία σε επίπεδο χρηματοπιστωτικών αγορών και απλώς οικονομικών αγαθών, όπως με την κρίση το 2008. Θα πρέπει λοιπόν να μπούμε στη λογική της διαχείρισης των κινδύνων, όπως είπατε, αλλά δεν μπορούμε έτσι να δεχόμαστε ότι οι κίνδυνοι μπορούν να γίνουν ε, αντικείμενο εξέταση τι καθεαυτή. Και το θέμα δεν είναι να του διαχειριζόμαστε, αλλά το πώ εμφανίζονται. Διότι έτσι στην αλυσίδα των γεγονότων ε, μπορεί να αποσπάσει κανείς κέρδος. Τι κερδίζει κανείς λοιπόν με την ε, δημιουργία κινδύνων. Ε, πρέπει να δημιουργήσουμε λοιπόν και κάποιες δεσμεύσεις, όχι μόνο κανόνες, και να εμποδίζουμε την απόσπαση κέρδους από την εμφάνιση κινδύνων. Αν μπορούσατε λοιπόν να μα δώσετε κάποιε περισσότερε εξηγήσει για το κανονιστικό ε, πλαίσιο, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον για μένα, που δεν είμαι ακριβώ ε, ούτε μελετήτρια ούτε ερευνήτρια, αλλά νομοθέτη. Σα ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ότι στο αναλυτικό έργο του ΟΗΕ από τη ΦΑΟ και τον ΩΣΑ για το G20 σε ό,τι αφορά τη μεταβλητότητα των τιμών τροφίμων, καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως ήταν προφανές ότι η συμπεριφορά των κερδοσκόπων συνέβαλε στη μεταβλητότητα των τιμών τροφίμων. Οπότε, κατά την κρίση μας, αυτή η κερδοσκοπία είναι σημαντικό συντελεστής του προβλήματος. Και εμείς έχουμε κάποιες προτάσεις για τους πιθανούς μηχανισμούς που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, αλλά χαίρομαι που οι πολιτικοί εντοπίζουν την ανάγκη δράσης. Θα ήθελα να αναφέρω τρία είδη κινήτρων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν νομοθετικά. Καταρχήν, εξελίξεις στις κάνες από τη διάσκεψη του G20. Δεύτερη όθηση θα μπορούσε να ήταν η συζήτηση που θα γίνει στα μέσα Οκτωβρίου στη Ρώμη, συνεδρίαση της ΦΑΟ, για την ε, ρευστότητα, την μεταβλητότητα των τιμών. Και ελπίζω να βρεθεί ε, στο επίκεντρο της προσοχής ε, αυτή η διάσκεψη και υπάρχει και ένα ψήφισμα που εκπονεί αυτή τη στιγμή η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με πρόταση της Δομινικανής Δημοκρατίας και θέμα τη μεταβλητότητα των τιμών τροφίμων. Και αυτό το θέμα θα μπορούσε να τύχει της δέουσας προσοχής, γιατί και οι τρεις αυτές περιπτώσεις θα μπορούσαν να δώσουν νέα όθηση στο πολιτικό περιβάλλον για να αναλυθούν και κάποιες δράσεις. Θα ήθελα να δώσω και πάλι το λόγο σε εμπειρογνωμονές μας, πρώτα στον κύριο Ζακέ. Έχετε λίγα λεπτά για να απαντήσετε. Merci, Madame la Présidente. Ευχαριστώ. Πολλές ερωτήσεις τέθηκαν, κυρία Πρόεδρε. Συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με τις παρατηρήσεις. Θα ήθελα να διευκρινίσω ορισμένα θέματα. Κυρία Κέλλερ, είπε στην ανάλυση της ότι το πρόβλημα σήμερα δεν οφείλεται στην παραγωγή αλλά στη διανομή. Επίσης είπε ότι το θέμα της πρόσβασης στα τρόφιμα είναι θέμα περισσότερο έλλειψης χαμηλού εισοδήματος παρά παραγωγής. Είπα και εγώ στην ομιλία μου ότι σίγουρα θα πρέπει να θέσουμε ζήτημα επιμελητίας, ε, διανομής δηλαδή, αλλά υπάρχει και μία σχέση ιδιαίτερες αναπτυσσόμενες χώρες μεταξύ της ε, γεωργικής παραγωγής και του εισοδήματος. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό σήμερα να αυξηθεί η παραγωγή στις αναπτυσσόμενες χώρες, γιατί δεδομένων των διατροφικών συνηθιών, δεδομένων του δεκυβέματος των κλιματικών αλλαγών και της ε, δημογραφικής αύξησης της επόμενης πεντηκονταετίας, θα πρέπει να αυξήσουμε και την γεωργική παραγωγή και την γεωργική παραγωγικότητα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αντίφαση μεταξύ των δύο αυτών θέσεων. Και αν υιοθετήσουμε μια στρατηγική ε, προσανατολισμένη στην παραγωγή, θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι αυτό που μας ενδιαφέρει καταρχήν είναι η φόρος γεωργία, η γεωργοοικολογία, ο σεβασμός ε, των γεών, η λήψη υπόψη των κλιματικών αλλαγών και φυσικά υπάρχει το θέμα της επιμελητίας ε, της δικής διανομής συμφωνώ με πολλά από αυτά που υπόθηκαν όπως είπα και με τις συστάσεις της Oxfam σε ό,τι αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο, το κανονιστικό πλαίσιο. Οι προτάσεις της Oxfam είναι ε, σωστές, αλλά προσοχή στη δικτατορία του βραχυπρόθεσμου. Σίγουρα βιώσαμε μια πολύ ακραία κρίση με μεγάλη μεταβλητότητα τιμών τροφίμων και των γεωργικών προϊόντων, αλλά δεν θα πρέπει ε, με το πρόσχημα της άμεσης δράσης ε, να ε, στραφούμε ε, σε αυτό το θέμα και να μην ξεχνούμε ότι η κερδοσκοπία υπήρχε και από πριν. Φυσικά θα πρέπει να ε, φροντίσουμε να περιορίσουμε την υπερβολική κερδοσκοπία, αλλά η επισητιστική ασφάλεια είναι κάτι πολύ πιο ευρύ από ότι η κερδοσκοπία. Και η κερδοσκοπία δεν είναι μόνο συντελεστή. Σίγουρα ε, ο εχθρό μα είναι ο κακό κερδοσκόπο, αλλά δεν θα πρέπει να επικεντρωθούμε μόνο σε αυτό το θέμα, γιατί υπάρχει πρόβλημα πείνα στον κόσμο και επισητιστική ανασφάλεια αυτό το διαπιστώσαμε περισσότερο τα τελευταία χρόνια όταν ε, ενέκυψε ε, η κρίση. Φυσικά θα πρέπει να ρυθμίσουμε τις χρηματαγορές ε, και νομίζω ότι εδώ έχουμε δύο βασικές κατευθύνσεις που θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε. Η πρώτη είναι η ιδέα της πιστοποίησης, δηλαδή να δεχτούμε στις αγορές διαπιστευμένους μόνο φορείς και μάλιστα οι πιστοποιήσεις θα δίνονται από ανεξάρτητους οργανισμούς που θα κρίνουν τον επαγγελματισμό για να αποφύγουμε την αύξηση στην αγορά φορέων που δεν έχουν καμία σχέση με το γεωργικό επάγγελμα και τη γεωργική παραγωγή. Και ε, επίσης ε, όρια θέσης. Είναι σημαντικό να θεσπίσουμε κάποια όρια στη θέση ενός παραγωγού. Τώρα για το G20, κύριε Γκερέρο. όλες οι χώρες είναι σημαντικές και είναι δύσκολο μερικές φορές να καταλήξουμε σε, κοινή, σε κοινό όραμα που θα δημιουργήσει μία δυναμική και θα ενθαρρύνει τη δράση. Δεν νομίζω ότι ο ρόλος του G20 είναι ρόλος άμεσης δράσης. Άλλωστε δεν ε, ε, λαμβάνει δράση εθνικά το G20 γιατί σε κάθε χώρα από την κοινωνία των πολιτών, από τους πολιτικούς, από τους ιδιωτικούς φορείς, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για δράση. Πάντως, ένα κοινό όραμα και μια κοινή ηγεσία που θα, θα αναλυφθεί από την G20 θα δημιουργήσει πρόσφορες συνθήκες για δράση. Και είναι πολύ πιο εύκολο να συνεδριάζουμε μεταξύ μας και να λέμε τι, τι, τι είναι το, ποιο είναι το δέον, παρά να ε, αντιληφθούμε τους λόγους για τους οποίους ε, δεν ε, ανελήθησαν μέχρι στιγμής δράσεις. Νομίζω ότι η σωστή διάγνωση είναι το μυστικό της δράσης. Για να δημιουργηθεί αυτό η πρόσφορη συνθήκη της δράσης θα πρέπει πρώτα να αναλύσουμε καλά τα προβλήματα. Και νομίζω ότι μια πολιτική συνοχή και ένα κοινό όρομα θα βοηθήσει την j Σε ό,τι αφορά την πιστιστική ασφάλεια, είμαι αρκετά αισιόδοξο. Εγώ δεν συμμετέχω στις διαπραγματεύσεις. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, που είναι ο πρόεδρος του G20, μου ανέθεσε συγκεκριμένη αποστολή, αλλά οι διαπραγματεύσεις στο G20 ε, δεν θα... είναι κάτι που, στο, στο οποίο δεν συμμετέχω. Ελπίζω ότι με το έργο που επιτελέσαμε και που είναι πολύ σημαντικό θα καταφέρουμε να τα λήξουμε σε κοινή θέση. Κάτι που είναι δύσκολο γιατί είναι διαφορετικέ ιδεολογίε, ε, οι σκέψει. Το να καταλήξουμε σε κοινέ διακηρύξει που έχουν περιεχόμενο και αυτό από μόνο το αποτελεί μια επιτυχία. Και τέλος κυρία Τόγια, θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με την ιδέα ότι δεν θα πρέπει ο κίνδυνος να αποτελέσει το μοναδικό στοιχείο της ανάλυσης ή ο σκοπός της ανάλυσης. Θα πρέπει να αντιληφθούμε και την ευάλωτη θέση των αναπτυσσομένων χωρών και των παραγωγών και καλλιεργητών αυτών των χωρών. Στο παρελθόν είχαμε χρεώσει χώρες χωρίς να λάβουμε υπόψη την ευπάθειά τους, τον ευάλωτο χαρακτήρα τους. Και αυτός ίσως είναι ένας λόγος τη κρίσης τους χρέου, γιατί υπερχρεώθηκαν χώρες που ήταν ήδη ευάλωτε. Δεν μπορούμε να κατηγορούμε πάντα την κακή διακυβέρνηση. Σίγουρα είχε το ρόλο της το πρόβλημα, αλλά ε, ο ευάλωτος χαρακτήρας των αναπτυσσόμενων χωρών είναι το βασικό πρόβλημα. Και νομίζω ότι από αυτή την άποψη πρέπει να κάνουμε μια ανάλυση των κινδύνων και να βοηθήσουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες να τις διαχειριστούν. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Χέρμαν για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ, θα ήθελα να απαντήσω σύντομα στην κυρία, στις κυρίες Τσίμερ και Τόια. Καταρχάς βεβαίως η Oxfam υποστηρίζει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση όπως τονίστηκε και από τους τρεις βασικούς ομιλητές της πρωινής συνεδρίασης. Αυτή η ολοκληρωμένη προσέγγιση σαφώς καλύπτει και το ζήτημα της κερδοσκοπίας. Όσον αφορά την πολιτική βούληση και τα, μέσα, τα μέτρα που έχουμε στο τραπέζι μας, δίνω ιδιαίτερη σημασία στη διαφάνεια. Μέχρι εχθές πιστεύαμε ότι ε, τα, τα ζητήματα αυτά θα προχωρήσουν γρήγορα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδαμε όμως μια αντιπροσωπεία να αντιτίθεται και να καταψηφίσει την ε, υπερψήφιση της ε, Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τη ρύθμιση των αγορών τροφίμων εμείς πιστεύουμε ότι αυτή η οδηγία θα ήταν ένα θαυμάσιο μέσον ε, για την επίλυση πολλών ε, προβλημάτων και στρεβλώσεων των αγορών τροφίμων. Ε, το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που έχουμε μια καλύτερη εικόνα των ε, αγορών, ε, η κατάσταση επιδεινώνεται περισσότερο. Βλέπουμε ότι είναι περισσότερο αρνητική. Η Κομισιόν αναθεωρεί την προσέγγιση της, την έχει αναθεωρήσει πολλές φορές ήδη. Πιστεύω ότι η Επιτροπή η Επιτροπή Ανάπτυξης μπορεί να δώσει πολύτιμες σύμβουλες ε, προς την Κομισιόν ε, αλλά και ειδικά στο θέμα της ε, επισητιστικής ασφάλειας ε, στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Αυτό που πρέπει να περιληφθεί στις προτάσεις της Κομισιόν και που βάσει πρόσφατων πληροφοριών δεν είμαι βέβαιος ότι θα καλυφθεί ενώ ο Επίτροπος Μπαρνιέ είπε ότι θα περιλάβει ρυθμιστικά μέτρα σε αυτή την αγορά. Αυτό το οποίο θέλαμε εμείς είναι να υπάρχει ένα όριο στις ε, θέσεις ε, των χρηματοοικονομικών ε, συναλλαγών. Αυτό όμως που προτείνει τώρα είναι μία θέση η οποία θα γίνεται διαχειριστική θέση, δηλαδή διαχειριζόμενη θέση. Εγώ δεν νομίζω ότι αυτή η προσέγγιση στις ε, χρηματιστηριακές συναλλαγές είναι επαρκής. Πρέπει να υπάρχει στις εμπορικές πλατφόρμες ένα σαφές όριο ε, κερδοσκοπίας ή επιτρεπόμενων ε, θέσεων και όχι μία επιτρεπόμενη διαχείριση των ορίων αυτών. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να αλλάξει η πρόταση αυτή, ιδίως στο θέμα των ε, βασικών αγαθών τροφίμων. Διότι τα αγαθά, τα διατροφικά αγαθά δεν είναι όπως άλλα άλλα αγαθά, έχουν μία άμεση επίπτωση στον επισητισμό ε, των πληθυσμών. Ε, δεν μας φτάνουν τα άλλα προβλήματα που έχουμε του πληθωρισμού, ε, της αστάθειας και της αδιαφάνειας Πιστεύω ότι οι κυβερνήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα του, των τροφίμων και του επισητισμού ως πρόβλημα που άπτεται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γι' αυτό ακριβώς εμένω στο ότι θα πρέπει να τεθούν όρια στις αλόγιστες διακυμάνσεις και μεταβολές στις τιμές των τροφίμων. Τα τρόφιμα λοιπόν πρέπει να διαχωριστούν από τα άλλα προϊόντα των χρηματαγορών. Πρέπει επίσης να ελέγξουμε τις ε, εμπορικές συναλλαγές υψηλής συχνότητας Βλέπουμε σε, στις ε, προτάσεις πάρα πολλές εξαιρέσεις στους κανόνες, δηλαδή διάφορα παραθυράκια να ανοίγονται όσον αφορά τη διαφάνεια, την τήρηση ορισμένων κανόνων κλπ. κλπ. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι οι εξαιρέσεις από τις βασικές ρυθμίσεις είναι δικαιολογημένες. Πιστεύουμε ότι είναι αποτέλεσμα πιέσεων των διαφόρων λόμπι, των διαφόρων ομάδων συμφερόντων. Παρ' ε, παραδείγματος χάρη, όσοι εμπορεύονται τα σιτηρά δεν θα πρέπει να καλύπτονται από εξαιρέσει για τις ε, χρηματοοικονομικές ε, θηγατρικές εταιρείες, για τα χρηματοπιστωτικά θηγατρικά ιδρύματα. Αυτά. Ευχαριστώ. Λέει η Πρόεδρος. Για αυτήν την συζήτηση με, την δέυτερο με, το δεύτερο, με τη δεύτερη στρογγυλή τράπεζα και περνάμε στην τρίτη για τις επενδύσεις και την αρπαγή γεών. Περνάμε λοιπόν στο θέμα των μαζικών επενδύσεων στις γεωργικές αγορές των αναπτυσσόμενων χωρών. Σύμφωνα με κάποιους αναλυτές, οι επενδύσεις αυτές μπορεί να είναι υποφελείς ε, όχι μόνο για τους επενδυτές θα έπρεπε να είναι και για τους τοπικούς πληθυσμούς. Η πραγματικότητα όμως μας διαψεύδει. Δεν είναι εύκολο να δημιουργηθούν καταστάσεις win-win. Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις και οι σύλλογοι ε, δείχνουν ότι υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις ε, και στην επιστημιστική ασφάλεια, στην διαχείριση των γεών, την κατάσταση των δικαιωμάτων το τι συμβαίνει με τους τοπικούς πληθυσμούς και τις τοπικές κοινωνίες. Έτσι ολόκληροι πληθυσμοί αποστερούνται από το δικαίωμα πρόσβασης της γης ε, που τους ανήκει από γενιές επειδή δεν υπάρχουν δικαιώματα κατοχής της γης ή δικαιώματα ε, γεωκτημοσύνης στις αναπτυσσόμενες χώρες. Θα ήθελα λοιπόν να μιλήσουμε με τον κύριο Ντισάλ για το Μαλάουι, για τη Σενεγάλη και για το τι συμβαίνει αλλού. Επειδή μας ανασχολούν αυτές οι αρνητικές ε, καταστάσεις, πολλά ε, διεθνή θεσμικά όργανα και περιφερειακά θεσμικά όργανα ξεκίνησαν πρωτοβουλίες για να αντιμετωπίσουν την απόκτηση γεών ε, μεγάλης κλίμακας. Σήμερα αποφασίσαμε να συζητήσουμε τις συνθήκες και του κανόνε που θα πρέπει να θεσπιστούν, ώστε οι ξένες να είναι συνεπείς με το ανθρώπινο δικαίωμα της διατροφή, την βιώσιμη ανάπτυξη και το σεβασμό του δικαιώματος αυτοδιάθεσης. Θα ήθελα λοιπόν να καλωσορίσω τους τρεις εμπειρογνώμονές μας. Την εξοχότητά του, την κυρία Μπραβ Ντιστάλ, που είναι πρέσβυρα του Μαλάουι στις Βρυξέλλες, η οποία έχει εργαστεί και στην Επιτροπή της Αφρικανικής Ένωσης για τα θέματα της Γεωργίας, καθώς και στην ΦΑΟ και το ΕΦΠΡΙ το Λορέντσο Κοτούλα, που είναι ερευνητής, senior ερευνητής στο Διεθνές ε, Ίδρυμα Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης του Ηνωμένου Βασιλείου. Έχει διεξαγάγει μια μεγάλη συμβέλεια μελέτη για την ανάπτυξη μεγάλη κλίμακα για τη ΦΑΟ και τη ΦΙΝΤΑ. Και τον Άγκου Σέλμπι, που είναι διευθυντή τη Altima Partners, μια επενδυτική εταιρεία που βασίζεται στο Λονδίνο και η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των γεωργικών γεών. Η διεθνή χρηματοπιστωτική κοινωνία ασχολήθηκε πρόσφατα, ανέθεσε μάλλον, άρχισε να συνεργάζεται πρόσφατα με την Altima Partners, επενδύοντα σε ένα ταμείο που θα στηρίξει του χωρικού και του γεωργού για την επισητιστική παραγωγή και τι αναδυόμενε αγορέ. Τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Ντισάλ για 10 λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Ζολή. Οι επενδύσεις σε ξένες yes, είναι ένα πολύ συζητημένο, πολύ συζητημένο και καυτό θέμα. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω. Η Αφρική είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο της επένδυσης, ε, των ξένων επενδύσεων σε αφρικανικές εκτάσεις ε, δεδομένου ότι η Αφρική αντιμετωπίζει προβλήματα επισητισμού των πληθυσμών της. Έχοντας με προσοχή παρακολουθήσει τις συζητήσεις σήμερα, θα ήθελα να σας παραθέσω τι είπε ο πρόεδρος του Μαλάουι το 2015 κανένα παιδί στην Αφρική δεν θα πρέπει να πεθάνει από πείνα, υποσυτισμό ή να υποφέρει από πείνα, να είναι πεινασμένο. Αυτό είπε ο πρόεδρο, πρόεδρος μας ε, στην ε, συνεδρίαση αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των Αφρικανικών χωρών. Έδειξε λοιπόν ο πρόεδρος ε, του Μαλάβη ότι το θέμα του επιστημισμού της Αφρικανικής Υπήρου είναι θέμα προτεραιότητα στην ατζέντα. Συμφώνησαν τότε αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων η Αφρική να, να γίνει εξαγωγική ήπειρος ε, στα τρόφιμα, ε, να βοηθήσει τον επιστημισμό άλλων υπήρων και, για να γίνει αυτό θα πρέπει το 10% των πλούτων παραγωγικών πηγών της Αφρικής να, να επενδυθούν στην γεωργία και στην παραγωγή τροφίμων. Αυτή τη στιγμή όμως αντιμετωπίζουμε ακριβώς αυτήν την εισρωή ξένων κεφαλαίων για την απόκτηση γεών. Γιατί έχει λοιπόν ανοίξει ξαφνικά αυτή η επενδυτική α, όρεξη ξένων επενδυτών θα, οδηγήσει, θα οδηγήσουν αυτές οι μεγάλες επενδύσεις στην εξάλληψη της πείνας, του υποσυτισμού και της λιμοκτονίας. Θα βοηθήσει στο να γίνει η Αφρική ε, το κέρας της αμασίας για τον υπόλοιπο κόσμο. Έχουμε λοιπόν αρμόδιους φορείς ε, που εξετάζουν ε, αυτά και αναλύουν αυτά τα ερωτήματα. Όμως είναι γεγονός ότι αυξάνονται η απόκτηση γεών από ξένους επενδυτές, αυξάνονται οι εκτάσεις ε, που αγοράζονται και η η IAAD και ο ΦΑΟ έχουν δείξει με τις μελέτες τους ότι 2,5 εκατομμύρια εκτάρια αυτή τη στιγμή ανήκουν σε ξένους επενδυτές σε πέντε χώρες, μόνο σε πέντε χώρες, 2,5 εκατομμύρια εκτάρια. Βλέπετε λοιπόν τον όγκο, το πόσο μεγάλο, μεγάλη έκταση έχει αυτό το φαινόμενο ε, ξένων επενδύσεων, επενδύσεων ξένων κεφαλαίων δηλαδή στην απόκτηση και αγορά γεών στην Αφρική. Δεν μιλάμε για εγχώριους επενδυτές, μιλάμε για ξένους αλλοδαπούς. Γιατί σημειώθηκε αυτό το φαινόμενο. Είναι, πιστεύω, μία πίεση και στην πλευρά της ζήτησης και στην πλευρά της αγοράς, προσφοράς, προσφορά και ζήτηση. Το πρώτο, η ζήτηση ε, άπτεται της επιζητιστικής ασφάλειας. Ε, υπάρχει ασφαλώς ένα έλλειμμα επιστημιστικής ασφάλειας διότι υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση. Ζήτηση μεγαλύτερη, η μεγαλύτερη ζήτηση οδήγησε σε αύξηση των τιμών. Οι τιμές αυξήθηκαν διότι δεν, δεν επαρκούει η προσφορά εγχώριων προϊόντων, άρα λοιπόν οι αγορές ζητούν την εισαγωγή προϊόντων από ε, τρίτες χώρες. Εν συνεχεία, το πρόβλημα των βιοκαυσίμων. Και αυτό το πρόβλημα είναι παγκόσμιο και όπως ε, μας είπαν και το πρωί, ε, πρέπει να πω ότι ορισμένες από τις εξελίξεις στις αγορές βιοκαυσίμων οφείλονται και στα στόχους που έθεσαν κυβερνήσεις. Ε, Υπάρχει και ζήτηση στα βιοκαύσιμα, αλλά έχουν δοθεί από πολιτικές πλευρές τεράτια, τεράστια επενδυτικά κίνητρα για την καλλιέργεια βιοκαυσίμων έτσι ώστε οικονομικά να συμφέρει πάρα πολύ η καλλιέργεια βιοκαυσίμων και όχι άλλων ε, προϊόντων, καλλιεργήσιμων προϊόντων. Ένα άλλο πρόβλημα βεβαίως είναι η πτυχή της κερδοσκοπίας, η οποία επικεντρώνεται στην πίεση επί των τιμών και έτσι υπάρχει πίεση στην πλευρά της προσφοράς. Η προσφορά πώς μπορεί να εξασφαλιστεί, η επαρκής προσφορά τροφίμων, με μακροχρόνιες επενδύσεις στο Μαλαουί ο αγροτικό τομέα είναι ο κατευθυντήριο τομέα, ε, ο ηγετικό τομέα της οικονομίας μας. Ε, αλλά ομιλώ για μια γεωργία, για έναν αγροτικό τομέα που βασίζεται στους μικρούς παραγωγούς και καλλιεργητές. Οι μικροκαλλιεργητές στη χώρα μου πρέπει να βοηθηθούν, πρέπει να υποστηριχθούν από πλευράς τεχνογνωσίας, παροχής κατάλληλων μέσων, τεχνολογίας κλπ. Για να μπορέσουν να ανταποκριθούν ακριβώς στην αύξηση της ζήτησης. σε ολόκληρη την Αφρική 5% ε, του πλούτου διοχετεύεται στη Γεωργία και 3% των ξένων, ε, της ξένης βοήθειας ε, διοχετεύεται στην Γεωργία. Αυτά δεν φτάνουν, πρέπει να αυξηθούν. Υπάρχουν όμως και τεράστιες, τεράστια ρίσκα. Υπάρχει κερδοσκοπία, υπάρχουν οι πιέσεις στις τιμές των τροφίμων και ποιος τελικά ζημιώνεται ο μικροπαραγωγός, ο μικροκαλλιεργητής. Οποιαδήποτε μέτρα και οποιαδήποτε βοήθεια διοχετεύεται στην Αφρική πρέπει να λάβει υπόψη τις τοπικές συνθήκες, τους τοπικούς παραγωγούς. Τι κάνει τώρα η Αφρική. Θέλω να τονίσω ότι υπάρχει ένα πλαίσιο κατευθυντήριων γραμμών που υιοθετήθηκε το 2010 από τη διάσκεψη κορυφής ε, της Ένωσης Αφρικανικών Κρατών. Αυτό που πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι και στις πέντε γωνίες της Αφρικής όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμμετάσχουν στην εφαρμογή αυτού του πλαισίου. Η εφαρμογή λοιπόν αυτού του ρυθμιστικού πλαισίου που υιοθετήθηκε από Ένωση, από την, ε, την Ένωση Αφρικανικών Κρατών είναι σωστό. Η θεμελιώδης όμως ερώτηση είναι αν αυτή η όρεξη για καλλιεργήσιμες γης μπορέσει να εξασφαλίσει την αηφόρο κάλυψη των αναγκών, των τοπικών αναγκών ε, των Αφρικανικών περιφερειών. Η, Ένωση, η Αφρικανική Ένωση, η, η Επιτροπή του ΟΗΕ για την Αφρική και άλλοι διεθνείς φορείς έχουν οργανώσει ε, ένα φόρουμ, ένα συνέδριο υψηλού επίπεδου για τη μελέτη ε, των ξένων επενδύσεων στην Αφρική θα γίνει στον, Αρόι, στον ε, και θα συμμετάσχει η κοινωνία των πολιτών, γενικές οργανώσεις, καταναλωτές, κέντρα αριστείας ε, και όλοι οι διεθνείς φορείς. Πρέπει λοιπόν αυτή, στη μεγάλη αυτή διάσκεψη, στο μεγάλο αυτό συνέδριο, να συζητηθεί αυτή η ισορροπία μεταξύ των ξένων επενδύσεων, της μαζικής εισδορής κεφαλαίων, αλλά και της προστασίας του μικροπαραγωγού. Το Ευρωπαϊκό, η Ευρωπαϊκή Ένωση με το ε, ψήφισμα της ε, στηρίζει ακριβώς αυτή την προσέγγιση. Ε, και σας επισύω την προσοχή ακριβώς στο πλαίσιο αυτό το οποίο νιοθέτησε και επικείωσε η διάσκεψη της Αφρικανικής Ένωσης και ας, ας μας οδηγεί ακριβώς αυτή η δέσμευση του Προέδρου του Μαλάουι ότι το 2015 κανένα παιδί στην Αφρική δεν θα πρέπει να υποφέρει από, λιμοκτο, από πείνα, λιμοκτονία και υποσυτισμό δηλαδή επικέντρωση στον άνθρωπο. Και τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Κοτούλα για 10 λεπτά. Merci. Κατά πρώτον, να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας που μου δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσω σε αυτή τη δημόσια ακρόαση τα στοιχεία μου και ήθελα να ξέρω το έργο σας ως τώρα, ιδίως το πολύ σημαντικό ψήφισμα που πρόσφατα εγκρίθηκε. Εργόζομαι για το Διεθνέ Ίδρυμα Περιβάλλοντο και Ανάπτυξη που έχει την έδρα του στο Ηνωμένο Βασίλειο και ήθελα να παρουσιάσω στοιχεία που αφορούν την εμβέλεια, τη γεωγραφική κατανομή και τα χαρακτηριστικά τη ε, αρπαγής Εκτιμάται ότι στη διάστημα ενός έτους από το 2008 έως 2009 6 εκατομμύρια εκτάρια αποκτήθηκαν διεθνώς, δηλαδή διάφορες 60 εκατομμύρια εκτάρια, ε, μία έκταση περίπου ίση με την ε, σημερινή έκταση της Ουκρανίας. Εδώ δεν μιλάμε για εκμισθώσεις μόνο οι αγορές γεών, αλλά οι περισσότερες αποκτήσεις έλαβαν χώρα στην Αφρική. Υπάρχουν αριθμοί και τιμές ε, τη Αφρική και των γεών που προσέλκυσαν μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον όπω την Αιθιοπία, το Σουδάν και την Μοζαμπίκη. Αλλά υπάρχουν ιδιαίτερα κοινά συμφέροντα που ενδιαφέρθηκαν για την απόκτηση γεών για αρδευτικούς σκοπούς και ούτω καθεξής, όπως στο Μαλί με μεγάλης ε, κλίμακας αποκτήσεις που ε, εντοπίζονται σε ένα τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα με την Ιγυρία, όπου υπάρχουν μεγάλα συμφέροντα αρδευτικά. Τα κίνητρα για το φαινόμενο αυτό προσφάτως έγιναν γνωστό και τα εντόπισε και η προηγούμενη ομιλήτρια. Τρόφιμα. Τα τρόφιμα των οποίων η τιμή περιμένουν οι επενδυτές να, αυξηθούν, να αυξηθεί λόγω της γεωγραφικής κατανομής, η αλλαγή των καταναλωτικών ε, τάσεων και η αστικοποίηση. Έπειτα τα βιοκάψιμα, τα οποία δημιουργούν ανάλογες ε, δημόσιες πολιτικές, όπως και συγκεκριμένες τάσεις κατανάλωσης των βιοκαυσίμων, ε, όπως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποιοι θέλουν επίσης να παράγουν χρήμα από τις πιστώσεις άντρακα, αλλά και υπάρχουν και χρηματοπιστωτικοί σκοποί. Δηλαδή κάποια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ενδιαφέρονται για τα εδάφη λόγω των εισοδημάτων που μπορούν να παραχθούν και από κεφαλογική ε, αύξηση και από αύξηση της παραγωγικότητας μέσω τεχνολογικών μέσων, διαχείρισης και αγροτικών ε, μεθόδων. Σε μέσα μαζικής ενημέρωσης χωρών όπω η Κίνα ή οι χώρες του αραβικού κόλπου. Είδαμε την προβολή έλαβε το φαινόμενο αυτό. Δεν βρίσκονται μόνο όμω οι ντόπιοι ε, στο, προς πρώτη γραμμή της απόκτησης γεών, αλλά και ξένοι επενδυτές όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εταιρείε, ανάλογα με τη διαφήμιση που γίνεται για την κάθε χώρα. Τι σημαίνει τώρα το φαινόμενο αυτό για τις δικαιούχες χώρες. Ε, υπάρχει η, η αντίληψη ότι κάποιες χώρες, κάποιες περιοχές ολόκληρες στην Αφρική είναι κενές, ανεκμετάλλευτες. Όχι, διότι οι άνθρωποι εκμεταλλεύονται τη γη τους ακόμα και όταν ε, δεν φαίνεται αυτό εμφανώς. Μπορεί να χρησιμοποιούνται για την ε, συγκομιδή ξυλίας ή για γρανάπαυση, αλλά σε κάθε περίπτωση μιλάμε για 200 εκτάρια τα οποία μπορεί να φαίνονται κενά αλλά χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς ή υπάρχουν άλλες δεσμεύσεις που κυρίως έχουν να κάνουν με τη χρήση των υδάτων. Οι άνθρωποι λοιπόν χρησιμοποιούν τη γη τους. Το θέμα όμως είναι τι δικαιώματα έχουν, τι δικαιώματα ιδιοκτησία, τα οποία μπορεί να μην καλύπτονται από τη διεθνή νομοθεσία. Οι διαφορέ είναι μεγάλε στην νομοθεσία μεταξύ των χωρών, όμω κάποιοι έχουν δικαιώματα χρήση τουλάχιστον στη γη του. Κατά πολλού τρόπου, τα δικαιώματα αυτά είναι αδύναμα λόγω των ε, εχεγγύων που προβλέπονται. Η κυβέρνηση λοιπόν θα πρέπει κατά τι διαπραγματεύσει να φροντίζει για τη διάθεση τη γη. Αλλά πολλέ φορέ υπάρχει έλλειψη διαφάνεια. Δεν είναι γνωστό το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων και πολύ λίγα πράγματα διατίθεται δημοσίω. Οι διαβουλεύσει προβλέπονται από, την, ε, τον νόμο και οι ειδικοί διακανονισμοί επίση, αλλά δεν εφαρμόζονται συχνά. Ε, Αναλύσαμε κάποιες από τις συμβάσεις που δημοσίως έγιναν γνωστές. Κάποια είναι προσφάτως ε, διαπραγματευμένα συμβόλαια. αλλά μιλάμε για συμβάσει λίγων σελίδων όπου δεν ήταν ε, σαφή τα στοιχεία, λίγα πράγματα λέγονταν, αλλά ούτε καν τα οικονομικά ωφέλη που αποκόμιζε η χώρα η οποία απολούσε τη γη Τι μας λέει λοιπόν αυτή η εικόνα, τι θα έπρεπε να συμβεί. Πρώτα απ' όλα, πολλή λόγο έγινε για την ανάγκη γεωργικών επενδύσεων. Σε πολλέ χώρε αυτό νομίζω ότι ισχύει και κανεί δεν λέει ότι αυτό θα έπρεπε να μην ε, συμβαίνει. Αλλά για τι είδου επενδύσει μιλάμε η ποιότητα των επενδύσεων είναι εξίσου σημαντικέ με την ε, ποσότητα. Την τελευταία τριετία υπάρχει τέτοια ένταση του φαινομένου αυτού που ο αντίκτυπο είναι ισχυρό για τον τοπικό πληθυσμό. Μεγάλα κομμάτια γη χάνονται για του τοπικού πληθυσμού και είναι πολύ δύσκολο να βρούμε πετυχημένα πετυχημένε περιπτώσει. Όπου και οι θέσει εργασία να έχουν διατηρηθεί και τα εισοδήματα να έχουν εξασφαλιστεί. Έτσι λοιπόν, επενδύσει χρειάζονται, αλλά χρειάζεται και ένα δομημένο σύστημα. Ε, η, εμπειρία και οι τεκμηρίε που διαθέτουμε από την ΦΑΟ και άλλου φορεί πρέπει να αξιοποιηθούν. Σημαντικό είναι ότι οι χώροι πληθυσμοί είναι αυτοί που θα πρέπει να ανελάβουν ηγετικό ρόλο εδώ, γιατί αυτού αφορά κυρίω το φαινόμενο. Πρέπει να γίνει ανοιχτή συζήτηση για το πώ προχωρά το πράγμα σήμερα και σε χώρε όπου μεγάλε περιοχέ όντω πολλούνται και αγοράζονται. Εδώ λοιπόν οι οργανώσει των γεωργών θα πρέπει να κάνουν τη φωνή του να ακουστεί σε τέτοιου είδου ε, συζητήσει. Στο Μαλί, λόγου χάρη, οργανώσει παραγωγών τον τελευταίο χρόνο υπήρξαν επιτυχημένοι σε αυτή την προσπάθεια. Θα πρέπει λοιπόν εκείνοι να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και κάποιε διεθνεί πρωτοβουλίε αναλαμβάνονται. Είναι σημαντικέ, οι ε, κατευθυντήριε γραμμέ αναπτύσσονται από την ΘΑΟ για την διακυβέρνηση τη γη και καλύπτεται και το θέμα αυτό εκεί. Επίση, υπάρχει ένα άλλο πρόγραμμα, μια διαδικασία που ονομάζεται υπεύθυνε γεωργικέ επενδύσει και όλα αυτά έχουν κάποια σημασία, διότι μπορούν να παράσχουν ε, καθοδήγηση για χώρε που θέλουν να υπάρξουν επενδύσει αυτέ, αλλά να κάνουν τα πράγματα σωστά. Και υπάρχουν προκλήσεις αυτή τη στιγμή και σε τοπικό και σε διεθνές επίπεδο. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ασχοληθούμε με το υπόλογο και την ε, διαφάνεια. Η λογοδοσία είναι ένα σημαντικό στοιχείο και οι προκλήσεις που ανέφερα προηγουμένως για τα νομικά πλαίσια. Τέλος, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι υπάρχουν οι ανάλογες δυνατότητες. Οι γεωργοί στις, τοπικές, στις περιοχές επιμέρους μπορούν να κάνουν τη φωνή τους να ακουστούν, οι οργανώσεις τους το ίδιο έχουν δικαίωμα να εκφράζονται και η κοινωνία των πολιτών μπορεί να εξετάσει τον τρόπο που προχωρά η σύμβαση και η σύναψη συμβάσεων. Όλα αυτά είναι σημαντικά για τις χώρες ολόκληρες. Τέλος, στα συμπεράσματα, να πούμε ότι εδώ μιλάμε για έναν τομέα όπου κάποιες θεωρίες οδηγούν τα γεγονότα στην πράξη, όπως ότι υπάρχουν μεγάλες περιοχές γης ελεύθερες στην Αφρική, αυτό είναι ένα τρόπο να προχωρήσει η Γεωργία, αλλά δεν μπορούμε να βασιζόμαστε μόνο σε υποθέσει. Χρειαζόμαστε και αποδεικτικά στοιχεία για το τι πραγματικά συμβαίνει στην πράξη. Τι μηχανισμοί μπορούν να αναπτυχθούν για να διαρθρωθούν έτσι οι επενδύσει ώστε τα ωφέλη να είναι φανερά για του ντόπιου πληθυσμού. Και πρέπει αυτό να χρησιμοποιείται και για συζητήσει ε, και επίγνωση των ε, ανθρώπων που του αφορούν οι επενδύσει αυτέ για το τι συμβαίνει ακριβώ και για τι ίδιε τι χώρε. Ευχαριστούμε πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Σέλιμπι για 10 λεπτά. Uh, um, Καλημέρα σας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και την Επιτροπή σας για την ευκαιρία που μου δίνετε να αναφερθώ και στη θέση του ιδιωτικού τομέα για το πρόβλημα. Θα ήθελα καταρχήν να βάλω κάποια σύντομα σχόλια σε ό,τι αφορά την έκθεση και το ψήφισμα. σίγουρα είναι πολύ θετικό προς τους μικροκαλλιεργητές και σχεδόν εις βάρος των ε, μέγαλο καλλιεργητών και της οργανωμένης ε, εκτεταμένης ε, γεωργίας και εις βάρος της απτής αναπτυξιακής βοήθειας που χρειαζόμαστε στον τομέα αυτό και επίσης στηρίζεται και τάσεται υπέρ του κρατικού φορέα, του δημοσίου φορέα σε ό,τι αφορά τη δρομολόγηση τη βοήθεια, ει βάρο και πάλι του ιδιωτικού φορέα, του ιδιωτικού κλάδου. Παρόλο που είμαι υπέρ των μικροκαλλιεργητών του soft finance και τη προσέγγιση υπέρ του δημοσίου φορέα, δεν θα πρέπει να αμελούμε τον ιδιωτικό φορέα, την εκτεταμένη γεωργία και τα πιο απτά στοιχεία τη υποστήριξη. Και από την άποψη αυτή θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να περάσουμε κάποια μηνύματα στη συζήτηση αυτή. Το πρώτο είναι ότι θα πρέπει να μας προβληματίζει η μακροεικόνα σε ό,τι αφορά την ε, ζήτηση και την προσφορά στη γεωργία. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μια μακροπρόθεσμη ε, προοπτική, αλλά να μην ενδίδουμε στον πανικό, γιατί υπάρχουν και ρεαλιστικές προσεγγίσεις. Είμαστε υπέρ των μικροκαλλιεργητών, αλλά είμαστε υπέρ και των μεγαλοκαλλιεργητών. Είμαστε υπέρ ε, το, των απτών πρωτοβουλειών ενίσχυση αλλά και πιο ήπιων πρωτοβουλειών ενίσχυση. Νομίζω ότι είναι μια πολυεπίπεδη αντιμετώπιση με πολλά φάρμακα. Α μην πολλώνουμε τη συζήτηση. Γιατί υπάρχει πραγματικά μια αρπακτική τάση αυτή τη στιγμή, άπληστη τάση ε, και για όλα θεωρούμε υπεύθυνου στους μεγαλοκαλλιεργητές και νομίζω ότι μια τέτοια κριτική είναι αντιπαραγωγική. Όχι ότι το μικρό είναι καλό και το μεγάλο είναι κακό. Αυτή η μονολυθική πολλωμένη αντίληψη είναι αφελής, για να μην πω και επικίνδυνη. Αυτή η υπεραπλούστευση είναι αφελής ως και επικίνδυνη. Τώρα, για να σας δώσω μερικά στοιχεία για το δικό μας έργο. Εγώ εργάζομαι σε ένα ταμείο private equity που επενδύει στη τη Γεωργία τα τελευταία 6-7 χρόνια και επενδύουμε σε τέσσερις ε, υπήρους. Δεν θεωρούμε ότι υπάρχει έλλειψη φυσικών πόρων. Δεν θεωρούμε ότι η έλλειψη φυσικών πόρων δημιούργησε τα διλήμματα αυτής της κρίσης. Περισσότερο η έλλειψη δεξιοτήτων. Η Γεωργία για 4-5 δεκαετίες από την πράσινη ε, επανάσταση προχώρησε με αργούς ρυθμούς, χωρίς πολλές επενδύσεις και οι πολιτικές επιδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΕΠΑ ουσιαστικά αναχέτησε την ανάπτυξη της γεωργίας της αναφιόμενες, αναδιόμενες οικονομίες και νομίζω ότι θα πρέπει για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις αυτές να δούμε και τον ανθρώπινο παράγοντα και τον επενδυτικό παράγοντα. Θεωρούμε ότι σε κάθε περιοχή υπάρχει ένα μείγμα κεφαλαίου, εταιρικής ε, διάρθρωσης, ε, διαφορών εργαλείων ε, διαχείριση του κινδύνου, αλλά και ταυτόχρονα χρειαζόμαστε και πρακτικές δεξιότητες και όλοι όσοι ασχολούνται με τον κλάδο γνωρίζουν ότι υπάρχει τεράστια διαφορά παραγωγικότητας μεταξύ των καλύτερων παραγωγών χαμηλού κόστου παραγωγής και των πιο μέτριων επιδόσεων. Η γεωργία δεν είναι μόνο επιστήμη, είναι ταυτόχρονα και τέχνη. Η επενδυτική μας στρατηγική προσανατολίζεται στον ανθρώπινο παράγοντα πρώτα και παρά στον οικονομικό παράγοντα. Και περίπου ένα εκατομμύριο εκτάρια, ε, σε ένα εκατομμύριο εκτάρια επενδύουμε παγκοσμίω και είμαστε δεκτήτες κάτω του 20% αυτή τη έκταση. Οι περισσότερες εκτάσεις καλύπτονται από μεσοπρόθεσμα leasing συμβόλαια με τοπικές κοινότητε, με τοπικές κυβερνήσει ή με ντόπιου παραγωγούς που έχουν τέτοιες συμβάσεις μαζί μας. Και για κάθε δολάριο που εμπεδίουμε σε υγιή, 2 με 3 δολάρια επενδύουμε στον κόσμο και στο παραγωγικό ε, εργατικό δυναμικό που συμβάλλει στην ε, έσοδια κάθε, κάθε χρονιάς. Εμείς ε, έχουμε 2.500 περίπου υπαλλήλου και μάλιστα 10% αυτών των θέσεων απασχόλησης της κληρονομήσαμε τις περισσότερες τις δημιουργήσαμε εμείς και έχουμε και ένα δίκτυο περίπου χιλίων ιδιωτικών ομάδων επενδύσεων. Από άποψη λοιπόν δημιουργία θέσεων απασχόληση και σε τοπικό επίπεδο, η συμβολή μα ήταν αισθητή. Σε ό,τι αφορά τι επενδύσει στην υποσαχάρια Αφρική, εμεί ε, δεν έχουμε αγοράσει 200 ε, εκατομμύρια εκτάρια όπως ε, ακούσαμε. μόνο 5.000 εκτάρια αγοράσαμε και μάλιστα πολύ προσεκτικές ε, ήταν αυτές οι αγορές. Έχουμε μια εγκάρσια ενσωμάτωση αυτών των εκμεταλλεύσεων σε μια στρατηγική που προσανατολίζεται στην τόπια αγορά και όχι στις εξαγωγές. Και ταυτόχρονα με το project αυτό έχουμε και ένα μικρής εμβέλειας γεωργικό πρόγραμμα και διαπιστώσαμε ότι οι επενδύσει στη Γεωργία αποφέρουν όταν πραγματικά προσανατολίζονται στις τοπικές κοινότητες και όχι τόσο στη μακροπρόθεσμη προοπτική. Δεν θα ήθελα να επιμείνω στο θέμα της φύσης της ε, μακροπρόθεσμης προσέγγισης. Είναι μάλλον θέμα καμπυλών ε, ε, ζήτησης. Φυσικά θα χρειαστούμε περισσότερη παραγωγή τα επόμενα 20-30 χρόνια. Αυτό που με ενισχύει περισσότερο όμω είναι το θέμα της ανασφάλεια, τη αβεβαιότητας στην προσφορά. Διαφωνώ με κάποιον που είπε προηγουμένω ότι ε, δεν είναι πρόβλημα η παραγωγή. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε πολλές ανασφάλειες από πλευρά προσφορά, Για παράδειγμα, ανασφάλειας ό,τι αφορά την παροχή ίδρυυση ιδιαίτερα σε πυκνοκατοικημένε περιοχές, όπως είναι η Νοτιοανατολική Ασία, η Κίνα, η Ινδία για παράδειγμα. Και είναι απρόβλεπτο και το θέμα του καιρού. Βλέπουμε ότι έχουμε αυξήσει στον ακραίο, αύξηση των ακραίων μετρολογικών φαινομένων, κάτι που μπορεί να πλήξει τη δυνατότητα αντίδρασής μας. Επίσης είναι μεταβλητές οι εμπορικές ροές και μεταβαλλόμενες και οι εμπορικές πολιτικές. Υπάρχει ε, αδυναμία πρόβλεψης λοιπόν σε πολλούς παράγοντες. Ε, έχουμε τρεις βασικές εναλλακτικέ λύσεις ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των προκλήσεων. Για παράδειγμα, μπορούμε να επικεντρωθούμε στη βελτίωση το, της συγκομιδής ή στην βελτίωση των ε, τεχνικών διαχείρισης σε περιπτώσεις που υπάρχουν κενά ή να, έχουμε, να αφιερώσουμε περισσότερες εκτάσεις στην καλλιέργεια που υπάρχουν στην νότιο Αφρική, στην Λατινική Αμερική. Βέβαια αυτό είναι αρκετά δαπανηρό και περίπλοκο. Η τρίτη εναλλακτική είναι να επενδύσουμε στις νέες τεχνολογίες. Πολύ συχνά με ρωτάνε ποιες από αυτές τις τρεις εναλλακτικές λύσεις θα πρέπει να υποστηριχθεί. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει ταυτόχρονα να υποστηρίξουμε και τις να προωθήσουμε και τις τρεις λύσεις αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε όλες τις προκλήσεις. Μία σύντομη επισκόπηση των βασικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε σε ό,τι αφορά την, τη γεωργία μικρής εμβέλειας. Δεν θα είναι η γεωργία αυτή η πανάκια στις αυριανές προκλήσεις για τα τρόφιμα της ε, επιστημιστικής ασφάλειας. Κάθε α, γεωργός έχει διάφορα στοιχεία, γη, δώρα, κεφάλαιο, τα συνδυάζει και ανά κάθε περίοδο έχει συγκεκριμένη εσοδεία. Πολύ συχνά θα χρειάζεται να την αποθηκεύσει ή να την διαθέσει στην αγορά και τέλος θα πληρωθεί ε, για την εσοδεία αυτή για να καλύψει το θέμα του management της διαχείρισης που είναι σημαντικό στοιχείο οποιασδήποτε εκμετάλλευση Και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κάθε γεωργός είναι τεράστιες. Δεν μιλήσαμε εκτενώς για τις προκλήσεις σε ό,τι αφορά τα ε, δικαιώματα στη γη, ιδιαίτερα στην Νότια Αφρική. Τα δικαιώματα στην γεωκτησία είναι και οι περιορισμοί σε αυτά ήταν ε, μίσο πρόβλημα στην Αφρική τις τελευταίες δεκαετίες. Δεν υπάρχουν και υποδομές. Η Αφρικανική Γεωργία Μικρού Επιπέδου είναι πολύ πιο πίσω από την αντίστοιχη Λατινοαμερικάνικη για παράδειγμα. Οπότε υπάρχει ανάγκη να περάσουμε από ένα σύστημα ε, που ουσιαστικά εξασφαλίζει την επιβίωση σε ένα σύστημα που θα αποφέρει και έσοδα. Αυτή η μετάβαση θα είναι χρονοβόρα. Επίσης, Πολύ συχνά οι μέθοδοι είναι παροχημένε, αναχρονιστικές, στηρίζονται σε απεικιοκρατικά συστήματα. Πριν από μία σαρακονταετία, πεντηκονταετία. Και επίσης ε, δεν ε, υπάρχει μεγάλη δυνατότητα αποθήκευση, μεγάλες αποστάσεις, ακριβές μεταφορές, απομακρυσμένε αγορές, αναξιόπιστες, ε, μη προβλέψιμε και κακή χρηματοδότηση. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις, η κατάσταση είναι δύσκολη και οι προκλήσει που αντιμετωπίζει μια τέτοια γεωργική κοινότητα μικρή κλίμακος είναι τεράστιες. Δεν λέω ότι ε, είναι αμελητέ αυτές οι προκλήσεις, είναι σημαντικές, γι' αυτό και χρειαζόμαστε μια πολυεπίπεδη προσέγγιση. Γιατί ε, η Γεωργία μεγάλη ευέλεια έχει καλύψει μερικά από αυτά τα κενά Γι' αυτό θα μπορούσαμε να προβλέψουμε μια συνεργασία μεταξύ των δύο σκελών, της μικρής ευέλειας και της μεγάλης ευέλειας γεωργίας, για να, διορθούν, να διορθωθούν αυτές οι ελλείψεις. Και δίνω το λόγο στην κυρία Τσίμαρ. Ευχαριστώ και εγώ όλους τους τρεις εμπειρογνώμονες ε, για τις παρεμβάσεις τους που έσυξαν και πολλά άλλα θέματα προς συζήτηση. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα που έσυξαν το θέμα της εξαγοράς ε, γεών και της αρπαγής γεών. Αυτό μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα διότι η επιδότηση με 20% ε, των βιοκαυσίμων οδήγησε στην αγορά τεραστίων εκτάσεων ε, και πιστεύω ότι αυτό συνδέεται άμεσα με την ενεργειακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και λυπάμαι ιδιαίτερα που δεν ε, είχαμε πλειοψηφία στο σώμα να εκφράσουμε τις επιφυλάξεις μας και να παγώσουμε αυτή την ενεργειακή πολιτική σε αυτό το θέμα των βιοκαυσίμων και να τη σταματήσουμε μέχρι ότου κάνουμε μία ανασκόπηση της κατάστασης. Θα ήθελα να κάνω ορισμένε παρατηρήσεις αυτά που είπε ο τελευταίος ομιλητής. Είπε ότι βεβαίω και οι ιδιωτικέ επιχειρήσεις μπορούν και πρέπει να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και στην επίλυση της ε, επισητιστικής κρίσης, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε και το εξής. Οι περισσότεροι άνθρωποι στον κόσμο δεν υποφέρουν στα μεγάλα αστικά κέντρα, στις μεγάλες πόλεις, αλλά είναι οι πληθυσμοί εκείνοι που στις αναπτυσσόμενες χώρες προσπαθούν να επιβιώσουν ως παραγωγή. Είναι οι μικροπαραγωγοί, οι μικροκαλλιεργητές, οι μικρές μονάδες. Ιδίως στην Αφρική, το 70% των αυτοαπασχολούμενων στη γεωργία είναι ακριβώς η μικρή, η μικρή παραγωγή που ε, προσπαθούν να επιβιώσουν. Και αυτό ακριβώς, αυτοί ακριβώς στήγονται από την κρίση, διότι ενώ ήταν αυτάρκης, τώρα πια δεν μπορούν να θρέψουν τις οικογένειές τους. Ο μικρός παραγωγός στην Αφρική τουλάχιστον, έτσι όπως το είδα εγώ, ε, είναι μία ηλικιωμένη γυναίκα η οποία προσπαθεί διαχειρός ε, να ε, οργώσει, να θερήσει ένα μικρό χωραφάκι και δεν έχει καμία πιθανότητα να ενεργήσει ανταγωνιστικά σε οποιαδήποτε αγορά, είτε τοπική είτε παγκόσμια δεν έχει επίσης καμία πρόσβαση να αντιμετωπίσει το κόστος των επιδοτούμενων προϊόντων που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, εάν δείτε τώρα τα προβλήματα υποδομών, ε, τις μεταφορές ε, και πόσες λίγες πιθανότητες έχει ο μικρός παραγωγός ε, να ε, μεταφέρει τα προϊόντα του στην αγορά ε, αλλά και τις ελάχιστες δυνατότητες μεταποίησης των προϊόντων, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε την ανάπτυξη των υποδομών, να, βοηθήσουμε, να ενισχύσουμε τις μικρές παραγωγούς και να προστατεύσουμε τις υπάρχουσες αγορές. Ε, στις χώρες αυτές. Δηλαδή να προστατεύσουμε με ένα δίκτυο τις τοπικές αυτές αγορές για να μπορέσουν να επιβιώσουν ε, τις ε, μανίες τις επενδυτικής μανίες και των εξαγορών από τις μεγάλες εταιρείες, ξένες εταιρείες. το δικαίωμα της διατροφής θα πρέπει ασφαλώς ε, να μας οδηγήσει στην ε, ε, δημιουργία προγραμμάτων με τη συνεργασία δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Τα δημόσιες ιδιωτικές, ιδιωτικές εταιρείες, οι οργανισμοί πρέπει να συνεργαστούν. Αυτά τα προγράμματα αυτά πρέπει να χρηματοδοτηθούν στο μέλλον. Δεύτερον, εφόσον χρηματοδοτήσουμε αυτή την ε, ιδιωτική δημόσια συνεργασία, πρέπει να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότησή τους και να παρακολουθήσουμε την εξέλιξή τους. Βεβαίως πρέπει να ξέρουμε πού πηγαίνουν οι πιστώσεις αυτές. Δεν λέω ότι οι ιδιωτικές εταιρείε δεν ε, στοχεύουν στο κέρδος, όμως το θέμα είναι ε, ότι πρέπει να παρακολουθήσουμε για ποιο σκοπό γίνονται αυτά τα προγράμματα και πού διοχετεύονται αυτές οι επενδύσεις. Καταρχάς, δεν είμαι αντίθετη ε, στη συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικών φορέων, αλλά πρέπει να δούμε ότι οι επενδύσεις αυτές γίνονται σωστά, φτάνουν στους δικαιούχους ε, και να μην ε, απαλλάξουμε τις, τους πολιτικούς φορείς και τους, τις εθνικές κυβερνήσεις από την ευθύνη που έχουν για τη διαχείριση αυτών των προγραμμάτων. Euh, Ευχαριστούμε. Και τώρα μου δίνω το λόγο σε μένα την ίδια. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Κοτούλα, ερευνητή για αυτού του είδους της συμβάσεις, το εξής. Μας είπατε ότι πολλές από τις εταιρείε με τις οποίες συνεργάζεστε έχουν ε, συνάψει τέτοιες συμβάσεις, αλλά δεν μας είπατε ποιοι είναι. Θέλω να ξέρω τα ονόματά τους. Επίσης, θα ήθελα να ξέρω που είναι η έδρα τους. Εάν είδατε τους λογαριασμούς τους, τα λογιστικά τους και τι φόρους πληρώνουν στις χώρες όπου λειτουργούν επί παραδείγματι. Είχατε εσείς καμιά θετική εμπειρία, καμιά περίπτωση με, θετικές, με θετικά στοιχεία και για τη χώρα δικαιούχο. Αυτό ήθελα να μάθω και να, λόγω, να δώσω το λόγο στην κυρία Στίφλερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ η ίδια που ε, θα πρέπει να πω ότι ξεπλάγει κάπω με την παρέμβασή σας, διότι από το πρωί εξηγούμε ότι θέληση όλων μας είναι να επιτρέψουμε στους γεωργού, τους μικρογεωργούς μάλιστα στι αναπτυσσόμενε χώρες, να γίνουν αυτόνομοι, να τα καταφέρουν, να σεβαστούμε τον τρόπο ζωής τους και να σεβαστούμε τις γεωργικές τους μεθόδους. Ωστόσο, μας λέτε ακριβώς το αντίθετο δεν θέλουμε καθόλου να οδεύσουμε σε αυτή την άγουσα. Λέγατε προηγουμένως ότι οι μικρογεωργοί πρέπει να πάρουν μια πολύ σοβαρή απόφαση σε ό,τι αφορά τα πολύ μικρά αγροτεμάχια που κατέχουν. Έχω την εντύπωση όμως ότι δεν τους αφήνεται και καμιά, κανένα περιθώριο, διότι οι μικροί αυτοί γεωργοί τελικά καταλήγουν να γίνονται κολύγοι ε, αν ακολουθήσουμε τη συλλογιστική σας, σε λίγα χρόνια στην Αφρική ή στις άλλες αναπτυσσόμενες χώρες θα έχουμε διεύθυνση Ευρωπαίων, Αμερικανών ή Κινέζων και δεν θα έχουν πλέον καμία δυνατότητα δική τους. Οπότε τι είναι αυτό, δική σας πολιτική τοποθέτηση. Απορία εκφράζω τώρα. Η παρέμβασή σας θα έλεγα ότι με τρομάζει. Αυτό λοιπόν ήθελα να θέσω ως ερώτημα. Τι κάνετε, όπως είπε και η κυρία Τσίμερ, με τις μικρές αυτές εκμεταλλεύσεις, με τις γυναίκες που πολεμάνε για να κρατήσουν με νύχια και με δόντια τα αγροκτήματά τους. Και αν ήταν τόσο αποτελεσματικά τα συστήματά σας, εδώ το εξηγήστε μου, γιατί βλέπουμε όλο και περισσότερο εκατοντάδες παιδιά να πεθαίνουν από ασυτεία καθημερινά. Και ενηλίκους φυσικά. Ευχαριστώ. Κυρία Τόγια, ευχαριστώ, πολύ. Να ευχαριστήσω όλους τους ε, παρεμβαίνοντες που μας είπαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Νέα πρόκληση προβάλλει μπροστά μας. Ποια θα είναι η συνεισφορά του ιδιωτικού κεφαλαίου εφόσον ακολουθήσει σωστή κατεύθυνση προκειμένου να αναπτυχθούν τοπικά και αυτές οι κοινωνίες. Αυτό μας ενδιαφέρει Ιδίω σε ό,τι έχει να κάνει με επενδύσεις που επιτρέπουν και τη διατήρηση της ε, μικρής κλίμακας γεωργίας σε τοπικό επίπεδο. Και κάτι που τα τελευταία χρόνια κυρίως αναπτύσσεται, ιδίως ό,τι αφορά την παράμετρο των γεών. Είχα την ε, δυνατότητα να διοργανώσω και εγώ συναντήσεις και λαμβάνω την ευκαιρία εδώ κυρία Ζολή για να πω ότι και εμείς εδώ οι Ευρωπαίοι έχουμε τις ευθύνες μας. Οι φορείς, οι επιχειρήσεις είναι αυτοί που συμβάλλουν από την Ευρώπη στην αρπαγή των γεών. Γνωρίζουμε πολύ καλά λοιπόν και εμείς τι συμβαίνει. Το ερώτημα μου αφορά περισσότερο τη δυνατότητα την αναπτυξιακή, μάλλον τη δυνατότητα ανάπτυξης του πλαισίου αναφοράς που εδώ αναφέρθηκε. Οι διαπραγματεύσει για την απόκτηση των γεών είναι τελείως ανισότιμες. Και βεβαίως την ευθύνη την έχουν και οι εθνικές κυβερνήσεις, οι τοπικές κυβερνήσεις και οι τοπικές ε, αρχές εξουσίας. Ε, βλέπουμε λοιπόν ότι γεννάται θέληση για διαπραγματευτική ικανότητα, αλλά θα πρέπει αυτό να συμβεί πρώτα από του τοπικούς πληθυσμού. Ποιοι να το κάνουν, οι γεωργοί μόνοι του, αλλιώ του πετάνε στην άκρη. Τι θα κάνουμε, θα του μετατοπίζουμε μαζικώς ε, η τοπική γεωργή λοιπόν και για τις συμβάσεις μίλησα με ερευνητέ, με μελεπτέ του φαινομένου αυτού που έχουν συλλέξει στοιχεία και λένε ότι κάποιες συμβάσεις είναι ολιγοσέλιδες με μια μόνη υπογραφή. Θα πρέπει λοιπόν να δείξουμε όλοι μας την επευθυνότητα, όλοι. Περισσότερη ευθύνη τοπική σίγουρα, αλλά και εμείς οι Ευρωπαίοι στα θεσμικά μας όργανα να παρακολουθήσουμε πώ εξασκούμε την αρμοδιότητά μα αυτή, τι γνώσει που διαθέτουμε, τα εργαλεία που έχουμε. Διότι όπου υπάρχει θέληση πρέπει να υπάρχει και συμβασιακή δυνατότητα χρήση των συμβάσεων, χωρί όμω να χάνονται οι τοπικοί πληθυσμοί. Θα πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε την ενοποίηση αυτών των πλαισίων που διαμορφώνονται. Πρόεδρε, ολοκληρώνω άμεσα. Αναφέρθηκε το γενικότερο πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί σε επίπεδο ΟΗΕ μια άλλη διαδικασία που έχει ξεκινήσει, η διαδικασία του Ναϊρόμπι. Υπάρχουν κάποια εφαλτήρια λοιπόν. Μπορούμε ως Ευρωκοινοβούλιο να τα αξιοποιήσουμε για να μην γίνουν αυτά τα σημεία ε, αφετηρίας μονολόγια, μια συνθήκη, μια συμφωνία, σημεία τα οποία θα πρέπει να τα σέβονται όλοι και στο Μιλάνο, στην Ιταλία, στην καρδιά της Ευρώπης, θα έχουμε την επόμενη διεθνή έκθεση, μετά την έκθεση της Σαγκάης. Δεν θα πρέπει να μας απασχολήσει το μέλλον του πλανήτη. Εμείς ε, θέτουμε το ερώτημα, πιθανότητας μια πρόκληση και στις τοπικές αρχές. Τι θα πρέπει να προσφέρουμε ως στήριγμα στις τοπικές ε, αρχές λοιπόν όταν αντιμετωπίζουν το θέμα των ξένων επενδύσεων που μπορούν να είναι πολύ χρήσιμες όπως υπόθηκε αλλά και πολύ βλαβερές. Θα πρέπει να βοηθήσουμε με διαπραγματευτικές δυνατότητες και λύσεις. Το τι θα γίνει στην πολιτική πραγματικότητα είναι άλλο ζήτημα, αλλά εμείς οφείλουμε να κάνουμε κάτι. Merci. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Ναβάρο και σε άλλους που δεν είναι μέλη τη Επιτροπής. Για δύο λεπτά το πολύ, κύριε Ναβάρο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Μέσα από το σύστημα του ΟΗΕ ε, ε, εργαζόμαστε επί τη βάση συγκεκριμένων αρχών. Καταρχάς, κάθε αγροτική μονάδα λειτουργεί επιχειρησιακά, είτε είναι μικρή είτε μεγάλη. Ε, δεύτερον, ιδιωτικές επενδύσεις γίνονται στον αγροτικό τομέα και μέχρι σε ενός βαθμού προσπαθούμε να συνεργαστούμε με κυβερνήσεις και παραγωγούς για να αυξηθούν αυτές οι επενδύσεις αλλά με στόχο την ενίσχυση των μικροκαλλιεργητών και μικροπαραγωγών έτσι ώστε να ωφεληθούν. Σε ορισμένε χώρε και οι κυβερνήσει ενισχύουν τι ιδιωτικέ επενδύσει διότι πιστεύουν ότι αυτό είναι ο καλύτερο τρόπο ανάπτυξη. Το έχουμε δει αυτό και στου εκτροφεί ε, και στα προκυπευτικά ε, και στην Αλία. Το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει στην Τανζανία, στη Μοζαμβίκη Έχουμε επίσης δει ε, ε, ε, παραγωγούς να ενώνονται σε συνεταιριστικές μονάδες έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν πιο ανταγωνιστικά ιδιωτικές εταιρείες, επιχειρήσεις ιδίω στην Τανζανία και στη Μοζαβίκη αλλά και στο Βιετνάμ και στην Ινδονησία προσπαθεί η κυβέρνηση να επιβάλλει μια σωστή ισορροπία μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικών φορέων και μη κυβερνητικέ οργανώσεις όπως η Oxfam και άλλες ε, συμβάλλουν ενεργά σε αυτήν την ε, συνεργασία. Ζητούμε λοιπόν από τα μέλη του σώματος εδώ να μην θεωρήσουν αυτομάτως ότι η ε, συμβολή του ιδιωτικού τομέα στην, στον αγροτικό τομέα γενικώ συνδέεται αποκλειστικά και μόνο με αυτές τις ανήθικες και ανεξέλεγκτες αρνητικές συμπεριφορές ορισμένων ιδιωτών και ιδιωτικών εταιριών. Ε, η μία τέτοια συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικών φορέων μπορεί ασφαλώς να συμβάλλει στην επίλυση πολλών προβλημάτων της επισητιστικής ανεπάρκειας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σούβιλ. Ο κύριος Σουβίλ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εκπροσωπώ την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα είμαι λακωνικός. Αν θέλουμε να επενδύσουμε στη γεωργία θα πρέπει να έχουμε πρόσβαση στους πόρους, κυρίως στη γη και στο είδωρ. Σε ό,τι αφορά τις γεές, τα εδάφη, συζητήσαμε στην ΟΚΕ και με την κοινωνία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αναπτυσσομένων χωρών και θα μπορούσα συνοπτικά να πω ότι κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στην εξασφάλιση των εγγύων δικαιωμάτων των μικροκαλλιεργητών και ε, να προσέξουμε τα επενδυτικά αλλοδαπά σχέδια. Θα πρέπει οι τοπικέ κοινότητε και οργανώσεις παραγωγών να συμμετέχουν ευθύ εξ αρχή σε οποιοδήποτε προγράμματα και να δίνουν την έγκρισή τους ε, σε περίπτωση που αλλάξει η διοκτησία των ε, γεών. Πριν τις ομιλίες ε, είχα προβληματιστεί ω προς το εξή. Μία ε, διαφανής έγκυο πολιτική που θα αναμειγνύει ενεργά τις τοπικές ε, κοινότητες. Πιστεύετε ότι είναι δυνατή και μετά τις ομιλίε που άκουσα θα ήθελα να ρωτήσω και το εξή. Πιστεύετε ότι υπάρχουν κάποιες θετικέ πρωτοβουλίε και πώς θα μπορούσαμε να τις επεκτείνουμε σε όσο το δυνατό περισσότερες χώρες και εξασφαλίζοντας παράλληλα, επαναλαμβάνω, ενεργό συμμετοχή των ντόπιων κοινοτήτων και των ντόπιων παραγωγών. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Σίσοκο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα, μετά από αυτά που είπε ο κύριος Ζακέ, να του πω ότι ε, επένδυση προϋποθέτει κινδύνους. Σήμερα ποιος επενδύει, ποιος επενδύει στη γεωργία στην Αφρική ή χωρικοί και οι μικροκαλλιεργητές. Αυτοί είναι που επενδύουν το 85% των, ε, του συνόλου των επενδύσεων. Εμείς ε, επενδύουμε φυσικά αναλαμβάνοντα τους κινδύνους, γιατί επένδυση σημαίνει κίνδυνος. Ενώ οι, ε, οι επενδύσεις ενδιαφέρονται για μία δεκαετία που δεν θα πληρώνουν φόρους και που θα παράγουν προσανατολισόμενοι προς τις εξαγωγές. Αν λοιπόν θα μπορούσαμε να δώσουμε μια δεκαετία αφορολόγητη ε, σε, στους αλλοδαπούς επενδυτές και ταυτόχρονα δεν κάνουμε τίποτα για αυτούς που καθημερινά επενδύουν, αυτό δεν είναι αδικία. Εκεί έγκυται το μείζον πρόβλημα. Επίσης, είπατε ότι θα πρέπει να εξετάσουμε τη συμπεριφορά και να διορθώσουμε τη συμπεριφορά των κερδοσκόπων και αναγνωρίσετε και στους ίδιους κύριε Ζακέ ότι πώς είναι δυνατόν να διαχωρίσουμε τη συμπεριφορά των κερδοσκόπων από το ίδιο το φαινόμενο της κερδοσκοπίας. Επίσης, ε, κύριε Ζακέ, ποιες είναι οι ευθύνε ε, των κρατών πέραν της ε, νομοθεσίας. Πώς είναι δυνατόν κάποιες κυβερνήσεις που έχουν που 70% του πληθυσμού τους και 100% είναι αγροτικός πληθυσμός μπόρεσαν να παραγάγουν βαμβάκι μέχρι, ακόμη και επηρεάζοντας την παγκόσμια παραγωγή βάμβακος. Οι μικροί καλλιεργητές, σαν κακάο, καφέ, σήμερα τα ελέγξαμε όλα αυτά και αντέξαμε το διεθνή ανταγωνισμό. Πώς λοιπόν δεν μπορούμε να κάνουμε και το τα υπόλοιπα. Το πρόβλημα δεν είναι να προσελκύσουμε ε, επενδυτές που θα ιδιοποιηθούν τις γιές μας. Ε, Απλώς χρειαζόμαστε πολιτικές, πραγματικές πολιτικές που θα οργανώνουν την αγορά, που θα την προστατεύουν, που θα τη διαφυλάσσουν από την καταχρηστική εισαγωγή προϊόντων. Τα προβλήματα, όσο δεν είναι σαφή, θα εφευρίσκουμε άσχετες ε, λύσεις. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα παραγωγής για τους μικροκαλλιεργητές. Γιατί είπε ο τελευταίο ομιλητή ότι οι μικροκαλλιεργητές έχουν προβλήματα. Μα τέτοια προβλήματα έχουν οι χωρικοί παντού στον κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε τη λύση με την κοινή αγορά. Οι Ηνωμένε Πολιτείε με το Farm Bill. Δεν ήταν οι προσκεκλημένοι αλλοδαποί επενδυτέ που έλυσαν τα προβλήματα. Τα προβλήματα τα έλυσαν εσωτερικά οι κυβερνήσει, προστατεύοντα του γεωργού, διαμορφώνοντα προποθέσει για να αναγνωριστεί το έργο των γεωργών και να εξασφαλιστεί το εισόδημά του. Πριν ε, διορθωθεί αυτή η κατάσταση, κανένα επενδυτή δεν ενδιαφερόταν στην ε, Ευρώπη. Από αυτή την άποψη είναι αξιέπαινο το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αξιομίμητο. Κύριε Πρόεδρε, το πρώτο έργο που θα πρέπει να επιτελέσουμε διεθνώς είναι να σεβαστούμε το δικαίωμα κυριότητας των, των τόπιων κοινοτήτων στα εδάφη τους, στα χωράφια τους. Αυτό είναι το μείζον ζήτημα. Είπαμε εμπλοκή των όποιων κοινοτήτων κτλ. Αν δεν κατοχυρώσουμε τα δικαιώματα ε, έγκυας ιδιοκτησίας δεν πρόκειται να βοηθήσουμε τις ε, τοπικές κοινότητες. Ε, προσελκύσουμε τους επενδυτές που θα αγοράζουν και να παράγουν λουλούδια και να τα στέλνουν στο δυτικό κόσμο. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να καλλιεργούμε και να παράγουμε τρόφιμα. Ευχαριστώ για δύο λεπτά. Ο επόμενος ομιλητής. Θα μιλήσω. Θα μιλήσω. Πιστεύω ότι αυτό που γίνεται με την αρπαγή γεών είναι ότι ε, ε καλύπτουμε, ε, μιμούμεθα ένα, ένα σύστημα το οποίο ήδη γνωρίζουμε. Αναπαράγουμε δηλαδή ένα γνωστό σύστημα. Ε, μία έκθεση η οποία έγινε για τη διεθνή επισκόπηση της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται στον αγροτικό τομέα λέει ότι δεν έχει λυθεί κανένα πρόβλημα κλειδί της γεωργίας διότι η γεωργία αποτελεί μία συντονισμένη πολιτική μεταξύ των πολιτών του περιβάλλοντος και της ε, ε, γης πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις γνώσεις που έχουμε να οργανώσουμε τα πράγματα διαφορετικά και αυτό που δεν άκουσα εδώ ακόμα είναι που είναι παραδείγματο χάρη ε, ε, ποια, ποιοι καινούργιοι φορείς, ποια καινούργια ιδρύματα ενισχύουν την αηφόρο γεωργική ανάπτυξη με το καινούργιο μοντέλο ε, που εκπαιδεύονται οι γεωργοί ποια είναι η υποδομή η τεχνολογικής εκπαίδευσης των παραγωγών, των γεωργών. Έχουμε δημιουργήσει οργανισμούς και ιδρύματα τα οποία διδάσκουν στους παραγωγούς πώς να χειριστούν ε, την παραγωγή τους, τα καινούργια μηχανήματα, την καινούργια τεχνολογία. Δεν άκουσα λοιπόν τίποτα όσον αφορά την ε, τεχνολογία και την εκπαίδευση και κατάρτιση. Merci. Για μια σύντομη απάντηση θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Χέρμαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε πολύ σύντομα για το κύριο Ναμπάρο αναφέρθηκε στην Oxfam. Πράγματι προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε και τον ιδιωτικό τομέα για να δούμε ποια μπορεί να είναι η δική τους η συνεισφορά ώστε να βοηθήσουν τους μικρούς γεωργούς να αυξηθεί να εμπλακούν μάλλον στην λυσίδα παραγωγή. Την όξο των την απασχολεί μικρή κλίμακα Γεωργία. Αλλά εδώ και δέκα μέρε έχουμε και μια πρόσφατη έκθεση για το νέο κύμα μεγάλων αγορών γεών. Η έκθεση αυτή διατίθεται στα αγγλικά, ισπανικά, γαλλικά και καταγράφει τα πιο πρόσφατα στοιχεία. Όπως είπατε λοιπόν, ναι, πρέπει να προσεγγίσουμε και τον ιδιωτικό τομέα για να αναζητήσουμε σχέσεις συνεργασίας, αλλά θα πρέπει να αναγνωρίσουμε και την σκοτεινή πραγματικότητα, την οποία αντιμετωπίζουμε με το φαινόμενο της αρπαγής γεών. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει μια πτυχή που συχνά αποσκεπάται, αλλά είναι πολύ σημαντική σε όλες αυτές τις διαπραγματεύσεις. είναι η ανεπάρκεια και η αδυναμία των θεσμικών οργάνων που δεν επιτρέπει να υπάρχει ισοτιμία στις ε, διαπραγματεύσει. Υπάρχει και μια κυρία από το κοινό που θέλει το λόγο, κυρία απέναντί μου με τα μπέζ. Για ένα λεπτό. Από την, από τη Διεθνή Οργάνωση Oxfam. ακούσαμε την έντονη ε, ε, δέσμευση του εκπροσώπου της ε, του κυρίου Σπίφερ, του προσώπου του Σάλτιμα Partner, ότι κανένας ε, γεωργός δεν εκτοπίστηκε, δεν έχασε τη γη του λόγω των επενδύσεων που έκανε. Όμως ε, οι εκθέσει της Oxfam δείχνουν μια διαφορετική ε, εικόνα. 20.000 άνθρωποι εκτοπίστηκαν μικροπαραγωγή δηλαδή από λόγω της απόκτηση γεών στην Ουγγάντα από ξένου επενδυτές. Έχουμε λοιπόν μια διαφορετική εικόνα εμεί στην Oxfam. Το θέμα, όπως είπε είπε ο κύριος Σέλμπι είναι ότι δεν υπάρχουν καθαροί τίτλοι ιδιοκτησία σε μικροεκτάσεις. Ε, θέλω λοιπόν να ρωτήσω ε, ποια είναι τα πρότυπα, ποιους κανόνες ακολουθεί η Altima Partners για να εξασφαλίσει ότι δεν χάνουν τα, τις μικρο, τα, μικροεδάφη, τους και τα χωράφια τους η τοπική παραγωγή, η μικροπαραγωγή τι, μέσα χρησιμοποιεί. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ζακέ. Ευχαριστώ. Θα συμφωνήσω με αυτό που είπε προηγουμένως ο κύριος Νάμπαρο. Γιατί η Γεωργία είναι σημαντικός ιδιωτικό τομέα στι αναπτυσσόμενες χώρε. Οπότε, όταν μιλάμε για κρατικέ πολιτικέ, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε απόψη και τι εταιρικέ σχέσει με τον ιδιωτικό τομέα. Βεβαίω για τι μεγάλε επιχειρήσει και το δίκαιο του ανταγωνισμού είναι τα θέματα κάπω διαφορετικά. Όμω για να υπάρχουν σωστέ, σωστά σχεδιασμένε κρατικέ πολιτικέ και να αξιοποιείται η ιδιωτική πρωτοβουλία, πρέπει να υπάρχουν εταιρικέ σχέσει μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Είναι καθοριστική σημασία σε αυτό όχι μόνο για το ιδιωτικό τομέα, αλλά αφορά την εξέλιξη των δημόσιων πολιτικών σε κάθε τομέα και μέσα στη δική μα τη χώρα. Και η σχέση μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα πρέπει να επινοηθεί και να σχεδιαστεί εκ νέου. Να αποφύγουμε τις εντάσεις και τις ε, παρεκτροπές. Πολλές από τις ανεπάρκειες που εντοπίσαμε μέσα από τις συζητήσεις μας σήμερα έχουν να κάνουν σε σχέση με τα κράτη έναντι των πληθυσμών τους πριν γίνουν παρεκτροπές του ιδιωτικού τομέα αυτού καθεαυτού. Ευχαριστούμε. Και τώρα ο λόγος της εμπειρογνώμονές μας ο κύριος Σέλμπι που θα πρέπει να προασπιστεί τις θέσεις του σε σχέση με πάρα πολλές ερωτήσεις που του τέθηκαν. Thank you. Ευχαριστώ. Το πρώτο που, η πρώτη μου απάντηση αναφέρεται σε κάτι που είπα στην αρχή της πρώτης μου παρέμβασης ότι η συζήτηση εδώ έχει τόσο πολλωθεί ώστε να καταλήγει πάντοτε ή στο απλοϊκό ε, παράδειγμα μικρή παραγωγή καλή, μεγάλη παραγωγή κακή ή το μικρό, μικρή κλίμακα καλή και σωστή μεγάλη κλίμακα κακή ε, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτό που πρέπει πιστεύω ε, να κάνουμε είναι μια συντονισμένη υποστήριξη όλων των πλευρών. Βεβαίως ε, ε, η γεωργία μικρής κλίμακας χρειάζεται περισσότερη ενίσχυση και στήριξη από τη η γεωργία μεγάλης κλίμακας αλλά όχι ότι οι μεγάλες κλίμακες είναι πάντοτε κακές και αρνητικές. Συμφωνώ ότι η πλειοψηφία των περιθωριοποιημένων οικογενειών στην Αφρική είναι σε αγροτικές περιοχές, είναι στην Ήπεθρο Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι στην επόμενη δεκαετία η πλειοψηφία των ε, πεινασμένων οικογενειών θα βρίσκεται στα μεγάλα αστικά κέντρα, στις τεράστιες πόλεις. Άρα λοιπόν υπάρχουν δύο όψεις ε, του νομίσματος. Συμφωνώ απαντώντας στη δεύτερη ερώτηση ε, που αφορούσε τη ρύθμιση του ιδιωτικού τομέα. Συμφωνώ, αυτό είναι προφανές. Το μήνυμα μου εδώ είναι περισσότερο ότι εμείς τα τελευταία 30-40 χρόνια έχουμε δει δισεκατομμύρια ευρώ να διοχετεύονται σε δημόσιους οργανισμούς και φορείς με πολύ λίγη επιτυχία και με πολύ ε, και με ένα πάρα πολύ μειονεκτικό και λοιπές πλαίσιο αναφοράς. Ε, και πάρα πολλά κονδύλια χάθηκαν χωρίς να βρεθούν οι υπόλογοι. Ε, επίσης, ε, δεν λέω ότι πρέπει να αγνοήσουμε τον, ή να αμελήσουμε τον μικροπαραγωγό, απλώς λέω ότι η οργάνωσή μου, η εταιρεία μου έχει ασχοληθεί για τρεις γενιές στην ε, παραγωγή τροφίμων ε, στην Αφρική από μικρούς παραγωγούς. Ε, απλώς αυτό το οποίο έδειξα είναι τους τεράστιους κινδύνους, το ρίσκο το οποίο οφείλεται στον καιρό, στις καιρικές συνθήκες, στην ξηρασία, ε, και επαναλαμβάνω εν κατακλείδη ότι χρειαζόμαστε και την μεγάλη και τη μικρή κλίμακα. Ο... Η μεγάλη γεωργία, στην πούμε έτσι, μπορεί να προσφέρει οικονομία σε κλίμακος και τη δυνατότητα συνέργειας με την μικρή γεωργία, σε παρένθεση, μικρή, τους μικροκαλλιεργητές. Όσον αφορά το σχόλιο του εκπροσώπου του ΟΗΕ Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια, ένας σαφής διαχωρισμός μεταξύ των υπεύθυνων επενδυτών και των γεωκερδοσκόπων. Ε, πραγματικά υπάρχουν, ε, ε έγιναν επενδύσεις και εξαγορές ε, εκατοντάδων χιλιάδων στρεμάτων γης χωρίς να γίνουν οι επενδύσεις και χωρίς να ωφεληθεί κανείς. Ε, μου ζήτησα να καταλήξω και η τελευταία ερώτηση από την κυρία της Oxfam. Πιστεύω ότι υπάρχουν πραγματικά σκιώδεις ενέργειες και πράξεις που γίνονται αδιαφανείς, αλλά υπάρχει και πάρα πολύ καλή δουλειά που έχει γίνει. Εμείς στην Άλτιμα είμαστε πρωτοπόροι στην εφαρμογή των αρχών για τις υπεύθυνε επενδύσεις. Συνεργαζόμαστε με την Παγκόσμια Τράπεζα, το ΦΑΟ, τις, ε, τα ψηφίσματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει και ένα, ένα συναισθηματικό φόρ, ένα μια συναισθηματική φόρτιση όταν συζητιούνται αυτά τα θέματα, διότι άπτονται βεβαίως τη διατροφή και των ανθρωπίνων αναγκών. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Κοτούλα για τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να μιλήσω για αυτό το θέμα της πόλωσης της συζήτησης. Εδώ χρειαζόμαστε επικοδομητική συζήτηση, όχι πόλωμένη συζήτηση. Ή, όντως υπήρξε μια πόλωση, αλλά αυτό ισχύει αμφίδρομα. Για παράδειγμα, αν δούμε τη γνώμη ε, των ε, χωρών δικαιούχων, διαπιστώνουμε ότι αυτέ ζητούν περισσότερο εκτεταμένη γεωργία, μεγάλη εμβέλειας. Και υπάρχει δυσπιστία σε ό,τι αφορά την ικανότητα των μικροκαλλιεργητών να διαδραματίσουν το ρόλο τους. Οπότε θα πρέπει να δούμε το θέμα σφαιρικά. Έχουμε αποδείξεις ότι και οι μικροκαλλιεργητές μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί και δυναμικοί. Έχω ένα συνεταιρισμό στην Κάνα, για παράδειγμα, 6.000 κοκοκαλλιεργητών και έχουν 45% μιας βρετανικής ε, ε, εταιρείε παρασκευή ε, σοκολάτα. Βλέπετε ότι όταν δραστηριοποιούνται οι μικροκαλλιεργητέ μπορεί να είναι πολύ δυναμικοί και δραστήριοι. Σίγουρα έχουμε πολλέ προκλήσει να αντιμετωπίσουμε. Είχαμε βέβαια για πολλά χρόνια ακιδεία σε ό,τι αφορά την κατάσταση γεωργίας στις αφρικανικές χώρες. Πολλές αναπτυξιακές οργανώσεις προσπαθούν να διορθώσουν την κατάσταση και επίσης ε, υπάρχει μια διχοτόμηση μεταξύ ε, μικροκαλλιεργητών και ιδιωτικού κλάδου. Δεν ε, είναι πάντα δεδομένη μια τέτοια αντιδικία. Πολλές φορές έχουμε συνεργασία μεταξύ ε, ιδιωτικών επενδυτών και μικροκαλλιεργητών και συμμετοχή μικροκαλλιεργητών σε τέτοιες επενδυτικές εταιρείες θα πρέπει να διδαχθούμε από τέτοιες βέλτιστες πρακτικές και να τις διευρύνουμε. Και φυσικά να εξασφαλίσουμε τα έγκαια ε, δικαιώματα και να μην είναι δυνατή η αγορά έγκαιας ιδιοκτησία ε, με ανεπίσημα έγγραφα και ουσιαστικά με μηδενικό τίμημα. Η εξασφάλιση των εγκαίων δικαιωμάτων είναι σημαντικό στοιχείο για την ε, προσέλκυση και υγιών επενδύσεων. Σε ό,τι αφορά τι ευρωπαϊκές εταιρείε, είναι πολλές ευρωπαϊκές εταιρείε, ε, πολλέ καθιερωμένες, ε, με μακροχρόνιες επιδόσεις ό,τι αφορά την τροπική γεωργία. μερικέ είναι καινούργιες, ε, startups επιχειρήσεις και πολλέ συμφωνίες. Τα ονόματα δεν είναι μυστικά, τα ονόματα των εταιριών, μερικέ είναι και κρατικές ή δημόσια τα αρχεία. Δεν θέλουμε να κατονομάσουμε κανέναν και να εκθέσουμε κανέναν και μερικές ε, συμφωνίες είναι πολύ φρέσκες. Θα δούμε πώς θα εφαρμοστούν και τι ε, θέσεις απασχόλησης θα δημιουργήσουν και τι εισοδήματα θα αποφέρουν. Στη Μοζαβίκη, στην Ταζανία είχαμε ε, μια τέτοια συμφωνία που δυστυχώ δεν μπόρεσε να απογειωθεί γιατί ήταν υπερβολικά φιλόδοξη, δεν πληρώθηκαν τα κονδύλια. Θα πρέπει να δούμε κάθε συμφωνία πώς θα εφαρμοστεί. δυστυχώ διακόπτει η πρόεδρος. Θα δώσω τώρα το λόγο για τρία λεπτά στην πρέσβυρα του Μαλάου, την κυρία Τάλερ. Τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα το συγκεκριμένο παράδειγμα του Μαλάου. Το Μαλάουι χωρίζεται σε ε, ενώσεις ε, γεωργικών παραγωγών και μικρά αγροτεμάχια. Όμως τη διαχείριση την έχουν αναλάβει μικρομεσαίοι γεωργοί. Γι' αυτό η κυβέρνηση βασιζόμενη σε χώρες πολιτικέ, δίνει κίνητρα ώστε να βοηθηθούν οι μικρότεροι γεωργοί. Έχει και στοχευμένα μέτρα για 1,6 εκατομμύρια που θα διατεθούν στου μικρότερου γεωργού. για να αντιμετωπίσουμε ζητήματα υψηλή ασφάλεια, διάρκεια των ε, καλλιεργιών και πλεονάσματο για εξαγωγέ. Ένα παράδειγμα είναι αυτό, αλλά το Μαλάουι χρησιμοποίησε τη συμβολή και του ιδιωτικού τομέα, διότι και οι μικρότεροι γεωργοί μπορούν να κάνουν εμπόριο με τον ειδικό τομέα και τους μοιράζουμε και κουπόνια. Ήταν σημαντικό να σας δώσω αυτό το παράδειγμα. Έπειτα, ναι, προφανώς υπάρχουν σοβαρές προκλήσεις για τους μικρότερους γεωργούς, διότι έχουμε τα παραδεδομένα συστήματα γεωκτησίας στην Αφρική, αλλά και αυτό πρέπει να το εξετάσουμε κυρίες και κύριοι. Όχι μόνο εξαρτάται από αυτό η επιβίωση των πληθυσμών, αλλά και η παραγωγικότητα και δυνατότητα επενδύσεων. Τα δικαιώματα γεωκτησίας πρέπει κανείς να τα βλέπει όμως επιτόπου στην πράξη. Για να στηριχθεί κανείς πρέπει να βεβαιώνεται ότι τα ζητήματα ακτιματολογίου έχουν επιληθεί. Δεν μπορεί το παραδεδομένο σύστημα που η Αφρική το γνωρίζει από γενιές να απομακρυνθεί ή να εξαλειφθεί. Τα συστήματα αυτά υπάρχουν, χρειάζεται βεβαίω και νέε λύσει, αλλά και δικοδόσμηση θεσμικών φορέων και οργάνων. Επένδυση σε αυτού του τομεί χρειάζεται. Δίνοντα περισσότερε δυνατότητε στι τοπικέ κοινότητε, Βοηθώντα του πληθυσμού να δεσμευτούν καλύτερα στην όλη προσπάθεια, θα έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα. Τέλο, υπάρχουν συνολικέ πρωτοβουλίε. Είπαμε για την ΦΑΟ, την Παγκόσμια Τράπεζα. Η έκκλησή μα είναι όταν μιλάμε για την Αφρική. Και εφόσον κάποιε περιφερειακέ πρωτοβουλίε όπω το πλαίσιο για την Αφρική αγνοούνται, σε αυτή την περίπτωση, μετά από έξι χρόνια διαπραγματεύσεων για συμβουλευτικά μέτρα με όλου του εταίρου, Ας σκεφτούμε εάν θα έχουμε συνολικά σφαιρικά μέτρα για την Αφρική και τότε να λαμβάνονται υπόψη και οι περιφερειακές πρωτοβουλίες που προπάρχουν, ώστε να μην ε, καταστρέφουμε τις ήδη ταπεινές προσπάθειες των κρατών μελών. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε όλους τους προκεκλημένους και τους γερμηνείς που τόσο παραπάνω δούλεψαν. Θα σας ξαναδώ στις 3 για την ακρόαση με τον Επίτροπό μας Σιόλος και τον κύριο Πίμπαλξ.